E, Καλημέρα σας. Ζητήθηκε από τις πανικές Αρχές ε, η άρση ασυλίας του Κάρλος Πουτσιτεμόν και του Αντώνιο Κομίν. προκειμένου να συνεχίσει η ποινική διεξεβάρωση των δύο αυτών βουλευτών, δυνάμει του κανονισμού υποβάλλεται στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων που είναι καθήλυνα αρμόδια το εν λόγω αίτημα. Και προχωρούμε στο πρώτο σημείο της μέσιας διάταξης προφορική ερώτηση με θέματα θεσμικά όργανα και οργανισμού τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση, πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία. Θέλω να σας ενημερώσω, αγαπητοί βουλευτέ. πως ε, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την μπλε κάρτα ή για τη διαδικασία Catch the Eye μπορείτε να υποβάλλετε το έτοιμά σας είτε ηλεκτρονικά είτε με τον παραδοσιακό τρόπο. Έχετε τις ε, οδηγίες στην ε, είσοδο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συντάκτρια της προφορικής ερώτησης, την κυρία Ιρένη Τινάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. 17 Σεπτέμβρη του 2019 ήταν. Και ο κ. Άνταμ Φάρκα ανακοίνωσε την παρέτησή του από τη θέση του σαν εκτελεστικό διευθυντή τη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Θα ισχύσει από την 31 Ιανουαρίου 2020. Για να ξεκινήσει από Φεβρουάριο, 1 Φεβρουαρίου 2020, πρόεδρος της ΑΦΜΕ, πασίγνωστης εταιρείας, ε, εταιρείας που σύμφωνα στη σελίδα είναι η φωνή ε, των χονδρεμπόρων, των, των, ε, των υπηρεσιών των χονδρεμπόρων και της Ένωσης. Ξέρετε, είναι υπεύθυνη η τράπεζα για να εποπτεύει το τραπεζικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να καθορίσει τεχνικές προδιαγραφές εφαρμόζοντας βασικούς χρηματοπιστωτικούς ε, κανονισμούς. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή είναι βασικός θεσμικός φορέας που ρυθμίζει και εποπτεύει τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Επίσης, βέβαια, συνεχώς είναι στόχος των ομάδων πιέσης. Η ΑΦΜΕ, όπω και άλλοι εμπλεκόμενοι φορεί, φαίνεται ότι έχουμε μόνιμη διάδραση με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Σύμφωνα με τον κανονισμό προσωπικού και του δοτολογικού κανόνε, το Εποπτικό Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ανέλαβε την απόφαση πιθανότατα να θέσει περιορισμού όσον αφορά τον εκτελεστικό διευθυντή όταν θα εκτελεί τα καθήκοντά στον Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και μετά την αποχώρηση από αυτόν τον φορέα. Όμω, οι περιορισμοί στον κύριο Φάρκα και στη μελλοντική απασχόληση δεν φαίνονται ότι είναι ρεαλιστικοί ούτε εφικτοί να εφαρμοστούν. Εκτό αν ο κύριο Φάρκα γίνει απλώ κάποιο άλλο υπεύθυνο τη ε, ΑΦΜΕ, δεν βλέπω κάποιο θέμα Τη ΑΦΜΕ που να μην εμπίπτει στην, στον τομέα τη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και εμείς σχετίζεται με τα καθήκοντα του κ. Φάρκας. Εν γέννη, δεν είναι σαφέ για μένα Ποιο θα παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή των ελόγω περιορισμών, πιο συγκεκριμένα εκείνων που προβλέπει ότι δεν μπορεί να δίνει συμβουλέ ή να έχει σε επαφή με τα λόμπι, επαγγελματικέ επαφέ με το προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για 24 ε, μήνε μετά την αποχώρησή του από αυτή την αρχή. Πώ θα το εφαρμόσουμε και θα το ελέγξουμε ότι εφαρμόζεται αυτό. Ποιο θα το κάνει αυτό. Λοιπόν, για αυτού του λόγου ζητούμε να γίνει αναθεώρηση τη απόφαση των εποπτικών, ε, της Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής Δυστυχώ δεν είναι η πρώτη περίπτωση του κυρίου Φάρκα, ούτε η τελευταία πιστεύουμε, για το θέμα ασχόληση στον ιδιωτικό τομέα μετά καθήκοντα στο δημόσιο φορέα που θέτει θέματα σύγκρουση συμφερόντων. Αλλά θα πρέπει απαραίτητα να δράσουμε ούτω ώστε αυτή είναι η τελευταία περίπτωση. Ελπίζω πραγματικά ότι αυτή θα είναι η τελευταία περίπτωση αυτές οι κυλιόμενες θύρες όπου κάποιος από το θεσμικό φορέα, από τα θεσμικά όργανα πάει στον ιδιωτικό τομέα να θέσει, από ρυθμιστέ, ρυθμιζόμενους, από εποπτικούς φορείς, εποπτευόμενους φορείς, δυστυχώς υπονομεύουν και την ακεραιότητα του ατόμου αλλά και την αξιοπιστία όλων των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι των δημοσίων φορέων και εμπιστοσύνη που έχουν έναντι των θεσμικών οργάνων οι πολίτες είναι η ραχοκοκαλιά των δημοκρατιών. Γι' αυτό δεν θα ανεχθούμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά μας όργανα και οι υπηρεσίες μας να χάσουν την αξιοπιστία τους διότι εξυπηρετούν συμφέροντα ατόμων και πάντα πρέπει να επαγρυπνούμε ούτως ώστε να εξασφαλίζουμε και να εγγυόμεθα ότι δεν θα επηρεάζονται αυτοί από συμφέροντα. Γι' αυτό το λόγο καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την παρούσα πρακτική για την απασχόληση μετά από δημόσια θέση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ώστε να επεκτεθεί αυτή η αναθεώρηση σε σε συγκρού συμφερόντων πριν αναλάβουν δημόσια καθήκοντα και να θεσπιστεί νομικό πλαίσιο που θα πρέπει να προβλέπει επέκταση τη δυνατότητα να μπλοκαριστούν επαγγελματικέ μετακινήσει και θα πρέπει να υπάρχει περίοδο απόσβεση που θα είναι ανάλογη με τη συγκεκριμένη περίπτωση και θα συνοδεύεται από, προσωρινά μέτρα. Και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλει να αξιολογήσει κατά πόσο είναι ενδεδειγμένο ότι αυτοί οι φορεί τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι όσον αφορά την επιβολή των κανόνων περί προλήψεω συγκρούσεων συμφερόντων και πώ μια συνεπή εφαρμογή των κανόνων μπορεί να εξασφαλίζεται. Με τα χαρά είδα πραγματικά ότι το ψήφισμα υποστηρίχθηκε από την ομοφωνία των μελών της Επιτροπής Οίκων, καμία ψήφο κατά, καμία αποχή. Ελπίζω να είναι σαφές μήνυμα αυτό και ότι η Ολομέλεια θα ψηφίσει με μεγάλη πλειοψηφία το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο έχει ο Επίτροπος ε, κύριος Λενερτσίτς. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα αυτής της αρχής να υπογραμμίσω ότι συμμερίζομαι απολύτως το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε υψηλά ηθικά πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Υπηρεσία γενικότερα. Αυτά τα υψηλά πρότυπα είναι κρίσιμα, ε, κρίσιμα συστατικά για να μπορέσει η δημοκρατία μας ε, να ευδοκιμήσει. Αυτό απαιτεί ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, πρέπει να είναι αμερόληπτοι και να λογοδοτούν στους πολίτες το ότι ο κύριος Φάρκας πέρασε από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή στον ιδιωτικό τομέα δημιούργησε κάποιες ανησυχίες. Το αντιλαμβάνομαι. Και αναφέρεται, το αναφέρεται αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε σχέση με την πολιτική της και το ευρύτερο νομικό πλαίσιο. Υπάρχει και το θέμα ε, της οριζόντιας ούτως ή αυτού του νομικού πλαισίου. Ο ιστορικός κανονισμός, οι εφαρμοστικοί κανόνες που έχει που έχει ε, Green Commission, αφορά όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός αν υπάρχουν ειδικοί ε, κανόνες από κάποια υπηρεσία που όμως ε, ε επικυρώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κάθε υπηρεσία από εκεί πέρα έχει και την εξαρτησία της, μιας και πρόκειται για ξεχωριστές νομικές οντότητες. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες αυτές, οι οργανισμοί αυτοί είναι υπεύθυνοι ανεξάρτητα ε, για την ε, ε, εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τους κανόνες και την ε, ε λήψη επιμέρους αποφάσεων για το προσωπικό τους όπως με την, υπόθεση Φάρκας. Η απόφαση για τον κύριο Φάρκας ε, πάρθη από το Διοικητικό Συμβούλιο Εποπτών ε, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Τα μέλη αυτού του Συμβουλίου είναι οι επικεφαλής των εθνικών δημοσίων αρχών που είναι υπεύθυνε για την ε, εποπτεία των πνευματοπιστωτικών οργάνων σε κάθε κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει σε αυτές τις συναντήσεις με έναν μόνο εκπρόσωπο, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αυτό ήταν η επιλογή του νομοθέτη. Όπως αναφέραμε, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, όπως όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δεσμεύεται από τον εσωτερικό κανονισμό. Και εκεί υπάρχει ένα σαφέστατο πλήρες ε, ηθικό πλαίσιο. Η τελευταία δημοκρατία του 2013 ενισχύει αυτό το πλαίσιο σε ό,τι αφορά ε, τους περιορισμούς μετά το τέλος ε, μιας θητείας. Απαιτεί ο ιστορικός κανονισμός ότι η ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να αξιολογείται κατά την πρόσληψη ε, μετά από μια περίοδο ε, αναχώρησης για προσωπικού λόγου, μιας άδειας αναποδοχών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό είτε όταν κάποιος παίρνει άδεια ναυτοδοχών, είτε όταν έχει αποχωρήσει από ένα θεσμικό όργανο. Σε ό,τι αφορά την αποχώρηση, η αξιολόγηση γίνεται αναπερίπτωση. Οι απαγορεύσει ή οι περιορισμοί πρέπει να είναι αναλογικοί και στοιχειοθετημένοι. Για την κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ τη ανάγκη να εξασφαλίσουμε την ακαιρεότητα της εργασίας του θεσμικού ε, ε, οργάνου μέσω προσωρινών περιορισμών και απαγορεύσεων και βεβαίως να σεβαστούμε και το δικαίωμα του ανθρώπου αυτού να μπορέσει να επιλέξει την επαγγελματική σταδιοδρομία ε, κατόπιν ε, της θητείας τους, όπως άλλωστε προβλέπεται στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προβλέπει εφαρμοστικούς κανόνες που ε, επικυροποιούνται τακτικά, ιδιαίτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δημοσιολαβητή και στα πλαίσια ε, του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπάρχει μια νέα απόφαση για τις εξωτερικές ε, δραστηριότητες ε, και επαγγελματικέ δραστηριότητες μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία. Το 2018 επάρθη σχετική απόφαση. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στην σημασία της διαφάνειας. Από το 2014 ο ιστορικός κανονισμός προβλέπει ότι πρέπει ετησίως να αναφέρονται οι πληροφορίες για τις απαγορεύσεις περιορισμούς ε, για ένα χρόνο ε, να μην μπορούν ε, οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι να εργαστούν σε λόμπι ή σε ομάδες πιέσεων όταν αυτά αφορούν τομέα στον οποίο ήταν υπεύθυνο ως κατά τη του για τρία έτη. Αυτό βοηθάει για περαιτέρω διαφάνεια ε, υπάρχει και δημοσίευση των συνεδριάσεων των, με τους επιτρόπους, με τους εξωματούχους. Ε, τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει συνεργαστεί στενά με τον Ευρωπαϊκό Δημοσιολαβητή στα πλαίσια ερευνών όπου εξετάζεται το θέμα αυτό των revolving doors Τελειώνοντα τον περασμένο Φλεβάρι τη δεύτερη ε, έρευνά τη, ο ερευνατού Ευρωπαίο Δημοσιολαβητή επιβεβαιώνει την υψηλέ προδιαγραφέ ό,τι αφορά την εξαρτησία και τη διαφάνεια και ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να δίνει το καλό παράδειγμα. Τον Ιούλιο πέρυσι, ε, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε μια έκθεσή του αναφέρεται στο ηθικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ελληνικό Συνέδριο και ο έλεγχο του επιβεβαιώνει ότι σε μεγάλο βαθμό ε, οι, τα θεσμικά όργανα αυτά έχουν θεσπίσει ηθικά πλαίσια κατάλληλα και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εξαιρετικά προχωρημένη. Το νέο κολέγιο των Επιτρόπων ε, θα έχει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις σε ζητήματα ηθικής και αυτό θα το κάνει με αποφασιστικότητα. Η αντιπρόεδρο, η κυρία Γιούροβα έχει αναλάβει κατόπιν εντολής τη Προέδρου να συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής ηθικής που θα περιλαμβάνει όλα τα θεσμικά όργανα. Η συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωση στη διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για να μπορέσει να στεφθεί από επιτυχία το όλο εγχείρημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φέρμπερ, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με μεταπίδηση ενός ψηλόβαθμου δημόσιου εξωματούχου στον ιδιωτικό τομέα, ε, αν υπάρξει, είναι κάτι το οποίο διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ένωση και στα θεσμικά της όργανα. Υπόθηκε επίσης ε, ότι δεν υπάρχει ταυτόχρονα και απαγόρευση σε κάποιον να αλλάξει η θέση. Αν δηλαδή ψηλόβαθμο ε, αξιωματούχος θέλει μετά από ένα, μια περίοδο μεταβατική να μεταπηδεί σε μια άλλη θέση, μπαίνουμε σε κάποια έτσι λίγο δύσκολα ε, χωράφια για το πώς θα το ρυθμίσουμε. Λέει η Κομισιόν ότι οι εκτελεστικοί οργανισμοί έχουν του δικού του κανόνε. Αυτό είναι η μία δυνατότητα. Η δεύτερη δυνατότητα είναι να σκεφτούμε ένα πλαίσιο ε, κανόνων. Ε, και φαίνεται ότι ε, δεν θα έχουμε τη στήριξη του Συμβουλίου ίσως σε αυτή την πρόταση και καλό θα ήταν να ήταν παρόν σήμερα το Συμβούλιο για να εκφράσει την απόψή του. Επίσης, οι ίδιες οι εποπτικές αρχές φαίνεται ότι δεν θα έπρεπε να έχουν τόσο ε, μεγάλη ελευθερία κινήσεων για να αποφασίζουν τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια άλλα κριτήρια, όπω αυτό ισχύει για ε, του. Ε, θα έπρεπε να ισχύει του Ευρωπαίου κορυφαίου αξιωματούχου. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, αγαπητοί συνάλφοι πρέπει να κρατάμε καθαρό τον οίκο μα, συνηθίζω να λέω, και έχουμε στο ψήφισμα πει ότι και για το Κοινοβούλιο, όχι μόνο για τους οργανισμούς. Ένα συνεργάτης των Πρασίνων ε, που είχε ε, εργαστεί για κάποιους ε, φορείς θα πάει σε ένα βρετανικό οργανισμό για τα μιλτήρια και αυτό δεν γίνεται αφού έχει μεσολαβήσει η λεγόμενη cooling period. Εμείς λοιπόν το λέμε ξεκάθαρα και στο ψήφισμά μας ότι Καλό είναι ε, να μην υπάρχει και στην περίπτωση αυτή εξαίρεση, δηλαδή να ισχύουν ε, τα περισσότερα συμφέροντα για όλους τους υπαλλήλους όλων των οργάνων. Ευχαριστώ πολύ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ε, το λόγο έχει ο Πολ Τάγκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα αισθάνεται κανεί καλά να είναι μέλο του αυτού κοινοβουλίου, που είναι θεματοφύλακ, όταν θεματοφύλακα των συνθήκων εθελοτυφλού επίτροπε. Αυτό ο θεσμό ανέλαβε την πρόκληση να υπερασπιστεί του κανόνε που εστερνιζόμεθα έχει μέτρα διαφύλαξη κατά των αλλαγών θέσεων και κίνητρα που απορρέουν από αυτό. Αυτοί οι κανόνες μας βοηθούν να εμποδίσουμε τους εργαζόμενους να αναλάβουν θέσει που είναι ει βάρο των συλλογικών μας συμφερόντων. Παρ' όλα αυτά, χωρί την εφαρμογή αυτών, την πραγματική, οι κανόνες τελικά γίνονται τελικά χάρτινη Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και στο κοινό ότι δεν θα αφήσουμε αυτού του κανόνε τελικά να μην είναι χρήσιμοι και να γίνουν άσχετοι. Με το ψήφισμα στέλνουμε μια υπενθύμηση σαφέστατη και ηχηρή και ζητούμε ο κύριο Φάρκα να μην μπορέσει να μετακινηθεί τελικά και αν τελικά δεν γίνει αυτό να τον απαγορεύσουμε, να το απαγορεύσουμε από το να έχει θέση στο κοινοβούλιο. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια ερωτική σχέση, θα λέγαμε, σχέση αγάπη που αναπτύσσεται μεταξύ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και Τσάφημα από την άλλη, Τώρα από Γκάρι Σκότ και εκείνο διορίστηκε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα σύγκρουση συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε δύο εβδομάδε θα πρέπει να ξεκινήσουμε αν ο κ. Φάρκα πραγματικά να λάβει τα νέα του καθήκοντα. Πιστεύω ότι η ηγεσία του Κοινοβουλίου θα εφαρμόσει το έτοιμά μα να μην πάρει ε, ο κύριο Φάρκα, να μπορεί να μπαίνει στα κτίρια. Κύριε Επίτροπο, παρακολουθούμε και εσά και άλλου συναδέλφου σα για να επαληθεύσουμε κατά πόσο ε, τελικά δεν θα συναντήσουμε τον κύριο Φάρκα εδώ τα, τα επόμενα δύο χρόνια. Είμαι περήφανο διότι είχαμε στεναρή θέση μαζί. Πρέπει να τονίσουμε όμω κάτι. Κανεί δεν φαίνεται, δεν έχει καλή εικόνα όταν βγαίνει από αυτά τα θέματα. Είναι καλύτερα να επεσοζόμαστε του κοινού μα κανόνε και να μην αμφισβητείτε καθόλου ισχύ αυτών των κοινών κανόνε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα Λουίς Γκαρικάνου, για τρία λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μάθαμε στη διάρκεια τη χρηματοοικονομική ε, κρίση ότι αν υπάρχει μεγάλη εγκύτητα μεταξύ ρυθμιστών ε, και ρυθμιζών, τραπεζών κτλ., είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει σημαντικέ επιπτώσει. Ε, και δεν μιλάμε για σαφήθηκα πρότυπα και κανόνε, αλλά για ουσιαστικού κανόνες που έχουν να κάνουν ε, με τα φορολογικά και επηρεάζουν και τους φορολογουμένους, γιατί αυτοί που κάνουν τους κανόνες δεν τους θέτουν, δεν τους ε, συντάσσουν ε, για ε, τους πολίτες ε, και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο οποίο θέλουν να στρέψουν κάποια στιγμή από ό,τι φαίνεται και δεν βοηθούν και τελικά ε, κορώνα γράμματα χάνει ο φορολογούμενος, κερδίζουν αυτοί. Και γι' αυτό είναι σημαντικό το θέμα και είναι σημαντικό ε, να προχωρήσουμε ως κοινοβούλιο. Συγχαίρω τον κύριο Τάγκ, την κυρία Τινάλη, τον κύριο Φέρμπερ, τον κύριο Γκίγκολτ από την Επιτροπή ε, Οικονομικών. Όλοι οι συνάδελφοι ομόφωνα συμφώνησαν και συνεχίζουμε για τη διατήρηση ε, ορίων ε, διαχωριστικών γραμμών μεταξύ ρυθμιστών και ρυθμιζομένων. Πέραν για τέτοιων ορίων είναι αυτό το ε, οποίο συμβαίνει και ουσιαστικά γελιοποιεί και τους κανόνες που, τους οποίους αναφέρατε, γιατί τους παρακάμπτουν ε, τα θεσμικά αυτά οργανισμοί, εκτελεστικοί αυτοί οργανισμοί. Εμείς δεν το παίρνουμε ελαφρά το πρόβλημα. Ε, θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση ώστε να υπάρχει ε, πλήρης εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού. Η πρότασή σας φαίνεται καλή επίτροπε. Τέλος πάντων, οτιδήποτε μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή την περίπτωση, αυτή, σε αυτά τα όρια μεταξύ των δύο πλευρών του τείχου, ε, θα είναι κάτι θετικό για τις οικονομίες και τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λέει πρόεδρος εκ των Πρασίνων, ο Σβέν Γκίγκολτ για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, η υπόθεση του Άνταμ Φάρκας σωστά και δικαιολογημένα ε, προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, διότι πρόκειται για προφανή σύγκρουση συμφερόντων υπαριθμών το 2 ε, ε, της ΕΑΤ πηγαίνει στην κορυφή μιας μεγάλης τράπεζας λόμπι της ΑΦΜΕ. Και πραγματικά αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ευρωπαϊκή δημοκρατία και στο πώς λειτουργούν οι θεσμοί. Ε, πιστεύω ότι όσο πιο ψηλά βρισκόμαστε, τόσο πιο πολύ πρέπει να υπάρχει ε, προστασία από τις ε, συγκρούσεις συμφερόντων. Σίγουρα υπάρχουν οι κανόνες, αλλά έχουμε αυτή τις, αυτές τις περιστρεφόμενες θύρες, αυτή τη δυνατότητα μεταπίδησης από το δημόσιο στον δυτικό δομή και εκεί οι κανόνες δεν είναι τόσο ισχυροί. Χρειάζονται πιο ισχυροί κανόνες. Κανόνες που ισχύουν μέχρι τώρα είναι κακό αστείο. Και το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση Φάρκας και τα επιχειρήματα τα οποία κατατέθηκαν. Πράγματι, ε, η Κομισιόν ευχαρμόζει αυστηρά τον κανονισμό και γνωρίζουμε ότι και για την περίπτωση Φάρκας δεν έγινε ε, τελικά ε, πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση γιατί συχνά δεν βλέπετε πολύ, με πολύ μεγάλη αυστηρότητα το τι συμβαίνει στις δικές σας ε, τις υπηρεσίες και το ίδιο ισχύει και για το Κοινοβούλιο. Ε, δεν είναι θέμα τώρα των βουλευτών τι θα κάνει ένας συνεργάτης. Ε, σίγουρα πρέπει να υπάρχουν ε, προϋποθέσεις ε, που θα συνδέονται με την ε, μεταπίδηση αυτών των συνεργατών από το δημόσιο ιδιωτικό Δόμα. Συμφωνώ λοιπόν να λάβουμε αυτή την πρωτοβουλία και το λέμε και στη δική μας την έκθεση. Θέλουμε ακαιρεότητα, θέλουμε διαφάνεια και λογοδοσία και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, και οι προτάσεις ήταν να περιοριστεί ε, αυτή η ε, δυνατότητα περιστρεφόμενου θεωρώ γιατί μέχρι τώρα δεν οριζόταν αρκετά περιοριστικά και μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν θέλουμε να λάβουμε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα θα πρέπει η απόφαση που έχει ληφθεί να αναθεωρηθεί και αν όχι να υπάρξουν συνέπειες και αν έρχεται ε, από το μεγάλο τραπεζικό λόμπι και ο νέος 2, ε, αυτό θα είναι επίσης ε, πάρα πολύ αρνητικό και θα πρέπει να πούμε όχι, διότι όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να τακτοποιήσουν τα του οίκου τους για να λάβουν υπόψη αυτά που λέει το ψήφισμα, να έχει πραγματικά επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εν ονόματι της Δημοκρατίας και ταυτότητας Αγιοκίμ Κούρς για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολλά ήδη υπόθηκαν και δεν θα ήθελα να επαναλάβω. Ε, τα πραγματικά περιστατικά τα γνωρίζουμε, η ανάλυση είναι προφανής και κάτι πρέπει να αλλάξει εδώ. Κατά την άποψή μου όμως, δεν μπορεί να επιτρέπεται οι θυγόμενες αρχές να είναι αυτές οι οποίες ορίζουν και τους κανόνες ε, και με βάση αυτούς τους κανόνες να επιλύονται και διάφορες ε, υποθέσεις ε, που μπορεί να προκύψουν. Νομίζω ότι θα πρέπει τα τρία θεσμικά όργανα, Κομισιόν, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού να αποτρέψουμε την επανεμφάνιση τέτοιων προβλημάτων. Ε, αν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες ε, υπάρχει και κόστος ε, και πραγματικά πολύ προσπάθεια πρέπει να γίνει. Αλλά το θέμα είναι ότι αν οι ίδιοι οι θυγόμενοι δεν το καταλαβαίνουν και δεν νιώθουν τι κακή φήμη και τι εντύπωση δίνεται, τότε κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. δεν μπορούμε εμείς να επιτρέπουμε ε, να γίνονται αυτά τα πράγματα είτε στο κοινοβούλιο είτε στα άλλα θεσμικά όργανα. Θέλω να υπάρχει και προσωπική ευαισθησία και ευθύνη, πευθυνότητα, ώστε να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εν ονόματι Ενωτικής Αριστεράς της ΓΚΟΕ, Σερ Γκουσμάου για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς ε, υποστηρίζουμε αυτό το ψήφισμα που θα ψηφιστεί σήμερα το πρωί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όπως συνήθως ε, δεν έδειξε μεγάλη ζέση για το θέμα αυτό. Μετά την κρίση του 2009 είχε αναφερθεί ότι πρέπει η επιρροή του χρηματοοικονομικού κλάδου ε, προς θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετριαστεί. Ε, αυτό το είχε πει ο κ. Ντουράο Μπαρόσο, ο οποίος μετά όμως όταν τελείωσε τη θητεία του πήγε στην Goldman Sachs. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο αφορά πολλά θεσμικά όργανα της Ένωσης και είναι ακόμα πιο σοβαρό κάθε φορά που συζητούμε για το χρηματοοικονομικό ε, σύστημα και τις ρυθμιστικές αρχές τους. Ε, είτε αλλού, είτε εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι αποφάσεις που παίρνονται από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, ε, στην περίπτωση του Άνταμ Φάρκας, είναι πραγματικά σαν ένα κακόγουστο αστείο. Αυτός ο περιορισμός ουσιαστικά δεν αποτρέψει καμιά περίπτωση να δώσει στους νέους συναδέλφους ο κ. Φάρκας ε, τον ε, τηλεφωνικό κατάλογο με όλους τους συναδέλφους του. Ε, όπως, και όπως και περιορισμός να μην χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που έχει συσσωρεύσει εδώ και 8 χρόνια ε, στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Μια θέση όπου υπάρχει άμεση σχέση με τα λόμπι και τις πιέσεις τους. Θα λαμβάνει λοιπόν ε, ε, μια αμοιβή ο κύριος Φάρκας να μπορεί να χρησιμοποιήσει ακριβώς τις πληροφορίες αυτές. Αυτό είναι το τίμημα. Γι' αυτό πληρώνεται. Μιλάμε για την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής εδώ, έτσι. Οι δημοκρατικοί θεσμοί που έχουν εκλέξει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Και ρυθμιστικές αρχές τόσο σημαντικές όσο η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ουσιαστικά είναι όμοιροι είναι σε ομοιρία αυτών των λόμπι, αυτών, αυτού του τομέα του χρηματοοικονομικού. Και πρόκειται για μια απόφαση που παίρνει ένας, Ευρω... ένας διευθυντής Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής που προέρχεται ήδη από λόμπι, από, το... από, τράπεζα ε, του ε, Σανταντέρ. Αυτό λοιπόν το Σιρίαλ βλέπετε έχει πλέον πολλά κεφάλαια και βεβαίω ε, δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για το, ε, τα εργασιακά δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Είναι αστείο. Δεν μπορεί να εργάζεται σε μια ομάδα πίεση. Τι σημαίνει ε, εργατικό δίκαιο. Αν ένα εργαζόμενο αν ένα εργαζόμενο είχε τόση προστασία όσο έχουν αυτοί οι άνθρωποι, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κ. Φερνάντε για δύο λεπτά. Ναι, Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμο κύριε ε, Επίτροπε, η τελευταία χρηματοοικονομική κρίση έδειξε ότι υπάρχουν πολλές φεζόνες όπου οι ρυθμιστικές αρχές, οι εποπτικές αρχές μοιράζονται πληροφορίες, μοιράζονται ανταλλαγές απόψεων με έναν τρόπο όπου τελικά επηρεάζονται οι αποφάσεις. Και αυτή η αντίληψη, η πρόσληψη από τον Ευρωπαίο πολίτη έχει φτάσει να είναι ότι οι δημόσιες αρχές δεν είναι όσων εξάρτητες θα έπρεπε να είναι απέναντι σε κάποιες ομάδες συμφερόντων. Και αυτή η πρόσληψη υπονομεύει την ε, εμπιστοσύνη στο δημοκρατικό μας σύστημα, υπονομεύει την εμπιστοσύνη, την πίστη στο ευρωπαϊκό όραμα τελικά, στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Η Επιτροπή Οικονομικών του Κοινοβουλίου ομόφωνα, ομόφωνα έτσι, όχι με ευρία πλειοψηφία, ε, έχει εγκρίνει μια σειρά από προαπαιτούμενα για να αποφύγουμε αυτά τα φαινόμενα των evolving doors ε, διότι δεν μπορούμε να δεχτούμε οι συνάδελφοι από τι εποπτικέ αρχές να είναι αυτοί που θα αξιολογούν κατά πόσο οι αξιωματούχοι αυτών των ε, οργανισμών θα μπορούν να εργάζονται σε δάδε στη δίνα επιχείρηση. Πρέπει να, είναι, να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή που θα αφορά όλα τα θεσμικά οργάνα της Ένωσης, που θα αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που με κάποιο τρόπο θα αξιολογεί σαφώς, με βάση σαφή κριτήρια, τα χαρακτηριστικά αυτών των μετακινήσεων των επαγγελματικών για να μπορέσει και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η εμπιστοσύνη προς την ευρωπαϊκή δημοκρατία και να ανοίξουμε ε, επιτέλους ε, ένα ε, πεδίο μεγαλύτερης πολιτικής ε, νομιμοποίησης και ευθύνης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νταμιάν Καρέμ έχει το λόγο για δυόμιση λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, όλοι το λέει, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Θα πρέπει να τελειώσουμε με την ε, δυσανάλογη και αδιαφανή επιρροή των λόμπι στη δημόσια ζωή μα για τα οικονομικά, πυρηνικά, ορυκτά, καύσιμα κλπ. Υπάρχουν πολλά λόμπι και οργανωμένα για να προωθούν τα ιδιωτικά συμφέροντα με συνέπειε που γνωρίζουμε για τους απορρίθμιση των τραπεζών και διάφορα άλλα. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια να πολεμήσουμε αυτέ τι σκοτεινέ δυνάμει, διότι πόρα που έχουμε από τον έχουμε ε, ξεμπερδέψει με τη διαφθορά, όπω και στη Γαλλία. Όπω ε, βλέπετε, την τελευταία έκθεση του Συμβουλίου τη Ευρώπη, 9η Ιανουαρίου του 2020, που λέει ότι υπάρχουν ζώνε γκρίζε στην καταπολέμηση τη διαφθορά και ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τι επαφέ του εκτελεστικού κλάδου και ομάδων συμφερόντων του, ώστε η επιρροή του αφορά τι αποφάσει να Για να ξαναβρούμε όλη την εμπιστοσύνη των πολιτών θα πρέπει λοιπόν να τεθεί τέρμα στην συνεργασία μεταξύ δημοσίου συμφέροντος και ιδιωτικού. Παραδείγματο χάρη, διότι αυτό μα ενδιαφέρει σήμερα, είναι ένα ανώτατο υπάλληλο, ο κ. Φαρκά, που ήταν υπεύθυνο για την εποπτική εποπτεία των τραπεζών, να μην μπορεί να γίνει από τη μια ώρα την άλλη διευθυντή του βασικού λόμπι για τα χρηματοπιστωτικά. Όμω αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και δεν είναι αποδεκτό. Χρειάζονται κανόνε αυστηρότεροι για να φυλαχθεί η ακαιρεότητα των θεσμικών μα οργάνων. Χρειαζόμαστε, παραδείγματο χάρη, να καθορίσουμε περιόδου μακρύτερε μεταβατικών μεταξύ δύο δραστηριοτήτων για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων με απαγόρευση να έχουν κάρτα εισόδου στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει πραγματική ανεξάρτητη υποπτία, ούτω ώστε όταν παρουσιάσετε αυτέ υποθέσει να γίνεται αυτό, χάρη δημιουργία αυτή τη ανεξάρτητη αρχή για τα δοντολογικά ε, που είχατε μπλοκάρει που θέλαμε να υποσχεστούμε τα δημόσια συμφέροντα. Θα πρέπει να συνεπείς γι' αυτό, ξεκινώντας αποδεχόμε τη διαφάνεια και τη σαφήνεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Άντζελο Τσόκα. Για ένα λεπτό έχει το λόγο δεν σκεφτόμαστε σήμερα να γίνει, να γίνει παρθένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά οργάνα χτυπώντας τον κόδωνα των συναγερμών για τις δεκαετίες που βλέπουμε ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η επιρροή των λόμπι, οι περιστρεφόμενες πόρτες, εναλλαγή καθηκόντων και η έλλειψη διοντολογίας επί σειρά ετών. Το κατηγορούμε αυτό, το καταγγέλουμε αυτό και οι πολίτες αυτά τα θεσμικά όργανα ε, εκόφευαν επί σειρά ετών. Διότι εντός αυτών θεσμικών οργάνων, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση υπάρχει μεγάλη επιρροή από τις ομάδες πίεσης. Τώρα είναι σημαντικό να πάμε να δούμε τι συνέβη, δηλαδή πού η Νομισματική Ένωση δημιούργησε ζημιά Υπάρχουν καταστήματα που έκλεισαν, επιχείρησει που έκλεισαν και πολίτε που έχασαν τη δουλειά του λόγω τη επιρροή αυτών των λόμπι. Λοιπόν, δεν περιοριζόμαστε, πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στη ρύθμιση του μέλλοντο, αλλά να βρούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτέ τι ε, δράσει, για αυτά τα σφάλματα και τις προσχεδιασμένες εγκληματικές ενέργειες που έλαβαν χώρα αυτά τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ο, ο κύριος Άλβετ Σάντ για ένα λεπτό έχει το λόγο η ρύθμιση της Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα θεσπίζεται μέσω σφαλμάτων καμιά φορά. Οι, τα υψηλά στελέχη έχουν σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν για να εφαρμόζουν ρυθμιστικά κείμενα και βάσει αυτών ε, νέε διοικητικέ δομέ και πρακτικέ ενδεχομένω θα πρέπει να αναπτυχθούν, διότι η Τραπεζική Ένωση και με ενιαία κεφαλογορά τα απαιτούν. Περίπλοκα συμφέροντα παίζουν ρόλο, εθνικά και υπερεθνικά συμφέροντα, κρατικά και ιδιωτικά συμφέροντα υπάρχουν περίπλοκες πιέσεις και εκεί που διαχειρίζονται τις μυθικές κινήσεις ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι και αμερόληπτοι. Θα πρέπει οι ρυθμιστικοί φορείς να έχουν τη διαβεβαίωση ότι αυτό ισχύει. Αυτή η διαβεβαίωση δεν είναι διαθέσιμη τώρα. Οι υπολογισμοί για τη νέα εργασία και οι προσδοκίες μπορούν να παρασύρουν κάποιους που θεσπίζουν κανόνες και ε, οι πληροφορίες που διαθέτουν αυτοί που αλλάζουν θέση από ρυθμιστές που αλλάζουν θέση ίσως να δώσουν ε, πλεονεκτήματα στο νέο εργοδότη. Δεν πρέπει να ανεχθούμε τις περιστρεφόμενες πόρτες. Υπάρχει και θέμα αντίθετο. Πρέπει να καταλάβουμε πως οι συγκρούσεις των συμφερόντων θα μπορούσαν να προκύψουν από θέσεις που κατήχαν κάποιοι πριν αναλάβουν δημόσια καθήκοντα. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δεν θα πρέπει να ανεχθούμε την μόλυνση τη ρυθμιστική ουδετερότητα που απαιτεί η Ευρωζώνη, αν θέλουμε να αναπτυχθούμε κανονικά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριο ε, ε, Μίκουλα Πέξα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι εδώ σήμερα για να καταγγείλω το πρόβλημα των περιστρεφόμενων πορτών μεταξύ ε, των Ευρωπαϊκών Συμφωνών Οργάνων και των ιδιωτικών ομάδων συμφερών. Πολύ συχνά Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φεύγουν από τις πιο βαθμές θέσεις τους και χρησιμοποιούν τα, τα, τις επαφές τους στον ιδιωτικό τομέα, τις εκμεταλλεύονται. Έχουν την υποχρέωση αυτοί οι ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ε, όταν αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα ε, να τα αναφέρουν. Αυτό όμως συχνά το αγνοούν. Πραγματικά είναι συστημικό πλέον το πρόβλημα και μπορεί να υπονομεύσει την ακεραιότητά μας, ε, τη, τη φήμη μας. Πρέπει να είμαστε ένα παράδειγμα διαφανών προτύπων, ηθικών προτύπων. Ζητούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει περισσότερα ε, για να μπορέσουμε να προλάβουμε αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο να δει ποιε μπορεί να είναι οι βέλτιστε πρακτικέ στον τομέα αυτό. Τον περασμένο Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε να επανεξετάσει ε, του σχετικού κανονισμού. για να βρωθούν και κάποιες λύσεις. Ε, δεν θέλω μόνο να επικρίνω, έτσι. Ζητούμε λοιπόν ένα αρμονισμένο νομικό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται, θα εφαρμόζεται τα ίδια ηθικά πρότυπα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Δεύτερον, η δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής ηθικής που θα εξετάζει όλες τις προβληματικές υποθέσεις. Τρίτον, υποχρεωτική περίοδος 12 μηνών όταν ολοκληρώνει τα καθήκοντά των σεξουαλικών αξιωματούχος για να εργαστεί σε οποιοδήποτε λόμπι. Να υπάρχει τερά, ε, απόλυτη διαφάνεια και οι δηλώσεις συμφερόντων και οι συγκρούσεις συμφερόντων να δημοσιεύονται επιγραμμικά και να είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ και τώρα τον λόγο έχει ο κύριος Μαξιμίλιαν Κρά. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Αξιότιμε Επίτροπε, ε, κύρια Πρόεδρε, έχουμε εδώ ένα αδιέξοδο. Ε, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ε, έχουν ε, μεταπηδήσει από τον δημόσιο ιδιωτικό τομέα ε, και αυτό μπορεί να εξοργίζει. Αλλά από την άλλη πλευρά, ε, τι θα κάνουν αυτοί οι δημόσιοι ε, αξιωματούχοι αν πρέπει να έχουν αυτή την περίοδο αναμονής, την περίοδο μετάβασης. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως θέλουμε να δουλεύουν για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ε, θα υπάρξει στη συνέχεια ε, είναι προπρογραμματισμένο αν θέλετε των με το αυτοί οι άνθρωποι ε, θα φύγουν μετά και αν τους δημιουργούμε προβλήματα δεν πρόκειται να έρθουν στο δημόσιο τομέα ποτέ και το είπε και ο συνάδελφος Κούς προηγουμένως ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία προσωπική και λογοδοσία ώστε να μπορεί κάποιος να ξέρει ότι θα επονιδιστεί στη στην ε, δημόσια κοινή γνώμη. Ε, και ε, δεν νομίζω ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα με κανόνες από τις εθνιστικές αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκραπίνη. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για σύγκρουση συμφερόντων και πώς μπορεί αυτή να προληφθεί. 24 Οκτωβρίου πέρυσι το ξανασυζητήσαμε για τελευταία φορά και τότε μας έλεγε ο Επίτροπος ότι ναι, μεν ε, πρέπει να δούμε το νομικό πλαίσιο, να το εναρμονίσουμε, να παληθεύσουμε, να δούμε πώς μπορούν να είναι ομοιόμορφες οι ρυθμίσεις σε όλες τις χώρες. Δεν έκανε τίποτα έκτοτε ο Επίτροπος, είχε υποσχεθεί συγκεκριμένα μέτρα η ρύθμιση των ε, ευρωπαϊκών χρηματαγορών σίγουρα ε, είναι κάτι που θα επηρεάσει το σύνολο της αγοράς. Δεν καταλαβαίνω το Συμβούλιο και την Κομισιόν που παραμένουν αδιάφοροι απέναντι σε τέτοιου είδους συγκρούσει συμφερόντων. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί ένας επίτροπος να λέει ότι σε αυτή την περίοδο θα επαληθεύεται η συγκρούση συμφερόντων. Μα είναι αργά. Πρέπει να υπάρχει πρόληψη εκ των προτέρων ελέγχονται όλα αυτά. Για την περίπτωση Φάρκα πρέπει να αντιδράσουν κατεπηγόντω. Δεν πρέπει να πάρει τα νέα του καθήκοντα. Ευχαριστώ κύριο Μπάλτ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι προ συμφέρον των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων να μπορέσει να προλάβει ε, την απάτη, την παραβίαση ουσιαστικά των κανόνων από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Το γεγονός ότι ο κ. Φάρκας ε, είχε με, με τέτοια σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή ε, Τραπεζική Αρχή ε, και που περνάει και εργάζεται πλέον σε αυτή την οργάνωση η οποία επηρεάζει την αγορά είναι πραγματικά ανησυχητικό. Είναι προ συμφέρον, επαναλαμβάνω, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να εντοπίζει και να προλαμβάνει τέτοιου καταστάσει. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να παρακολουθήσει τι εργασίε τη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, καθώ ε, και τη ένωση αυτή ε, ε, στην οποία θα εργάζεται ο κ. Φάρκα. Μήπω θα ξεχαστεί τελικά η επιρροή του κυρίου Φάρκας ή θα πρέπει παρακολουθούμε στενά την υπόθεση αυτή. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Τράιαν Μπασέσκου, για ένα λεπτό παρακαλώ. Λείπει, όχι, εδώ είναι ο κ. παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για την πιο σημαντική πηγή απάτης ε, το ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα. Η σύγκρουση συμφερόντων είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι συνεχώς επίκαιρο. Δυστυχώς είναι κάτι που ρυθμίζεται και που ερμηνεύεται διαφορετικά από χώρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έλλειψη αυστηρών κριτηρίων ε, στην νομοθεσία περί σύγκρουσης συμφερόντων είναι που κάνει και τη διαφορά από τη μία χώρα στην άλλη. Σε κάποιες χώρες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα αυτό. Σε κάποιες άλλες πάλι η νομοθεσία ε, είναι πιο χαλαρή. Η σύγκρουση συμφερόντων όμως ε, επηρεάζει τις εργασίες των διοικητικών αρχών, των δημοσίων υπηρεσιών σε κεντρικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση ρύθμισης του σύγκρουση συμφερόντων που να ισχύει για το σύνολο των κρατομελών της Ένωσης και για όλους τους κλάδους, διότι αυτή είναι η πηγή της διαφθοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπόγκταν Γιόνσα. Ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, λέει ο κύριος Ζόνσκα, συγγνώμη. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα στο οποίο αναφέρεται όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το νέο Green Deal. Θα διατεθούν σημαντικά κονδύλια στο project αυτό. Συμμετέχω στην νομοθετική διαδικασία και διαπιστώνω ότι οι ομάδες συμφερόντων ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτά τα project, αλλά και οι χρηματαγορές δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το στάδιο να γίνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ αυτών που εργάζονται γύρω από αυτή την νομοθετική διαδικασία και αυτών που στη συνέχεια θα γίνουν σύμβουλοι ή πρόεδροι ε, σε αυτές τις ε, ε, εταιρείε που θα υποφεληθούν από αυτά τα κονδύλια τα οποία θα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Φοβούμε ότι μπορεί να δημιουργήσουμε νέες χρηματοοικονομικές φούσκες και απάτες. Ε, και δίνω μεγάλη έμφαση στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Λέναρτσιτς, στο όνομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, άκουσα προσεκτικότατα τα σχόλιά σας. Είναι σημαντικό το θέμα, πολύ σημαντικό, σας διαβεβαιώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αδιαφορεί για τα θέματα αυτά ενδεχομένων συγκρούσεων συμφερόντων και δεύτερον σίγουρα δεν παρατηρούμε ελαφρά την καρδία αυτή την υπόθεση ούτε άλλη όσον αφορά ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα παίξει το ρόλο συμβούλου για απόφαση που θα λάβει ένας εξάρτητος φορέας που είναι το Εποπτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Θεωρούμε όμως ότι μπορούμε να ρίξουμε περισσότερο φως θα το προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό υπό το φως των σχολείων που ακούστηκαν. Καταρχάς, ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Εποπτικό Συμβούλιο, που επαναλαμβάνω δεν έχει δικαίωμα ψήφου, προσπάθησε να έχει τους αυστηρότερους δυνατούς περιορισμούς, διότι πραγματικά πόρισμα ήταν ότι αυτή η υπόθεση συνεπάγεται το σύγκρουση συμφέροντων. Το Εποπτικό Συμβούλιο εξέτασε προσεκτικότατα το ζήτημα και θεώρησε ότι η σύγκρουση των συμφερόντων μπορούσε να αντιμετωπιστεί με συμπληρωματικού περιορισμούς που ξεπερνούν τις ελάχιστες συνθήκες που εφαρμόζονται σαν νότερα στελέχη. Η διάρκεια της περίοδου απαγόρευσης επαφής με τα λόμπι είναι διπλάσια από τη διάρκεια που προβλέπεται στο ελάχιστο. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες των περιορισμών, αλλά το Συμβούλιο έπρεπε να σταθμίσει την κατάσταση να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των δημοσίων συμφερόντων από τη μία πλευρά και των δικαιωμάτων των ατομικών από την άλλη να επιτρεπεί σε αυτόν τον άνθρωπο ε, να συνεχίσει τη δουλειά του. Σημαντικό ερώτημα ετέθη μεταξύ άλλων. Ποιος θα παρακολουθεί και θα εξασφαλίζει την εφαρμογή αυτής της απόφασης. Ε, πρέπει να σημειώσουμε ότι η απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής αρχής συμπεριλαμβάνει διάταξη περί Οι περιορισμοί που θα επιβληθούν θα κοινοποιηθούν στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και θα πρέπει να λογοδοτούν στον Πρόεδρο για επαφές με τον κύριο Φάρκας από τη στιγμή που θα έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία της CBA. Η EBA υπόκειται στην υποχρέωση να ενημερώνει το δημόσιο κάθε έτος για την εφαρμογή της απαγόρευσης όσον αφορά την παροχή συμβουλών και την επαφή με τα λόμπι και τις υποθέσεις που εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν. Ο κύριος Φάρκας, όπως οποιοδήποτε, άλλ, οποιοδήποτε άλλος μέλος του προσωπικού που είναι ενεργό, υπόκειται στον κανονισμό του καταστατικού και στις διοικητικές ε, Διαδικασίε που ίσω να ακολουθηθούν σε περίπτωση παράβαση, ακόμα και όταν αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Όταν η υποπτική αρχή ή τη CBA ή όλα εντοπίσουν κάποια μη εφαρμογή των κανόνων μετά από έρευνα και ε, πειθαρχικέ διαδικασίες, ο κ. Φάρκας ίσως θα πρέπει να υποστεί διοικητικά μέτρα που καθορίζονται στον κανονισμό περιπροσωπικού. Ε, νομίζω λοιπόν ότι αυτό εξηγεί ότι δεν έχουμε αφήσει τα πάντα στην τύχη. Υπάρχουν διατάξεις που θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι αυτοί οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν ορθώς. Κλείνοντας, να επαναλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει ή προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι ύψιστες προδιαγραφές δεντολογικές εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες έχοντας ένα αρμονισμένο νομικό πλαίσιο. Όμως είναι ευθύνη Εν τη αυτή περιπτώση του Υποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής η εφαρμογή του νομικού πλαισίου λαμβάνοντας αποφάσεις ανεξάρτητα ε, για τους περιορισμούς μετά την ε, απασχόληση σε αυτό το φορέα βάσει του κανονισμού και του κανονισμού προσωπικού. Επίσης είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της EBA να εξασφαλίζει ότι θα πρέπει να παρακολουθείται η εφαρμογή των αποφάσεων. Τέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα επιδιώκει τη βελτίωση του υφισταμένου πλαισίου. Το εντολογικό πλαίσιο το παρόν συνεχώς αναθεωρείται. Θέλουμε να επιφέρουμε βελτιώσει συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων. Θέλουμε να έχουμε ανεξάρτητο εποπτικό φορέα και προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και άλλους θεσμούς στην όλη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κλείνεται περατούτε αυτή η συζήτηση. Έλαβα ένα σχέδιο ψηφίσματος που θα υποβληθεί σε ψηφοφορία σήμερα. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Πάμε στη συζήτηση για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ε, δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η πρώτη συζήτηση θα αφιερωθεί στο Μπουρούντι και ιδίω στην ελευθερία της έκφρασης. Να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να λάβετε το λόγο μέσω γαλάζιας κάρτας, παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά, βρίσκονται στην είσοδο της αίθουσας οι ηλεκτρονικές συσκευές για να ζητήσετε το λόγο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Έλλη Σόμς, η οποία έχει δύο λεπτά στη διάθεσή της. Έχετε το λόγο, κυρία μου. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Μπουρούντι είναι μια όμορφη χώρα. Αλλά έχει βιώσει πολλά δράματα και τραγωδίες. πάνω από 4.000 με 140.000 θύματα ανακαλύφθηκαν. Και σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας έκφρασης, ε, της ελευθεροτυπίας ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ακρογωνή λύθη της δημοκρατίας ε, και της βιώσιμης οικοδόμησης της ειρήνης. Συζητούμε αυτό το θέμα σήμερα λόγω της καταστολής, ε, του πρόσφατου παραδείγματος κυβερνητικής καταστολής, δημόσιος αγγελέας 30 Δεκεμβρίου ζήτησε 15 ετή κάθεξη για τέσσερις δημοσιογράφους και, τον, και την οδηγό τους. Ότι τον οδηγό συνελήφθησαν τον Οκτώβριο ενώ κάλυπταν τις ε, συγκρούσεις ε, διαδηλωτών ε, με τις κυβερνητικές δυνάμεις και θεωρεί, καταγορήθηκαν για υπονόμευση του, του κράτους. Δεν είναι η πρώτη δημοσιογράφη. Τον Ιούλιο του 2016 ο Ζαμ Τζιρουμάν, ένας άλλος δημοσιογράφος, ρεπόρτερ, εξαφανίστηκε και έκτοτε δεν υπάρχουν νέα του. Ένας άλλος δημοσιογράφο το 2015 μαζί με τη γυναίκα και τα παιδιά δολοφονήθηκαν στην Μπουζουμπούρα και πάλι δεν διαλευκάνθηκε αυτή η υπόθεση. Μάνου Ρουκούκη, ακτιβιστή για την ε, κατάργηση των ε, βασανιστήριων, καταδικάστηκε πέρυσι 30, σε 32 χρόνια κάθυρξης ε, μεταξύ άλλων. Καλούμε άμεσα και άνεφόρον να απελευθερωθούν οι δημοσιογράφοι που κρατούνται, όπως και οι περασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε εκλογέ το 20, σημαντική στιγμή για τη χώρα. Ο πρόεδρος είπε ότι δεν θα επιδιώξει πανεκλογή, αλλά αν θέλουμε να είναι αξιόπιστες αυτές οι εκλογές πρέπει να γίνουν αλλαγές, να αλλάξει κατάσταση ε, σε ό,τι αφορά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απευθύνω έντονες εκκλήσεις να κάνει ό,τι πρέπει το Μπουρούντι για μια βιώσιμη δημοκρατία. Και χαιρετίζω τον αγώνα των δημοσιογράφων και των υπερσπών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο στη δεύτερη συντάκτρια του ψηφίσματος, την κυρία Άννα Φωτίγκα, για ένα λεπτό. Το Μπουρούντι είναι μια από τι φτωχότερε χώρε στον κόσμο. Έχουμε ένα πολύ αναλυτικό σχέδιο ψηφίσματος που ακριβώς ε, απεικονίζει πολύ εύληπτα την κατάσταση όταν ε, πλησιάζουν προεδρικές γενικές εκλογές. Η κατάσταση και των ε, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εκπροσώπων του τύπου είναι δυνότατη. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορούν να διεξαχθούν ελεύθερες εκλογές αν δεν υπάρχει πληροφόρηση της κοινή γνώμης και μάλιστα με εύλογο τρόπο, με αξιόπιστο τρόπο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για το πολύ καλό ψήφισμα και ολοκληρώνω την παρέμβασή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Μαρία Αρενά για δύο λεπτά παρακαλώ. Η πολιτική κρίση στο Μπουρούντι έχει καταστροφικές συνέπειες στον πληθυσμό. Τα οικονομικά και θεμελιώδη δικαιώματά τους ε, αυτή τη στιγμή πλήττονται. Ε, δεν μπορούν εύκολα να ψηφίσουν. Άνθρωποι οι οποίοι είναι αντιφρονούντες με την ευρία έννοια έχουν ε, μπει στη φυλακή, έχουν εξοριστεί, έχουν ε, εκτελεστεί ορισμένε φορέ. Ε, είναι όλο και πιο περιορισμένη η ελευθερία του τύπου. 22 Οκτωβρίου του 2019, τέσσερι ε, δημοσιογράφοι της ομάδας Ιουάκου καθώς και ο οδηγός τους ε, συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν ε, για ε, θέσεις εκείνων της ασφάλειας της χώρας. Ένας άλλος δημοσιογράφος από την ομάδα Ιουάκου επίσης έχει, είναι, έχει εξαφανιστεί από το 2016 σε ό,τι αφορά αυτές τις ε, ε, και τις ε, συλλήψεις είναι σαφές ε, ότι έχει πληγεί το κράτος δικαίου. Δεν δεχόμαστε αυτές τις αυθαίρετες συλλήψεις. Ζητούμε την απελευθέρωση όλων των δημοσιογράφων της ομάδας Ιουάκου που απλά άσκησαν το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Για να σταματήσει η ένταση στην περιοχή ζητούμε από την Αφρικανική Ένωση να στείλει παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπουρουντή και ζητούμε από τα Ηνωμένα Έθνη να ξεκινήσουν ανεμερόληπτε έρευνε για όσου είναι ύποπτοι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητούμε από τα κράτη-μέλη τη Ένωση Επίση. να να βοηθήσουν οικονομικά την κοινωνία των πολιτών τη χώρα αυτή και οι κατευθείαν γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα να γίνουν σεβαστά να γίνουν σεβαστές παρακολουθώντας τις δίκες αυτών των ακτιβιστών και, επισκε... και οργανώνοντας επισκέψεις στη χώρα αυτή και στους ακτιβιστές αυτούς. Πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις απέναντι στον Μπορουντή ε, εστιασμένε κυρώσει που έχουν αποφασιστεί από το Συμβούλιο και δεν πρέπει να έρθουν σήμερα. Θα ήταν ένα λαθασμένο, καταστροφικό πολιτικό μήνυμα σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Μπουρούντι. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βουλευτή και τώρα η κυρία Βιλιανούεβα Ρουίθ για δυόμιση λεπτά έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ε, πρόκειται για μια γενικευμένη διαδικασία ε, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα από χώρα σε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω νομοθεσιών ε, που ε, ουσιαστικά οδηγούν σε ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας ενώ η ακροδεξιά αλωνίζει στην Λατινική Αμερική ισχύει το ίδιο στην Μέση Ανατολή με τη δημιουργία ενός μιας μαύρης τρύπας ατιμορρησίας όπου οι οργανώσει για, για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαγορευμένε και αυτό ισχύει και στο Μπουρούντι βέβαια. Η πολιτική οικονομική κρίση στο Μπουρούντι εδώ και τέσσερα χρόνια όλο και επιδεινώνεται. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολιτική υφή που έρχονται από την κυβέρνηση και η κατάργηση δημοσίων και ατομικών ελευθεριών αυξάνεται καθώ πλησιάζουν οι ε, προεδρικέ ε, και βουλευτικέ εκλογέ το 2020. Πρέπει να υπάρξει άμεση απελευθέρωση και χωρί όρου όλων των κρατουμένων που εκφράζουν απλά τι απόψει του. Πρέπει να σταματήσει ε, η βία, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι απειλέ κατά τη των πολιτών. Θα πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά για την ε, ελευθερία έκφραση, να σταματήσει ο περιορισμό των ΜΚΟ να γίνουν σεβαστέ οι διεθνεί συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατά των ε, βασανιστήριων. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το να σταματήσουν αυτοί είναι ε, εκ των νουκ άνευ για να μπορέσουν να ξεκινήσει μια διαδικασία πολιτικού διαλόγου, ειρηνικού διαλόγου. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει εάν εμεί στην Ευρώπη δεν ε, εμπλακούμε. Θα πρέπει να αποφασίσει η Ευρώπη τελικά τι ρόλο θέλει να παίξει στον κόσμο σήμερα. Χρειάζονται συγκεκριμένε δράσει. Η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει ότι δεσμεύεται για την ειρήνη ε, δίνοντας καθεστώς πρόσφυγα και για όσους ε, ζητούν άσυλο τον από τον Μπουρούντι, όπως άλλωστε ε, ζητούν τα Ηνωμένα Έθνη και να υπάρξει βοήθεια και για την ανάπτυξη στην περιοχή αυτή για να μπορέσουν και οι γειτονικέ χώρες να υποδεχθούν τους πρόσφυγες. Θα πρέπει οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εργάζονται στον Μπουρούντι να σέβονται τους διεθνούς, τις διεθνή αυτή πρότυπα. Ήταν πάντα δύσκολη η σχέση μας με την ε, Αφρικανική Ένωση. Δεν μπορούμε ε, να είμαστε περήφανοι για την δράση μας στην Αφρική. Ήρθε η στιγμή η Ευρώπη να ξεκινήσει μια σχέση με στόχους εξωτερικής πολιτικής που να ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα του πληθυσμού της υπήρου αυτής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Άρμπα Κοκαλάρη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόκειται, πρέπει να θυμίσουμε ότι η ελευθερία της έκφρασης και τα ανεξάρτητα μέσα είναι θεμελιώδης σημασία για τη δημοκρατία και μια ελεύθερη κοινωνία. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση επιδείνωσης της κατάστασης σε όλο τον κόσμο και βάσει του δίκτυου. World um, Freedom όσον αφορά την ελευθεροτυπία βλέπουμε επιδείνωση και εγώ ανησυχώ πολύ. Στο Μπουρούντι βλέπουμε ότι είναι μία από τις χώρες εκείνες στην οποία η κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης ε, καταστέλλονται. Υπάρχει μία σειρά ακτιβιστών και δημοσιογράφων που είναι ένα παράδειγμα που πλήττονται από αυτό και υπάρχει ε, μεγάλος κρατικός έλεγχος. Και τον Οκτώβριο τέσσερις δημοσιογράφοι και ο οδηγός τους ε, ε, συνελήφθησαν ενώ ασκούσαν τα καθήκοντά τους, κάναν τη δουλειά τους. Αυτό σημαίνει ότι τώρα θα πρέπει να δράσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις όσον αφορά τον Μπουρούντι. Θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε τον Μπουρούντι να σέβεται τις διεθνείς συμφωνίες και να απελευθερώσει αμέσως όλους αυτούς τους δημοσιογράφους. Και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα πρέπει να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών και θα πρέπει να αυξήσουμε τις κυρώσεις ε, έναντι εκείνων στο Μπουρούντι που ε, κάνουν όλες αυτές τις ε, πράξεις. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία ε, λειτουργούν και θα πρέπει να λειτουργούν. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Και τώρα το λόγο έχει ο Γιάνν Κριστόφ Όιτεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Το Μάιο έχει εκλογές στο Μπουρούντι και Στην ε, περίπτωση του Μπουρούντι ε, η κατάσταση έχει κλιμακωθεί εδώ και χρόνια και όχι μόνο εν ώψη των εκλογών όπως ήθιστε να γίνεται και καταστέλλονται δημοσιογράφοι, αντιφρονούνται οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων. Μπαίνουν στη φυλακή, δικάζονται ε, και πολλοί θανατώνονται, δολοφονούνται. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρέπει να στρέψουμε αλλού το βλέμμα, αντίθετα να υψώσουμε τη φωνή μας και να υπερασπιστούμε τους ανθρώπους αυτούς. Συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις ε, υπόθηκαν ε, ήδη από τους συναδέλφους ε, ε, Τσόνης και Αρενά και δεν θέλω να επαναλάβω αλλά να πω ότι θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να αφαιθούν αμέσως ελεύθεροι να τους δοθεί χάρη και υπό καμία προϋπόθεση, άνευ κανενός όρου. Αυτό είναι ξεκάθαρο και πρέπει να το πούμε κατηγορηματικά στο Μπουρούντι. Μπορεί κανείς ε, να έχει ε, διαφορετική άποψη, δεν είναι ένα έγκλημα αυτό, είναι κάτι που είναι αξιέπαινο και θα έπρεπε να το υπερασπιστούμε από πλευρά της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει λοιπόν να πούμε στο Μπουρούντι, αφήστε ελεύθερου ανθρώπους, ανθρώπου, δεν κάναν τίποτε κακό. Και θα πρέπει να αυξήσουμε τις πιέσεις ε, και να τις διατηρήσουμε ε, απέναντι στις αρχές του Μπουρούντι. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι διεθνής κοινότητα, να ε, φροντίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των πολιτών και η ελευθερία της έκφρασης να γίνονται σεβαστές ώστε να μπορέσουν φέτος να γίνουν σε ασφαλείς και δημοκρατικές συνθήκες αξιόπιστες εκλογές. Ευχαριστώ, Πρόεδρος εκ μέρου ε, του ΕΛΚ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κέλλη. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συζητάμε ξανά το θέμα του Μπουρούντι. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα και πριν και δεν έχουμε να πούμε τόσα πολλά πράγματα. Δεν είναι ευχάριστα. Υπάρχει έλλειψη ελευθεροτυπίας, και χρειάζεται να συζητούμε το θέμα αυτό σήμερα το πρωί. Το Μάρτιο 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε την υποστήριξη των οικονομική στην κυβέρνηση του Μπουρούντι. Μετά τι προεδρικέ εκλογέ διαμορφώθηκε αυτή η σχηματιστική κυβέρνηση. Την μποϊκοτάρισε ε, και η αντιπολίτευση και το παρατηρητήριο του ΟΗΕ. Καταδικάζουμε την καταστολή τη ελευθερία έκφραση και τη αυτοτύπη του Μπουρούντι του 2018 και το 2019 τα μέσα ε, καταπιέστηκαν και παρενοχλήθηκαν στις αρχές του Μπουρούντι, ε, τους αφαιρέθηκαν άδειες. Όπως και το BBC την άδειά του οι αρχές του Μπουρούντι, ε, συλλαμβάνουν ακόμα ανεξάρτητους μουσιογράφους και στο δίκτυο για την ευθεροτυπία το Μπουρούντι είναι στην 159η θέση από τις 180 χώρες το 2019 και αυτό τα λέει όλα. Η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του τύπου και όλα αυτά καταστέλλονται εκλογέ θα γίνουν το κοινοβουλευτικές του 2020 και αυτό θα είναι τεράστιο θέμα. 22 Οκτωβρίου 2019 η αστυνομία του Μπουρούντι συνέλαβε τέσσερις δημοσιογράφους σαν συνενόχου ε, και απειλή, σε απειλή κατά του κράτους και σε 30 μέρε θα ληφθεί απόφαση. Είναι σημαντικό γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ύπατος εκπρόσωπο αμελητή να κινηθούν και να κάνουν τα κατάλληλα διαβήματα και να μην ε, τελικά εφαρμοστεί η ποινή 15 ετούς, 15 κάθερξης. Και θα πρέπει να συνεργαστούμε και την κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής και την Αφρικανική Ένωση για να προστατεύσουμε τον πληθυσμό του Μπουρούντι. Μόνο βελτίωση μπορούμε να επιφέρουμε, διότι η κατάσταση είναι φρικτή σε αυτή τη φάση εκεί. Ευχαριστώ πολύ και εν ονόματι των σοσιαλιστών η κυρία Ιζαμπέλ Σάντος έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αν πατήστε όμως το μικρόφωνο σας κυρία Σάντος. Ναι, τώρα λειτουργεί, ναι. Η ελευθερία έκφρασης στο Μπουρούντι έχει πληγεί. Οι δημοσιογράφοι και ο οδηγός τους ε, που συνελήφθησαν τέλη 2019 είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις παραβίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Τα Ηνωμένα Έθνη, μέσω του Γενικού Γραμματέα, αλλά και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δημοσίευσαν τις σημαντικές ανησυχίες, δημοσιοποίησαν τις σημαντικές ανησυχίες που υπάρχουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα ε, και για την ελευθερία έκφρασης, ε, ε, αυθαίρετες συλλήψεις, δολοφονίες, ε, βασανιστήρια, όλα αυτά αναφέρονται από τα Ηνωμένα Έθνη σε ένα κλίμα απόλυτης ατιμορρησίας στη χώρα αυτή. Οι, παρα... παραβίασης ε, δικαιωμάτων έκφρασης που συζητούμε σήμερα είναι μόνο ένα παράδειγμα αυτής της ευρύτερης καταστολής και πραγματικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποδοκιμάσουμε. Ζητούμε την απελευθέρωση των τεσσάρων δημοσιογράφων που συνελήφθησαν στα τέλη του προηγούμενου έτους ο κύριος Μουκουσέση, η κυρία Ρημάδα, η Κριστίν Καμισάδη, Καμισάγη, καθώς και ο οδηγός τους, ο Αδόλφο Μασαμπαρακάση και να ζητήσουμε, τις, να, ζητήσουμε να υπάρξουν συνθήκες ε, για ελεύθερες και δίκες εκλογές. Ε, και ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για τη Ρηνιού, η κυρία Χαράντσοβα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Τον Μπουρούντι αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις τα τελευταία πέντε χρόνια όσοι θεωρούνται ε, στην αντιπολίτευση οι αντιφρονούντες ε, εξαφανίζονται, βασανίζονται, δολοφονούνται. Οι ε, δημοσιογράφοι απειλούνται ή συλλαμβάνονται αυθαίρετα. Υπάρχει απόλυτη ατιμορρησία για αυτούς που διαπράττουν αυτές τις πράξεις. Χιλιάδες πρόσφυγες από τον Μπουρουντή φεύγουν για να αποφύγουν αυτή την κρίση και την ανθρωπιστική ένδυα προεδρικές εκλογέ φέτος ε, ενδέχεται να δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερη αστάθεια και ενδεχόμενη βία. Υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι αρχίζουν να στρατολογούνται από ένοπλες ομάδες ε, αντίδραση. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσει η κυβέρνηση του ε, πολίτες, τους, να επικρατήσει τα δικαιώματά του. Θα πρέπει να απελευθερωθούν οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στη φυλακή και οι ακτιβιστές κοινωνία των πολιτών. Πρέπει το κράτος δικαίου να γίνει σεβαστό, η δημοκρατία να ενδυναμωθεί. Ιδάλω ε, θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση τη κατάσταση. Υπό αυτέ τι συνθήκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε άλλη επιλογή από το να διακόψει την οικονομική βοήθεια προς την κυβέρνηση του Μπουρούντι. Δεν πρέπει όμως να καταλήψουμε το λαό του Μπουρούντι. Πρέπει να ενισχύσουμε την ε, συνεργασία για την ανάπτυξη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βρεθεί, για να λάβει η χώρα μια ειρηνική εκλογική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για τους πράσινους ε, το λόγο έχει η Άλλη Σκούνκε για ένα λεπτό. Οι επιθέσεις που γίνονται κατά του τύπου και ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουμε προσοχή όσον αφορά την κατάσταση στο Μπουρούντι ούτως ώστε να μην αποσιωπούμε αυτά τα συμβάντα. Όμως η δίωξη των δημοσιογράφων θα πρέπει να σταματήσει και η κυβέρνηση θα πρέπει να απελευθερώσει κάθε δημοσιογράφο. Εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα και μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε αυτό να συμβεί. Θέλουμε να καλέσουμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξουν την Ένωση των Δημοσιογράφων, τα κινήματα των γυναικών στον Μπουρούντι, τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ άλλων, πρέπει να εφαρμόσουμε πραγματικά τη Συμφωνία της Αρούσα και θα πρέπει να υποστηρίξουμε και την κοινωνία, ούτω ώστε να υπάρξει διάλογος σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Εν ονόματι του ECR. Ρίτσαρτ Σαρνέσκη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ε, έχω πάει στο Μπουρούντι και στις γειτονικέ χώρες, στη Ρουάντα, παραδείγματο χάρη, στην Τανζανία και στην ε, Δημοκρατία του Κόγκο. Πιστεύω ότι γνωρίζω την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Είναι μια χώρα με μακρές ιστορικές παραδόσεις. Ήταν το βασίλειο των Τούτσι που είχε δημιουργηθεί ακόμα πριν δημιουργηθούν κάποια κράτη στην Ευρώπη. Είναι, σημαντικό να παρέμβουμε λοιπόν να στηρίξουμε την ελευθερία των δημοσιογράφων, να ζητήσουμε την άνοιξη, να διεξαχθούν ελεύθερες εκλογές. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι σημαντικά πέραν αυτών. Πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις, αναστέλλοντας την οικονομική βοήθεια για μια χώρα που δεν σέβεται ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Φάμπιο Μάσιμο Καστάλτο. Αλλά δεν τον βλέπω να είναι στην αίθουσα. Οπότε, δίνω το λόγο στον κύριο Κάλλος Ζουρίνιο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πλησιάζουν οι εκλογές στο Μπουρούντι και αυτό αυξάνει την ένταση. Βλέπουμε και πώς λειτουργεί το κράτος ουσιαστικά με την αστυνομική βία για να περιοριστούν τα δικαιώματα των πολιτών όπως η ελευθερία έκφρασης δεν λαμβάνει υπόψη ε, τα Ηνωμένα Έθνη κυβέρνηση του Μπουρούντι, ούτε τη ΜΚΟ. Η ελευθερία έκφραση λοιπόν κινδυνεύει. φυλακίσει ε, φυλακίσεις ε, και γενικότερα ένας λόγος επίσημος που είναι επιθετικό απέναντι στην ελευθερία έκφραση. Πολλοί δημοσιογράφοι που να κάνουν τη δουλειά τους. Θα πρέπει οι μελλοντικέ εκλογέ να είναι δίκαιε και δημοκρατικέ. Κάνω μια έκκληση προς την υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, και προς τους διπλωμάτες μας. Οι δράσεις των Εθνών ε, πρέπει να ξεκινήσουν για να μπορέσουμε να τιμωρήσουμε όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπουρούντι. Η συμφιλίωση, η ειρήνη στον Μπουρούντι είναι απαραίτητη για να μπορέσει να αναπτυχθεί η χώρα αυτή και να φύγει από αυτό το φαύλο κύκλο στον οποίο έχει περιέλθει. Ε, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα δίνω το λόγο στον Φιλ Μπένιον για δύο λεπτά από του Renew. Ο λαό του να εξακολουθεί να υποφέρει από, από των ποινών δικαιωμάτων. Στην έκθεση των ΗΠΑ του περασμένου Σεπτέμβρη φαίνεται ότι η αστυνομία, οι μυστικέ υπηρεσίε, ακόμα και η νεολαία του κυβερνητικού κόμματο είναι υπεύθυνοι για τι δολοφονίε, τι εξαφανίσει, τι αυθαίρετε συλλήψει ε, αντιφρονών πολιτικών και των οικογενειών τους ένα από τα πρώτα βήματα ε, για να μπορέσει να υπάρξει λογοδοσία είναι η ελεύθερη έκφραση, η ελευθερία έκφρασης. Όμως και αυτή η ελευθερία έκφραση βρίσκεται υπό ε, επίθεση. Το BBC του αφαιρέθηκε η άδεια από τις αρχές του Μπουρούντι. Δεν μπορούν οι πολίτες, ε, απαγορεύεται στους πολίτες να δίνουν πληροφορίες στο BBC. Ακόμα και τα παιδιά δεν είναι ασφαλή από τη δίωξη τέσσερες μαθήτριες ε, συνελήφθησαν επειδή έπαιζαν ε, με την εικόνα ε, του Προέδρου. Πιο πρόσφατα ε, συνελήφθησαν ε, τέσσερις δημοσιογράφοι από μία οργάνωση τύπου και ο οδηγός τους και κατηγορούνται με, και απειλούνται με ποινέ έω και 15 έτη μόνο και μόνο, και μόνο επειδή ασκούν το δικαίωμα ελευθερία έκφραση. Πρέπει να πιέσουμε για να πλεθρούν αυτοί, οι δημοσιογράφοι, να σταματήσει η δίωξη την ανεξάρτητη των μέσων ενημέρωση και των πολιτικών τη αντιπολίτευση και να επανέλθει η ελευθερία έκφραση. Έχει υπογράψει στον Μπουρούντι ε, την Διεθνή Συμφωνία για τα ε, πολιτικά δικαιώματα μεταξύ των οποίων ε, υπάρχει και ελευθερία έκφραση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό έτσι ώστε οι μελλοντικέ προεδρικέ εκλογέ να είναι ελεύθερες και δίκαιες. Είναι και ο καλύτερος δρόμος για μια ειρηνική και αμυγός δημοκρατική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει ο Νέιθαν Γκίλ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, είμαστε εδώ και συζητούμε την ελευθερία έκφρασης στο Μπουρούντι. Εγώ όμως δεν μπορώ να εκφράσω ε, την δική μου άποψη βάζοντας το σημαίακι πάνω στο έδρανό μου. Βάζουμε ε, μαθήματα ε, σε άλλους και δίνουμε όταν καταστέλουμε εμείς και αρνούμαστε εδώ στους συναδέλφους μας το δικαίωμα υπερήφανα να επιδείξουν τις εθνικές τους σημαίες. Τι φοβάστε. Ναι, ας βοηθήσουμε άλλους να βελτιώσουν ε, τις χώρες τους, αλλά ας ε, τακτοποιήσουμε και τα του οίκου μας. Εμείς οι Βρετανοί θα πάρουμε μαζί μας τα σημαίακια μας και τις σημαίες μας ε, και θα την κάνουμε από εδώ. Μην είστε εσείς υποκριτές όμως, αφήστε τους συναδέλφους σας να μπορούν ελεύθερα να εκφράζονται όπως και τους ψηφοφόρους τους και την ταυτότητά τους και να μπορούν να κρατάνε πάνω στο γραφείο τους και στο έδρανό τους τη σημαία της χώρας. Ευχαριστώ. Η κυρία Νίνα Γκίλ. Έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μετά από την ε, προηγούμενη παρέμβαση δυσκόλευα με παρτολό αλλά τέλος πάντων θα εστιάσω στο Μπουρούντι ε, και στις, ε, στους δημοσιογράφους Κριστίν Καμικά, Ζεγνές Νιουντιουμπούσα, Τέρας Μπονζένση και Ιζίτ Καριμάνα, τέσσερις μεσόρες που κάναν τη δουλειά τους και καλούσαν την κυβέρνηση να λογοδοτήσει. 15 χρόνια φυλακή ε, τους περιμένει. Υποτίθεται ότι υπονόμευαν την κρατική εσωτερική ασφάλεια. Όμως ε, ουσιαστικά ο στόχος είναι να μην γνωρίζει ο έξω κόσμος ε, σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γίνονται στο Μπουρούντι. Στις ερωτήσεις μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, περιλαμβάνει σε εξής. Τι θα κάνει ώστε να απελευθερωθούν αυτοί οι τέσσερι δημοσιογράφοι, πώ ε, θα ασκήσετε ε, αυτά τα πιέσεις που σα δίνουν η δυνατότητα μάλλον τα 400 εκατομμύρια που δίνετε ω επίσημα αναπτυξιακή και πώ θα βοηθήσετε ενώπιση των εκλογών του Μαΐου ο πρόεδρος να προστατεύσει έστω ότι έχει απομείνει από την ελευθερία έκφραση στον Μπουρούντι και να γίνουν ελεύθερες ειρηνικές εκλογές. Ίσως είναι η τελευταία μου παρέμβαση στην Ολομέλεια, αγαπητή πρόεδρε. Ήταν τιμή, ήταν προνόμιο να έχω τη δυνατότητα να μιλήσω για άλλους που δεν μπορούσαν να το κάνουν. Χρησιμοποίησα αυτή την πλατφόρμα για να μιλήσω κατά το παραβιάσεων των δικαιωμάτων στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δυνατότητα. Εμείς ευχαριστούμε τον πρόεδρος, και Μπάλτ, έχει τώρα το για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η ελευθερία έκφραση, η ελευθερία λόγου είναι μια πολύ σημαντική αξία που έχει να κάνει με την δημοκρατία. Μας βοηθά να ξέρουμε την αλήθεια, εξασφαλίζει την ε, αυτονομία ε, την ανεξαρτησία σε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δυστυχώ οι αρχέ του Μπουρούντι σήμερα δεν επιτρέπουν την ελευθερία λόγου και χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Όσοι δεν προσπαθήσουν να περάσουν τι προφορές εκτό συνόρων βασανίζονται, βιάζονται, εκτελούνται, ενίοτε ή καταδικάζονται σε ισόβια. Δεν σέβεται ε, τον νόμο ε, τον Μπουρούντι. Δεν υπάρχει δημοκρατία στη χώρα για να υπάρχει κάτι πολύ εύθραυστο. Η Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθούν την κατάσταση, ιδίω εν ώψη των εκλογών, για να μην υπάρξει χειραγώγηση και για να υπάρξει ειρήνη, ελευθερία λόγου και δημοκρατία στη χώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Καστάλντο έχει το λόγο τώρα. Για Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το 2020 μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα έτος μεγάλων αλλαγών για τον Μπουρούντι. Επιτέλους, στι 20 Μαΐου θα γίνουν οι εκλογέ οι προεδρικέ και οι κοινοβουλευτικέ. μετά από μια περίοδο φρικτή που ξεκίνησε με τις αφιζητούμενε εκλογές του 2015 μεταξύ των Μπορούντι παραμένει θέατρο παραβιάσεων σοβαρότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος Κουρουτζίτσα, διέπραξε εγκλήματα ε, για να διατηρηθεί στην εξουσία κατά τη βούληση του λαού. Εματηρή καταστολή των διαδηλώσεων εφάρμοση. Σφαγέ έγιναν και εξοδικαστικέ εκτελέσει ε, μελών τη κοινωνία των πολιτών. Την 1η Μαου του 2019 ξεκίνησε μεγάλη περίοδο ε, δολοφονιών πολιτικών και απειλών κατά των αντιπολιτευόμενων ο χώρος για τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών όλο και περισσότερο περιορίζεται και δέχονται παρενοχλήσεις και απειλές και διαδικασίες δίκες εικονικές στη δημοσιογράφη. Πρέπει να εξάσουμε ανησυχία για εξελίξει. εξελίξεις που βλέπουμε πόσο αντιδημοκρατική μπορεί να είναι η φύση των επερχόμενων εκλογών. Πώς μπορούμε να κοιθούμε ε, ισότιμη εκλογική ε, αναμέτρηση υπό το φως τέτοιας καταστολής των ανεξαρτήτων μέσων ενημέρωσης. Το Μπουρούντι χρειάζεται πολιτική λύση διαρκείας. Αλλά η παρούσα κυβέρνηση δεν σέβεται τις διεθνείς συνθήκες. Συμφωνία του Ρούσα του 2000 και το Σύνταγμα του Μπουρούντι δεν σέβεται και δεν δέχεται καμία συμφιλίωση, τίποτα για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη δεν δέχεται. Πρέπει να εισακουστεί η φωνή τη Ευρωπαϊκή Ένωσης τώρα περισσότερο από πρωινή. Πρέπει να γίνουν σεβαστέ ε, ε, η συμφωνία του Κοτονού να γίνει συμβαστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνεί άλλε συνθήκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κύριε Βουλευτά, μπορείτε να φορέσετε τα ακουστικά σα, Δέχεστε μια ερώτηση στα πλαίσια τη διαδικασία τη γαλάζια Κάρτα. Ναι, βλέπω. Ο κ. Τόμισλαφ Σόκολ έχει μια ερώτηση και δίνω 30 δευτερόλεπτα για την ερώτηση. Καλώ, ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ συνάδελφοι. Αναφερθήκατε στα προβλήματα στον Μπουρούντι, αλλά δεν είναι η μόνη χώρα όπου τέτοια πράγματα λαμβάνουν χώρα, κυρίω στην Αφρική. Τα συζητάμε πολύ εδώ στο Κοινοβούλιο αυτά τα θέματα. Τι πιστεύετε πραγματικά, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε πραγματικά να επηρεάσει τα θέματα που συζητούμε σε αυτέ τι χώρε, ούτω ώστε ε, να χορηγείται η αναπτυξιακή βοήθεια σωστά. Πώς μπορεί να έχει ενιαία φωνή η Ευρώπη για θέματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πώς μας ακούεται σε παγκόσμιο προσκήνιο η Ευρώπη και μιλάμε μια φωνή. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Καστάλτο να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ για τη σημαντική ερώτηση. Λέω κύριο Καστάλτο, καταρχάς να σας πω ότι αληθεύει δεν είμαι η μόνη χώρα που υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό τώρα από ποτέ να ζητήσουμε να γίνεται σεβαστή η ρήτρα για ανθρώπινα δικαιώματα της Συμφωνίας του Κοτονού που ποτέ πραγματικά δεν εφαρμόστηκε και πάνω απ' όλα θα πρέπει να όχι μόνο να στείλουμε τη συνεργασία μας και τα χρήματα που δίνουμε στη συνεργασία αλλά να εφαρμόσουμε και στοχευμένες κυρώσεις κατά των υπευθύνων των φρικαλαιοτήτων μιλάμε για τον Μπουρούντι όπου έχουμε και καλυμμένη γενοκτονία διότι υπάρχει ακόμα σύγκρουση μεταξύ Ρούντου και Τούτσι στη χώρα όπως έγινε και στη Ρουάντα αλλά να πω επίση ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα πίεση και να έχουμε ενιαία θέση ε, των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάποια κράτη-μέλη δικά μα να διαπραγματεύονται πισόπλατα, μη σεβόμενα την επίσημη θέση του ΙΠΑ του εκπροσώπου και βεβαίω την επίσημη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ε, έχουμε καταρχάς τον κύριο Πόσπισιλ που θα λάβει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τη συζήτηση. Συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους. Η κατάσταση στον Μπουρούντι πραγματικά είναι κρίσιμη και ευχαριστώ τους συντάκτες αυτού του εγγράφου. Το περιεχόμενο αυτού περιγράφει την παρούσα κατάσταση. Σε έξι μήνες θα γίνουν δύο εκλογές, οι προεδρικές και οι βουλευτικές στον Μπουρούντι και θα πρέπει να συζητήσουμε κύριε Επίτροπε από εσά μέσω διπλωματικής οδού με οικονομικά μέσα να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι εκλογές να εξελιχθούν δημοκρατικά διότι μπορούμε να επαναλαμβάνουμε πόσο τραγικά είναι τα πράγματα και πώ αντιμετωπίζονται οι δημοσιογράφοι στον Μπουρούντι, αλλά στόχο μας θα πρέπει να είναι να κάνουμε τα μέγιστα, ώστε το Μάιο οι εκλογές να είναι στο μέτρο του δυνατού δημοκρατικές και αν ο πρόεδρος ο παρόν δεν θέλει πλέον να ε, είναι υποψήφιο, αντίθετα λένε οι αναλυτέ, θα είναι εκ νέου υποψήφιο. Αυτό θα αντιβαίνει το σύνταγμα του Μπουρούντι αν είναι εκ νέου υποψήφιο ο παρόν πρόεδρο. Θα πρέπει να κάνουμε τη δυνατόν να είναι δημοκρατικέ εκλογέ που θα διεξαχθούν. Ευχαριστώ. Όγκεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι εδώ όμως. Παρακαλώ. Κύριε Λόπεθ όχι. Ο Έουγεν Τόμακ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να μιλήσω για το θέμα αυτό διότι θεωρώ ότι είναι πολύ καλό ότι γίνεται αυτή η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία έκφρασης όταν δεν γίνονται σεβαστά σε αυτές τι ελευθερίες ανά τον κόσμο, διότι εκατομμύρια άνθρωποι κοιτάζουν με ελπίδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε το θεσμικό όργανο εκείνο που υπερασπίζεται αυτές τις αξίες. Και αυτές ήταν και οι αρχές ε, ε, όσων δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν του δημοσιογράφου οι οποίοι εργάζονται, ασκούν το επάγγελμό τους ε, σε, σε χώρες όπου η δημοκρατία είναι εύθραυστη. Έχουμε το πιο ευρύ διπλωματικό σώμα του κόσμου. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης λοιπόν πρέπει να συμμετάσχει πιο ενεργά. Έχουμε, παραλαμβάνω, το μεγαλύτερο δίκτυο διπλωματών παγκοσμίω και περιμένουν πολλά οι πολίτες, έχουν, εναποθέσει ελπίδε ελπίδες σε εμάς. Ε, Αγγιλάρ έχει το λόγο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τον περασμένο Νοέμβρη είχα την τιμή να συμμετάσχω στην ε, συνάντηση την κοινοβουλευτική Αφρικής, Καραβικής και Ειρηνικού όπου μιλήσαμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχέσεις της με τις χώρες αυτές μετά τη Συμφωνία του Κοτονού. Σε αυτήν την κοινοβουλευτική συνέλευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπαν, ανέφεραν ότι το Μπουρούντι που είναι ε, όμορη χώρα με την Ρουάντα που έζησε αυτή τη γενοκτονία της δεκαετίας του 1990 παραβιάζει το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού λόγω της καταστολής που συνεχίζεται στη χώρα αυτή. Το Μπουρούντι είναι από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου. Το 50% του προπολογισμού του εξαρτάται από εξωτερική ενίσχυση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει την ενίσχυσή της από 90 σε 120 εκατομμύρια ευρώ. Ανθρωπιστική ενίσχυση σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε λοιπόν ε, ε το καθήκον να απαιτήσουμε οι εκλογές που θα λάβουν χώρα φέτος, οι προεδρικές, οι βουλευτικές και τοπικές, ε, να μην ε, επιτρέψουν την καταστολή των ακτιβιστών, των δημοσιογράφων ή εξαφανίσεις, οι συστηματικές τα σημερινά βασανιστήρια, οι αυθαίρετε συλλήψει, έχουμε τη δυνατότητα να το πετήσουμε αυτό και το καθήκον. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Επίτροπο, στον κύριο Λέναρτσιτ έχει το λόγο. Στον όνομα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ Πρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη. Συμμερίζομαι τι ανησυχίε σα ό,τι αφορά την κατάσταση στον Μπουρούντι. Σα θυμίζω ότι τον περασμένο Δεκέμβριο το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την ανάγκη να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα με βάση το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού μέτρα κυρώσεων απέναντι στον Μπουρούντι. Πρέπει ε, να είναι ψηλά στις προτεραιότητες ε, της ατζέντα μας το θέμα του Μπουρούντι, να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας στα, στα Ηνωμένα Έθνη, την Αφρικανική Ένωση, τις τοπικές αφρικανικές, περιφερειακές αφρικανικές οργανώσεις. Ε, έχουμε σημάδια ότι μπορεί να αυξηθεί η ένταση εν ώψη των εκλογών του 2020 οι παραβιάσεις ε, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των, των ε, θεμελιών ελευθεριών, ιδιαίτερα το δικαίωμα έκφρασης, το δικαίωμα συνάθρησης. είναι όλο και πιο έντονες αυτές οι πιέσεις. Η, η σύλληψη των τεσσάρων δημοσιογράφων αναφέρθηκε από πολλούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί πολύ στενά την υπόθεση αυτή στη σχέση της με τις αρχές του Μπουρούντι. που έχουμε θέσει το θέμα και είμαστε και σε συντονισμό με τους εταίρους μας. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε την υπόθεση αυτή. Η Ερευνητική Επιτροπή για τον Μπουρούνι στην έκθεση του Σεπτέμβρη ε, αναφέρεται ότι υπάρχει ένα κλίμα φόβου και απειλών προς οποιονδήποτε δεν υποστηρίζει το κόμμα που είναι στην κυβέρνηση. Η Κομισιόν έχει σηκώσει κόκκινες σημαίες και για μια σειρά παραβιάσεων που έχουν λάβει η χώρα μεταξύ των οποίων ε, υπάρχουν και διεθνή εγκλήματα. Δεν πιστεύω πάντως ότι μπορούμε απλά να, θεωρούμε, να θεωρήσουμε ε, ότι είναι αναπόφευκτο τα πράγματα, ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Αυτό δεν είναι προς συμφέρον κανενός και σίγουρα δεν είναι προς συμφέρον του Μπουρούντι και του πληθυσμού του. Θέλω να σας διασφαλίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία πρόθεση ε, να ε, εγκαταλείψει τον Μπουρούντι. Μέσω της ανάπτυξης για τη συνεργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται στη χώρα αυτή συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, με τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πιο ανθεκτικό κλίμα για τον πληθυσμό. Τους επόμενου μήνες εν των εκλογών θα είναι κρίσιμο το Μπουρούντι να εξασφαλίσει μια αξιόπιστη, διαφανή και συμπεριληπτική εκλογική διαδικασία να ανοίξει ένα χώρο πολιτικό, ένα χώρο για κοινωνία των πολιτών, να σταματήσουν οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να σταματήσει η ατιμορρησία ο σεβασμός και του πνεύματος και του γράμματος της Συμφωνίας Τσαρούντα είναι κρίσιμη. Ε, βεβαίως ε, υπάρχουν πολλά στοιχεία πάνω στα οποία πρέπει να οικοδομήσουμε. Ένας κώδικας συμπεριφορά που, που να υποστηρίζεται από τα πολιτικά κόμματα και βεβαίως υπάρχουν οι ανακοινώσει, ε, η ανακοίνωση του Προέδρου ότι δεν πρόκειται να είναι ξανά υποψήφιος για τέταρτη φορά. Εάν ακολουθεί αυτή η οδός στον Μπορούντι, τότε μπορεί να υπάρξει και βοήθεια και στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο Λέναρ Σίτς. Υπάρχουν έξι σχέδια ψηφίσματο. Κλείνει η υπόθεση αυτή. Τα ψηφίσματα αυτά θα τεθούν σε, σε ψηφοφορία σήμερα. Κλείνει λοιπόν το θέμα αυτό για σήμερα, η συζήτηση. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο τη διάταξη. Συζήτηση για την Ιγυρία και ιδίω ε, για τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στη χώρα αυτή. Σας θυμίζω για άλλη μια φορά ότι για να πάρετε το λόγο, ε, για να ζητήσετε μπλε κάρτα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε είτε την παραδοσιακή οδό είτε την ηλεκτρονική οδό. Υπάρχουν ε, οι σχετικές οδηγίες στην είσοδο. Δίνω τώρα ευθύ αμέσω το λόγο στην κυρία Ασίτα Κάνκο για ένα λεπτό. Bring φέρετε πίσω τα κορίτσια μας. Το θυμάστε αυτό το hashtag πριν 6 χρόνια που συσπήρωσε τον κόσμο ε, και απέθεσε την έκκληση ε, κατά τη Ισλαμιστική Οργάνωση, τη Τρομοκρατική Οργάνωση Μπόκο Χαράμ για να απελευθερώσει μαθήτρε που είχε απαγάγει. Πραγματικά είναι σπαρακτικό να σκέφτεται κανεί ότι πάνω από 100 κορίτσια δεν έχουν ακόμη επιστρέψει στα σπίτια του. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει, αυτή η μοίρα του για τι οικογένειέ του, για τι ίδιε. Ε, είναι η κυρία για πάρα πολλά χρόνια πλήττεται από την ε, εθνοτική και θρησκευτική βία. Προσπαθεί να αναπτύξει το οικονομικό δυναμικό. Ουσιαστικά αυτό όμως ξοδεύεται. Ενώ θα μπορούσε να είναι ένα ηγετικό παράδειγμα για την περιοχή. Καθημερινά όμως πεθαίνουν οι Γυριανοί από τη βία, από τον τρόμο. Κατομμύρια τρέχουν για τη ζωή τους ε, ή ζουν σε συνθήκες τρόμου. Πρέπει να στηρίξουμε τους Νιγηριανούς, να προωθήσουμε την ε, διεθνή συνεργασία και να προωθήσουμε μεταρρυθμίσεις για την ασφάλεια, για το στρατό και αλλού. Η αποφασιστικότητά μας, οι προσπάθειές μας μπορούν να βοηθήσουν ε, και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να αφιστούμε αυτών των προσπαθειών για να βοηθήσουμε τις γυναίκες ε, και να πάψει η τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έρικ Μάχαρκάρτ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που μέσα σε σύντομο χρονικό ε, διάστημα συμφώνησαν μαζί μας αυτό το εκτεταμένο ψήφισμα για να μιλήσουμε για την ανθρωπιστική ε, έκτακτη κατάσταση. 36.000 ε, ε, άνθρωποι έχουν στη ζωή τους από τη δράση της Μπόκο Χαραμετά. το Ιράν και το Αφγανιστάν στην τρίτη θέση στο δίκτυο για την τρομοκρατία η Νιγηρία. 2 εκατομμύρια εκτοπιστέντες και 7 εκατομμύρια χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα. Και ναι, καλό είναι να λέμε ε, και για τους χριστιανούς ε, που διώκονται, αλλά ε, επίσης πολύ καλά κάνουμε και διευκρινίζουμε στο ψήφισμά μας ότι αυτό που γίνεται στην Ιγυρία δεν είναι θρησκευτικό πόλεμος, ουσιαστικά έχει να κάνει με την διανομή του πλούτου των φυσικών πόρων και τελικά η κλιματική κρίση επηρεάζει και την οικονομική σταθερότητα και τις αντιπαραθέσεις της ε, πραγματικά έχουμε τη δράση των τρομοκρατικών οργανώσεων σε έφορες περιοχές, ε, εκεί που θα μπορούσαν να ζήσουν ε, σε αξιοπρεπείς συνθήκες οι Νιγηριανοί. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, δεν ξέρω, έχω το αίσθημα και ελπίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για την αναπτυξιακή πολιτική που πολύ συχνά ε, την καθορίζουν τα δικά μας συμφέροντα μέχρι στιγμής. Και καλό είναι που λέμε στο ψήφισμα ότι η αναπτυξιακή συνεργασία θα πρέπει να έχει ως στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας κυρίως και όχι άλλους στόχους θέλουμε ε, να φεύγουν λιγότεροι από την Νιγηρία, αλλά ε, δεν είναι τόσο απλό. Ε, δεν μπορεί να κλείσουν τα σύνορα και να ασκηθούν πιέσεις ε, και το είπε και η ανταποκριτή ε, της Ολλανδικής Εφημερίδας. Είναι πραγματικά κάτι στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο εκεί και όχι απλά να φροντίζουμε, να τους κλείνουμε το δρόμο για να μπορούν να, να φύγουν από εκεί. Πρόεδρος, ευχαριστώ να σας χαιρετήσω. Καλή σας μέρα και σε εσά και στου ε, ε, κάτω εκατομμύρια ανθρώπου που μα ακούνε. Ο κύριο Μπέργκ. Εγώ υποστηρίζω αυτό το ψήφισμα γιατί έχουμε τις διώξεις χριστιανών και ιδίως 26 Δεκεμβρίου ε, ε, την, ε, τον αποκεφαλιμασμό που είχαμε εκείνη την ημέρα είναι μια αποτρόπη βάρβαρη πράξη ε, και πραγματικά πρέπει να μιλούμε. Ε, μιλάμε για συστηματική εξόντωση χριστιανών αλλά δεν υψώνει αρκετά τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και νομίζω ότι ε, πρέπει να αρχίσουμε στο να αναγνωρίζουμε ε, αυτή την κατάσταση και σε αυτό το κοινό ψήφισμα γίνεται μια αρχή για να μπορέσουν να το κάνουν και άλλοι. Είδαμε για να επιθέσει σε βάρο ε, των χριστιανών, θεολοφονεί χριστιανών στο όνομα του Ισλάμ. Βέβαια δεν πρέπει να καλύπτονται αυτά από άλλα. Ε, υπάρχουν ε, χριστιανικές κοινότητες που διώκονται από τους Ισλαμιστές και αυτό δεν πρέπει να το κρύβουμε. Αποκεφαλίζονται γιατί ήταν χριστιανοί από την τρομοκρατική οργάνωση, δολοφονούνται με αποτρόπαιο, με βίαιο τρόπο χριστιανοί. Ε, υπάρχει πραγματικά έκτακτη ανάγκη ε, για την Νιγηρία, για την Ανατολική Αφρική. Πρέπει να προστατευτούν οι χριστιανοί που διώκονται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζωρίνιο έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ. Να επαναλάβω ότι αν κάποιο θέλει ε, να πάρει το λόγο στο τη, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ηλεκτρονικά το σύστημα το ηλεκτρονικό ή παραδοσιακά. Η βία που υπάρχει στην Ιγυρία από την Μπόκο Αράμ είναι πραγματικά τρομακτική. Δύο εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτοπισμένοι, εκατομμύρια άνθρωποι που βρίσκονται σε ανθρωπιστική κρίση, βία, ε, σεξουαλική βία κατά των γυναικών, έλλειψη εκπαίδευσης, ε, όλα αυτά λόγω αυτής της σύραξης, λόγω αυτού του φαύλου κύκλου ανασφάλειας και βίας. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις πραγματικά χρήζουν μιας ε, στρατηγικής ε, αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής προστατεύοντας ε, τους τοπικούς πληθυσμούς και τους χριστιανικούς και τους μουσουλμανικούς από τους φανατικούς Ισλαμιστές που δεν επιτρέπουν ε, ε, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πρέπει οι τοπικές οργανώσεις να υποστηριχθούν για να μπορούν να, να, με τη σειρά τους να κάνουν τη δουλειά τους, να υποστηρίξουν δηλαδή ιδιαίτερα τις γυναίκες, τις έγκυες γυναίκες, τα παιδιά. Υπάρχει και κλιματική αλλαγή η οποία επιδεινώνει την κατάσταση. Είναι σημαντικό λοιπόν μεσοπρόθεσμα να εργαστούμε και για πρόσβαση στους φυσικούς πόρους ε, στη χώρα αυτή. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό για την ειρήνη, αλλά και για την οικονομική σταθερότητα και κοινωνική σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Οι μεταναστευτικές ροές από την Ιγυρία και από τις προσυγητενικές χώρες δημιουργούν νέα προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν συντονισμένη δράση από την ε, διεθνή κοινότητα και με ενισχυμένη συνεργασία για να αντιμετωπιστεί βεβαίω η τρομοκρατία. Η καταπολέμηση οποιοδήποτε θρησκευτικής ακρότητας, ε, θρησκευτικού φωτομεταλλισμού. Αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα ε, και, σε, και εκεί και εδώ. Η κατάσταση στην Ιγυρία έχει να κάνει και με τη δική μας ασφάλεια. Όπου και αν ζούμε, αυτό που συμβαίνει στην Αφρικανική Ήπειρο επηρεάζει το σύνολο του κόσμου και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την ε, κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ουρμπάν Κρέσπο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Νιγηρία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στην Αφρική. Είναι άλλο ένα παράδειγμα μιας πλούσιας χώρας σε πόρους, όπου όμως ο μισός πληθυσμός ζει στη φτώχεια. Επιπλέον η βία στη χώρα αυτή είναι ακραία. Πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι είναι εκτοπισμένοι. Οι γυναίκες και παιδιά βιάζονται, είναι προϊόν εκμετάλλευση σεξουαλική. ε, κάποιοι φυλακίζονται από το κράτο, κάποιοι άλλοι απαγάγονται από την Μπόκο Αράμ. Το κράτο υπονομεύει την ανθρωπιστική βοήθεια ε, και την δράση των ε, ΜΚΟ μιλώντας ε, για καταπολέμηση τρομοκρατία. τρομοκρατίας. Δεν μπορεί οι τρομοκρατικοί νόμοι να καταργούν ελευθερίες και δικαιώματα. Πουθενά πρέπει να υπενθυμίσουμε στο κοινοβούλιο αυτό το σεβασμό του, ανθρωπισ... του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ε, και υπάρχουν οι αρχές, υπάρχει η αρχή της ουδετερότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας όταν προέρχεται από ευρωπαϊκούς πόρους. Ζητούμε ευθύνη και για τις, προς τις επιχειρήσεις μας για την για την καταστροφή του περιβάλλοντος και για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάμε στο Κοινοβούλιο για το New Green Deal τόσες μέρες. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι το Δέλτα του Νίγηρα είναι από τα πιο ε, μολυσμένα σημεία του κόσμου και λόγω των ευρωπαϊκών πολιεθνικών. Η φτώχεια, η ε, βία οδηγεί τους ανθρώπους αυτούς να, να φύγουν από τη χώρα, να βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Αυτές ε, τις οδούς της επικίνδυνης μετανάστευσης, ε, είναι ε, θύματα σκλαβιάς, βίας. Εμείς μιλάμε πάντα για ασφάλεια βέβαια και υψώνουμε τύχη. Πρέπει να δώσουμε έμφαση όμως στους λόγους, στις αιτίε, στις ευθύνες του συνόλου των ευρωπαϊκών πολιτικών και των δράσεων των ευρωπαϊκών πολυεθνικών στην Ιγυρία και σε άλλες χώρες του Νότου για να καταλάβουμε ακριβώς γιατί λαμβάνουν χώρα αυτές τις μεταναστευτικές ροές. Δεν αρκεί να εγκρίνουμε χρηματοδότηση της Αφρικής. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να αλλάξουμε 180 μοίρες τις, τις οικονομικές, πολιτικές και γεωστρατηγικές πολιτικές της Ευρώπης στην Ήπειρο αυτή. Κυρίες και κύριοι, δεν θέλουμε κενά λόγια, δεν θέλουμε φιλανθρωπία. Πρέπει να είμαστε συνεπείς στα λόγια μας και στις δράσεις μας. Πρέπει να αλλάξουμε ε, πολιτική στην Αφρική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για δύο λεπτά ο κύριος Τσεκόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Προτείναμε ένα ψήφισμα που αφορά την Ιγυρία από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά 11 χριστιανούς που εκτελέστηκαν. Φρικτή πράξη έλαβε χώρα. Οι ένοπλες δυνάμεις απήγαγαν τέσσερις ιεραποστόλους. Εάν συνδέσουμε αυτή την πράξη με άλλες βιοπραγίες, με βιασμούς που έχουν γίνει, με εκτοπισμό πληθυσμών και άλλες πράξεις κατά της ανθρωπότητας, βλέπουμε μπροστά μας να σχεδιάζεται ένα φρικτό τοπίο των τεκτενομένων στην Νιγηρία. Πάνω από 6.000 χριστιανοί δολοφονήθηκαν, καθώς και μουσουλμάνοι τα τελευταία πέντε χρόνια. 3.600 αγόρια και κορίτσια βρίσκονται σε στρατόπεδα ή κρατούνται σε φρικτές συνθήκες. Δύο εκατομμύρια άνθρωποι ε, εκτοπίστηκαν να κάποια στοιχεία από αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ιγυρία. Το κράτος δεν έχει κανέναν έλεγχο όσον αφορά ε, τις διάφορες ένοπλες ε, ομάδες. Το Boko Haram είναι ένας από τους μεγαλύτερους ε, οργανισμούς φορείς που κάνει φρικαλαιότητες και στοχευμένη γενοκτονία. Αυτές οι φρικαλαιότητες μπορεί να συγκριθούν μόνο με τους Ναζί ή φρικτά κομμουνιστικά καθεστώτα. Ε, παρόμοια συμβαίνουν στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Θα πρέπει η κυβέρνηση της Νιγηρίας ε, να ε, πιέζεται για αυτά τα θέματα, πρέπει να βρει λύσεις όσον αφορά αυτή την κατάσταση. Διότι δεν είναι δυνατόν μόνο να λαμβάνει βοήθεια, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζει την κατάσταση και τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπενιόν έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Η Νιγηρία πλησίασε πολύ στο να είναι χρεοκοπημένη, αποτυχημένη χώρα για δεκαετίε. Κυρίω λόγω μικροσυγκρούσεων μεταξύ των δύο βασικών κομμάτων. Αυτό οδήγησε σε πλήρη αποτυχία να αντιμετωπιστούν πραγματικά προβλήματα τη χώρα. Παραδείγματο χάρη Παρά κάποιε πρόοδου των στατιωτικών, η Μπόκο Χαράμ εξακολουθεί να απειλεί την ασφάλεια στι βορειοανατολικές περιοχές. Έχουμε απαγωγέ ε, βόμβες αυτοκτονία, επιθέσεις κατά πολιτών από την Μπόκο Χαράμ. Εξακολουθεί να δολοφονείται κόσμος. Και βεβαίω η Μπόκο Χαράμ επίσης ε, ε, στοχεύει τις επιθέσεις και αλλού, και στο Καμερούν και στο Τσάντ, και συνοριακά. Δεκαετίες ε, κοινοτικών ε, συγκρούσεων μεταξύ νομαδικών ομάδων στο κέντρο της χώρας εντατικοποιήθηκαν πρόσφατα και επιδίνωσαν ακόμα περισσότερο την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στη χώρα. Παιδιά και γυναίκε είναι οι πλέον ευάλωτε ομάδε αυτή τη συγκρούση. Τα παιδιά πολύ συχνά στατολογούνται από τι τρομοκρατικέ ομάδε, χρησιμοποιούνται σαν παιδιά στρατιώτε ή ε, σαν ε, βομβιστέ αυτοκτονία εκτοπίζονται πληθυσμοί λόγω όλων αυτών των βιοπραγιών. Η κοινωνία των πολιτών ηγείται της εκστατείας κατά των συλλήψεων, βασανισμών, αλλά θα πρέπει οι Νιγηριανές αρχές αυτές που θα έπρεπε να εγγυώνται το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και να ηγηθούν τις μάχη για αυτά. Ο πρόεδρος Μπαχάρη επανεξελέγει το 2019 υποσχόμενος ότι θα καταπολεμήσει τον βίο εξτρεμισμό των τρομοκρατικών ομάδων όπως η Μποκο και είναι η ώρα να επικεντρωθούν οι προσπάσεις κυβερνήσεως ώστε να τηρηθεί αυτή η υπόσχεση αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας ε, μία πλήρη στρατηγική. Η στρατηγική έχει θεσπιστεί αλλά δεν έχει εφαρμοστεί. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη πρέπει να βοηθήσουν μέσω τεχνικής αρρωγής. Τι ούτω τρόπος θα πρέπει να υποστηρίξουμε στα εναρά της προσπάθειας της Νιγηρίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα, εν ονόματι των πολιτικών ομάδων, εν ονόματι του ΕΛΚ, η συνάδελφος κυρία Ζόφκο έχει το λόγο για τις ε, μπλε κάρτες ε, μπορείτε αφού έχουν ε, εκφράσει τις απόψεις τους η εκπρόσωπη ομάδα να καταθέσετε αιτήσει. 80 εκατομμύρια χριστιανοί, οι μισοί Νιγηριανοί και υπάρχουν ιστορικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Βορρά και Νότου που έχουν οξυνθεί λόγω ε, της ε, ε, δράσης του Ισλάμ. Έχουμε την Μπόκο Χαράμ και άλλες χώρες και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις που τρομοκρατούν απειλούν χριστιανούς και τόπους λατρείας. Έχουν χάσει τη ζωή τους 6.000 χριστιανοί τουλάχιστον από το 2015 από τις τζιχαντιστικές ομάδες. Τελευταίες αναφορές της προηγούμενης εβδομάδας, 8 Ιανουαρίου, δείχνουν ότι στο χριστιανικό χώρο της κεντρικής Νιγηρίας, το βασικό, δεκάδες άμαχοι τη ζωή τους από μουσουλμάνους. Επίσης, ε, είδαμε και το Δεκέμβρη επιθέσεις ε, σε χριστιανικά χωριά. 30 άνθρωποι τουλάχιστον έχασαν τη ζωή τους. Ε, και η Ισλαμιστική οργάνωση της Δυτικής Αφρικής Islamic State θεωρεί ότι είναι, έχει αναλάβει την ευθύνη για την εξόντωση του Αλ ε, baqtadi λήψη μέτρων είναι απαραίτητη, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε παρκή μέτρα. Οι Νιγηριανείς ε, δυνάμεις ασφαλείας πολλές φορές ε, παραγνωρίζουν τα φαινόμενα αυτά, δεν τους δίνουν τη δέουσα σημασία. Υπάρχουν όμως ε, αυτές οι βιαιότητες απέναντι στις χριστικές μειονότητες. Θα πρέπει η Διεθνής Κοινότητα να αναγνωρίσει και τη δίωξη των χριστιανών. Είναι μια βαθιά θρησκευτική ήπειρος η Αφρική δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται οι θρησκείες για την παρότριση σε μίσος. Πρέπει η Ένωση να επενδύσει με οικονομική βοήθεια στο μέλλον της χώρας. Προστατεύοντας τις θρησκευτικέ μειονότητες, θα πρέπει η Ένωση επίσης να εστιάσει περισσότερο στον διαθρησκευτικό διάλογο, στις διπλωματικές της σχέσεις με τρίτες χώρες. Πριν από ένα μήνα, το Ευρωκοινοβούλιο έδωσε το βραβείο Ζαχάροφ ε, σε έναν μουσουλμάνο και έτσι ε, είναι συμβολική η κίνηση αυτή, αλλά δεν θα πρέπει ε, και τα άλλα εγκλήματα σε βάρος χριστιανών να τα κατονομάζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μέρο ομάδα Σοσιαλ και Δημοκρατών, κυρία Αρενά, Νιγηρία, επί πιο πολυπληθή ε, χώρα τη Αφρική, 200 εκατομμύρια. Και θα φτάσει στα 500 μέχρι το 2050. Είναι η μεγαλύτερη οικονομική νοτιοαφρικανική δύναμη. Και τη λένε γίγαντα τη Αφρική. Αντιμετωπίζει πολλέ εντάσει. Ε, Τάπαμε. Η Μπόκο Χαράμα ε, στα βορειοανατολικά. Στα βορειο ε, χιλιάδες ε, δολοφονίες, εκατομμύρια εκτοπίσεις. Επίσης, ε, γεωργοί και βοσκοί. Ε, εδώ δεν μιλάμε για μια αντιπαράθεση εθνοτική θρησκευτική, αλλά μια σύγκρουση λόγω τη κλιματική αλλαγή. Και οι βοσκοί έτσι έρχονται στα πιο πρόσφαρα εδάφη που, καλεί, που έχουν αυτή τη στιγμή οι γεωργοί. Επίση, κυκλοφορία όπλων από τη Λιβύη. Άρα ε, το Λιβικό επηρεάζει την περιοχή του Σαχέλ και την Ιγυρία. Και πρέπει να έχουμε μια απάντηση σφαιρική. Πρώτον, να υποστηρίξουμε ε, τη Λιβική λύση και ε, τον έλεγχο του εμπάργου όπλων. Σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μέταλλα, θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν αυτά για τον πληθυσμό. Η ΣΕΛ δέχτηκε επίθεση από τον τοπικό πληθυσμό γιατί είχε προκαλέσει σημαντική ρήπανση ε, και σφετεριζόταν τους πετρελαϊκούς πόρους. Επίσης έχουμε ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη για τις χιλιάδες θύματα. Έλεγχο επίση παγκόσμια εγκληματικότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό λόγω λάθρεμπορίων, ναρκωτικών, όπλων, ε, πορνεία. Όλα αυτά τα διευκολύνει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα που επιτρέπει τη φοροδιαφυγή στην Ιγυρία. Και τέλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει την Ιγυρία να τη κατά προτεραιότητα εταίρος ό,τι αφορά τη στρατηγική ένωση Αφρικής, διότι η σταθερότητα της Νιγηρίας είναι πολύ σημαντική για την περιοχή. Τσάτ, Καμερούν, ε, Νίγηρα 4.000 ε, ε, σύνορα, Σαχέλ, αλλά και ο κόλπος της Γουινέας που είναι ο χώρος διακίνηση και για όλη την Αφρικανική Ήπειρο. Πρέπει να παραμείνει λοιπόν για όλου αυτού τους λόγους προνομιακό εταίρος τη Ένωση η Νιγηρία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην ομάδα ε, Ρινιού και στον κύριο Ροντρίγκε Ράμου. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Νιγηρία είναι η τρίτη χώρα ε, που έχει πληγεί από την τρομοκρατία στον κόσμο. Είναι τρίτη στη λίστα μετά το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Μετά από τόσα χρόνια βίας από την ε, Μπόκο Αράμ υπάρχει επιδείνωση και λόγω της βίας της ε, εθνοτικής, ε, της θρησκευτική ε, μεταξύ μουσουλμάνων, χριστιανών και βεβαίως πιο πρόσφατα γίνεται και μια μάχη για αυτούς τους λίγους πόρους που υπάρχουν μεταξύ γεωργών και βοσκών, κτηνοτρόφων. Υπάρχει λοιπόν μια αύξηση των φαινομένων βίας, η κατάσταση επιδεινώνεται για τους πιο ευάλωτους, τις γυναίκες, τα παιδιά. Οι γυναίκες υπόκεινται σε γενικευμένες διακρίσεις, σε βία, σε ε, ε, υποχρεωτικούς γάμους, σε ιστρεκτομή. Ε, ζουν πραγματικά δραματικές στιγμές και τα παιδιά τα οποία στρατολογούνται από τους τρομοκράτες, χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις αυτοκτονίες, κρατώνται αλλά και από τους στρατιωτικούς ε, στην ε, ε, Νιγηρία κατηγορούμενη για συνεργασία με τρομοκρατία χωρίς στοιχεία. 3.600 παιδιά, τα μισά είναι κορίτσια, έχουν, είναι υποκράτηση και ο στρατός δεν επιτρέπει την πρόσβαση στα κέντρα κράτησης, στα στρατιωτικά. Ζητούμε λοιπόν από τις αρχές της Νιγηρίας τα παιδιά αυτά να μπορούν να τα επισκεφθούν μη στρατιωτικές αρχές. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το δικαστικό και αστυνομικό πλαίσιο πρέπει να προστατεύει ε, τους πολίτες και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους πολίτες. Ζητούμε λοιπόν από τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να υποστηρίζουν ε, σε τεχνικό επίπεδο την οικοδόμηση της ειρήνης στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Βλέπω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 η γενική αδιαφορία στην Ιγυρία οδηγεί σε χιλιάδες ε, ε, χριστιανού άνευ λύπης να, από του Ισλαμιστέ να δολοφονούνται και σφαγιάζονται. Τρομοκρατία δεν έχει ακόμα κρυζωθεί και αυτά που συμβαίνουν στην Ιγυρία ε, από τους ε, το αποδεικνύει. Εδώ και μερικέ μέρε, η Μπόκο Χαράμ έδωσε ένα βίντεο όπου σκοτώνονται 11 χριστιανοί φυλακισμένοι. Μία βίαιη δολοφονία που έγινε τα Χριστούγεννα πραγματική χειρονομία πρόκληση κατά τη ε, χριστιανοσύνη τη Δύση. Σύμφωνα με ανθρωπιστικέ οργανώσει, τουλάχιστον 30.000 είναι οι πολίτε που δολοφονήθηκαν και 30 εκατομμύρια οι εκτοπιστέντε από την αρχή τη επίθεση των τζιχαντιστών το 2009. Από πλευρά των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων που προωθούν την ειρήνη και την ανοχή και το σεβασμό των αμοιβαίων, τίποτα δεν έγινε συγκεκριμένο για να σταματήσει αυτή η συνεχή βαρβαρότητα. Κάθε μέρα τίθεται σε κίνδυνο η ζωή εκατομμυρίων αθών. Και το μόνο ε, του είναι χριστιανοί. Ο φανατισμό ο ισλαμιστικός ε, εξελίσσεται, διαδίδεται στη χώρα. Αλλά όχι μόνο Μποκοχαράμ ε, και ίση, αλλά και άλλοι, άλλε ομάδες ε, δολοφονούν ατιμωρητοί και δολοφονούν ανθρώπους σε χωριά. Θέλουν να εξισλαμίσουν δια της ισχύω στην Ιγυρία. Αυτή η μακρά μετοχυσία πρέπει ταχύτερο να σταματήσει. Δεν θα πρέπει να εθελοτυφλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προάσπιση των χριστιανών στην Ιγυρία σημαίνει προστασία τη Δύση από τον φανατισμό των Ισλαμιστών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το λόγο έχει ο και εκ ε, των συντηρητικών. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Μιλάμε για μια χώρα που έχει μακρά ιστορία, πάνω από χίλια χρόνια ιστορίας, ε, με μεγάλη ιστορία στον αφορά τη σιδηρουργία. Έχουμε πάρα πολύ όμορφα γλυπτά πύληνα που γινόταν στην αρχαιότητα. Μακρά ιστορία. Τι, θα, τι θέλει να κάνει αυτή τη χώρα η Μποκοχαράμ, πώς θέλει να την αλλάξει, τι κάνει με αυτή τη χώρα. Ε, τώρα ποια είναι η εικόνα που έχει αυτή η χώρα. Έχει υποφέρει αυτή η χώρα μετά από δολοφονίες χιλιάδων χριστιανών. Ε, νομίζω ότι η φωνή μας σήμερα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ε, ηχηρή. Δεν θα πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια βλέποντας αυτά που κάνουν οι τρομοκράτες κατά των χριστιανών και όχι μόνο κατά των χριστιανών είναι καθήκον μας να μιλήσουμε με δυνατή φωνή και να ζητήσουμε από τις αρχές της Νιγηρίας μία στεναρή καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο για... Τελειώσαμε τις παρεμβάσεις των ομάδων και περνάμε τώρα στους αγορητές, τους ε, μεμονωμένους και είχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε και με τη γαλάζια κάρτα. Μπορείτε να ζητήσετε παρέμβαση παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά, άμα θέλετε. Κύριε Βαντάλεν, για το ΕΛΚ έχετε το λόγο. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει τώρα να δράσει. Είναι απαράδεκτα αυτά τα δεινά που υφίστανται οι χριστιανοί στην Ιγυρία. Τώρα θα πρέπει να δράσει η εξωτερική μας πολιτική δεν ε, μπορεί να συγχυστεί αυτή η κατάσταση. Να το διατρανώσουμε προς την κυβέρνηση. Φτάνουν τα λόγια. Έργα τώρα. Έχουμε εμπορικές ε, συναλλαγές και άλλες σχέσεις με την Ιγυρία. Θα πρέπει αυτά να παγώσουν μέχρι να αρχίσει να προστατεύει τους χριστιανούς στην Ιγυρία και να πιάσει τον πόκο Χαράμ και οι επιχειρήσεις πρέπει να παίξουν το ρόλο τους. Δεν είναι δυνατόν να βγάζουν λεφτά στη χώρα αυτή ε, όπου ε, οργιάζουν η διαφθορά και η κατάχρηση εξουσίας. Έχει περάσει η ώρα των ωραίων λόγων και των μεγαλώστων δηλώσεων. Εδώ και χρόνια στενάζουν οι ε, χριστιανοί στην ε, Νιγηρία. 170 κορίτσια από το 2014 έχουν απαχθεί και 112 ακόμα λείπουν και όσες έχουν γυρίσει πολλές φορές ε, έχουν βιαστεί και ε, φέρουν ψυχολογικά τραύματα. Θα, πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Οι ομόθρησκοί μας ε, υποφέρουν. Ο επίσκοπος στην Ιγυρία καταδίκασε την κατάσταση και είπε ότι η μοναδική διαφορά ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Μπόκο Χαράμ είναι ότι το Μπόκο Χαράμ ε, βάζει βόμβες. Ο Πρωθυπουργός το 2015 δεσμεύτηκε να πιάσει τους τρομοκράτες. Αυτά είναι κενά λόγια. Τώρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υψώσει το ανάστημά της απέναντι ε, στο άδικο αυτό που γίνεται. Να τα βάλετε όλα στο ψυγείο μέχρι να συλληφθούν και να αντιμετωπιστεί αυτή η ελληνική κατάσταση με τον Μπόκο Χαράμ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαντάλεν. Βάλτε σας παρακαλώ τα ακουστικά σας γιατί ε, υπάρχει μια μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Ο κύριος Σόκολ θέλει να σας κάνει ερώτηση με την ε, γαλάζια κάρτα. Δέχεστε? Μάλιστα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφε, οι χριστιανοί διώκονται περισσότερο σε όλο τον κόσμο είναι ένα θέμα που δεν το συζητούμε στη Δύση, ούτε στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Γιατί? Γιατί έχουμε τις διώξεις κατά των χριστιανών και γιατί δεν ομιλούμε για αυτές τις διώξεις. Γιατί σαζόμεθα για τη δίωξη άλλων θρησκευτικών ομάδων και εμείς σαν ευρωβουλευτές τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε αυτή την αντίληψη του κοινού απέναντι σε αυτές τις διώξεις. Πρόεδρε, συμφωνώ πολύτως με τον συνάδελφο συστηματικά καταπιέζονται και δολοφονούνται οι χριστιανοί στην ε, Νιγηρία και τα μέσα ενημέρωσης δεν δίνουν σημασία. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η συζήτηση. Και υπάρχει μια διακομματική ομάδα ε, για τα θρησκευτικά θέματα και την ε, ανοχή τη θρησκευτική. Έχει επανασυσταθεί αυτό το Intergroup και θα φροντίσω αυτό το θέμα να προωθηθεί στην ημερήσια διάταξη οι διώξει, η διωγμοί κατά των χριστιανών, ιδιαίτερα στην Ιγυρία, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ξαναβάλτε παρακαλώ τα ακουστικά σας κύριε Βαντάλεν, γιατί έχουμε και άλλη ε, γαλάζια κάρτα από την κυρία Μαρία Αρενά, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Αρένα και Παρακαλώ. uh, please. Ε, σημειώνω αυτό ε, αυτά που λέτε προσεκτικά ότι θέλετε να ζητήσετε από τις επιχειρήσεις ε, να σέβονται με τη συμπεριφορά τους τον πληθυσμό. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το κόμμα σας και η ομάδα σας το ΕΛΚ συστηματικά καταψηφίζει μέτρα επίγουσας φρόνησης για ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ιγυρία και σε άλλες εμπόλεμες περιοχές η ομάδα σας ε, στο εξή θα αρχίσει να υπερψηφίζει ε, τα μέτρα που προτείνουμε για τις εταιρείε που δραστηριοποιούνται εκεί και θα πρέπει να έχουν τη δέουσα και αρμόζουσα συμπεριφορά. Έχετε 30 δεύτερα για να απαντήσετε κύριε Βαντάλεν. Σωστό είναι αυτό, συνάδελφε. Όταν μιλάμε για ε, ελευθερία της λατρείας, ε, θα πρέπει να ασχολούμαστε με τις χώρες που το κάνουν αυτό. Αυτό ισχύει για τη Σαουδική Αραβία, την Ινδία, την Ιγυρία και πάει λέγοντας. Αυτό που κάνετε εσείς και η ομάδα σας θα πρέπει να συνεχιστεί και στη δική μου ομάδα πραγματικά έτσι ώστε στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της θρησκευτική λατρείας να προοδεύσουμε. Ε, με χαρά να συνεργαστούμε, αν το κάνετε κι εσείς αυτό. Ε, πρόεδρος, και τώρα το λόγο έχει η κυρία Τζόνς, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταδικάζουμε πλήρως οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια και ιδιαίτερος και αυτήν στην Νιγηρία. Οι παραβιάσεις ε, δικαιωμάτων γυναικόπαιδων είναι παντού στον κόσμο. Είναι οι πιο ευάλωτοι, αυτούς στοχεύουν πάντα και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους προστατεύσουμε έναν τον κόσμο και ειδικά στην Ιγυρία. Είδαμε πολλά κορίτσια θύματα εμπορίας ε, ανθρώπων. Η πολυεθνική κοινή δύναμη πρέπει να κάνει τη δουλειά της ε, σε συνεργασία θεωρώ εγώ με την Αφρικανική Ένωση και όλους τους υπόλοιπους ε, παράγοντες της Αφρικανικής Υπήρου. Για την τελευταία μου ομιλία στο Στρασβούργο θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, όλους όσους εκπροσώπησαν την Ουαλία ανά ε, το ε, Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές και τους βουλευτές που πέρασαν και τις φιλοευρωπαϊκές ομάδες στην Ουαλία και σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο που εμφανίστηκαν μετά από το δημοψήφισμα. Ας συνεχίσουμε και μια μέρα θα επιστρέψουμε εδώ. Και προς τους συναδέλφους ευρωβουλευτές, ε, ήσασταν εξαιρετικοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και κουράγιο. Σας ευχαριστούμε και εμείς, λέει η Πρόεδρος. Περνάμε τώρα στην ομάδα Renew και την κυρία Χάρντσοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Μπόκο Χαράμ τρομοκρατεί την Ιγυρία εδώ και δεκαετίες. Ε, πάνω από 36.000 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί και η ισχύ του Μποκοχαράμου και άλλων τρομοκρατικών ομάδων αυξάνεται. Και βεβαίω οι επιθέσεις αυτές προκαλούν σοβαρή ανησυχία και η Νιγηρία αντιμετωπίζει έθνο-θρησκευτική και ενδοκινοτική βία. Επιπλέον ε, τα εγκλήματα αυτά μένουν ατιμόρυτα Χιλιάδες Νιγηριανοί φοβούνται για τη ζωή τους, φεύγουν από τα σπίτια τους και χρειάζονται βοήθεια, αλλά οι κίνδυνοι ασφαλείας έχουν οδηγήσει στην αποχώρηση των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Η κυβέρνηση της Νιγηρίας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να ανταποκριθεί στο καθήκον που έχει να προστατεύσει τους πολίτες της, να εγγυηθεί τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και να προστατεύσει το κράτος δικαίου. Σε μια κατάσταση που είναι ήδη άσταθής, η κυβέρνηση πρέπει να αποκλιμακώσει τις εθνοσκευτικές εντάσεις. Όμως η τρομοκρατία, όπως ξέρουμε, δεν έχει σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Νιγηρία και αλλού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μπίλντε τώρα από την ομάδα ID. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ισλαμική διείσδυση στη Δυτική Αφρική φαίνεται στην Ιγυρία να έχει βρει ε, ε, το πιο φρικτό απόγειό της. Ε, τρομοκρατικές επιθέσεις, ενοπτικές εκτελέσεις, απαγωγές, ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα. Ποιο αμφιβάλλει ότι η χριστιανική θρησκεία είναι η πιο διοκόμενη και στην Αφρική και αλλού κατά τα άλλα. Μα πώ θα μπορούσε να είναι διαφορετικά ενώ η διεθνή κοινότητα εξακολουθεί να ε, παραμένει ε, άπρακτη. Στο Σαχέλ μόνο η Γαλλία σηκώνει αυτό το σταυρό τη καταπολέμηση τη τρομοκρατία σε 8 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση όσο την Ευρώπη. Χειρότερο ε, φαίνεται η Δύση να παρεμποδίζει τις χώρες αυτές που αντιμετωπίζουν την τρομοκρατία με τρόπο ηρωνικό. Κυνηγάνε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ενώ έχουμε πάρα πολλές ε, ε, ενδείξεις ε, ότι χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Ο πόλεμος αυτός θα κερδιθεί μόνο από κυρίαρχα κράτη και από κανέναν άλλον. Σας ευχαριστώ. Μπίλαν από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η Νιγηρία είναι μια από τις πολυπληθέστερες χώρες της Αφρικής, 200 εκατομμύρια άνθρωποι. Και δυνητικά μια πολύ πλούσια χώρα, γιατί έχει τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου, παραδείγματος χάρη. Όμως, οι συγκρούσεις, η διαφθορά που πλήττουν την χώρα ε, σημαίνει ότι δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τον τεράστιο φυσικό πλούτο. 88 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στη φτώχεια. Το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας ε, είναι η τρομοκρατία. Η Νιγηρία είναι στην τρίτη θέση από το τέλος μετά από το Ιράκ και το Αφγανιστάν σε θέματα ασφαλείας. Οι χριστιανοί είναι η πιο διοκόμενη ομάδα στη χώρα. 20.000 άνθρωποι έχουν ήδη δολοφονηθεί λόγω της ε, πίστης τους. Απευθύνουμε έκκληση στον πρόεδρο από το 2015 να προστατεύσει τους πολίτες της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε μία μπλε κάρτα, την δέχεστε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την συζήτηση. Είναι μια απαραίτητη συζήτηση, πολύ σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη στάση το θέμα αυτών των τραγωδιών στην Αφρική, ειδικά στην Νιγηρία. Οι διώξεις των χριστιανών αναφέρθηκαν. Έχω λοιπόν ένα ερώτημα. Βλέπετε να υπάρχει κάποια δυνατότητα να ξεκινήσει μια συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο ε, γενικά για την κατάσταση των χριστιανών ανά τον κόσμο. Ε, ε, κοίταξτε, η μπλε κάρτα είναι για ερωτήσεις. Ε, αν είναι για δηλώσεις, ε, μπορείτε να πάτε στο KTI. Έχετε το λόγο, εν πάση περιπτώσει, για να απαντήσετε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο συνάδελφος. Οι χριστιανοί είναι η πιο διοκόμενη ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Σήμερα συζητάμε την Ιγυρία. Τον Οκτώβριο συζητούσαμε την Αίγυπτο. και εκεί πέρα διώκονται οι χριστιανοί. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια συζήτηση και σε αυτήν τη θητεία γενικά για την κατάσταση των χριστιανών στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τα Χριστούγεννα ανήμερα όντως ε, χριστιανοί αποκεφαλίστηκαν. 8 Ιανουαρίου ε, τέσσερις ε, φοιτητές θεολογική σχολή, 18 με 23 ετών. Την ίδια μέρα 13 έχασαν τη ζωή τους σε μια επίθεση σε ένα χριστιανικό χωριό. Αυτά τα ονόματα έρχονται να προσταθούν στις 35.000 που ήταν άμεσα θύματα του τζιχαντισμού την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα του Μπόκο Χαράμ. Για τρεις λόγους. Πρώτον, είναι αυτές οι σειράξεις που βρίθουν εκεί και ευημερούν και δεν γίνεται τίποτα για να σταματήσουν γιατί κανείς δεν βλέπει δεν θέλει να δει ότι πίσω από τις φιλετικές σειράξεις ε, ε, έχουμε ένα πεδίο μάχης του Ισλαμισμού που παγκοσμίω προσπαθεί να βάλει σφήνες, ε, να σκοτώνει και να διαιρεί. Το δεύτερο λόγο είναι η απάθεια, η παθητικότητα και καμιά φορά η συνενοχή τη κυβέρνηση σε κάποιων σωμάτων ασφαλεία που δεν επεμβαίνουν. Και θα πρέπει να φέρουμε την κυβέρνηση απέναντι στι ευθύνε τη, γιατί έχει τη δυνατότητα να επέμβει και θα πρέπει να εγγυάται ε, τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και ο τρίτο λόγο είναι η δική μα εύθραυση στάση. Γιατί ε, από την Αφρική αποσύρονται οι ΗΠΑ, η ίδια Ευρώπη είναι ξεπερασμένη από τι εξελίξει και ενώ που αφήνουμε έρχονται να το καλύψουν άλλε δυνάμεις. Η Κίνα φυσικά, αλλά η Τουρκία, το Κατάρ, όλε αυτέ οι χώρε που έχουν συμφέρον φυσικά οικονομικό, αλλά όχι μόνο και χωρίς καμιά αμφιβολία και ιδεολογικό συμφέρον να δρούν σε μια τέτοια περιφέρεια και να την κάνουν ακόμα πιο εύθραυστη. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι συνεπής στο ραντεβού της για να εγγυηθεί ε, το σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ιδιαίτερα των χριστιανικών, που χρειάζονται την προστασία μας. Και για να υπάρχει ισορροπία στην περιοχή θα πρέπει να φέρουμε ενώπιον των ευθυνών τη την Νιγηριανή κυβέρνηση. Θα πρέπει σήμερα η Ευρώπη να δράσει στην Νιγηρία. Ευχαριστώ κύριο ε, Τσουχοντάρου, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαστε σε ναρκοθετημένο πεδίο. Φαίνεται ε, να μην υπάρχει εύκολη λύση. Εγώ είμαι γιατρός, επιγοντολόγος στην ε, Ρουμανία. Ε, είναι μια τραγωδία αυτό που συμβαίνει. Αν ε, δούμε τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στην ε, Νιγηρία δεν ήταν επαρκή. Θα υπερψηφίσω το ψήφισμα αυτό σήμερα χωρίς καμιά δυσκολία. Ε, μπορεί έτσι κάπως να στρίξουμε τα θύματα, αλλά χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα για να περιοριστεί η υποκρισία σύμφωνα με την οποία εμεί προστατεύουμε δίθεν τους Νιγηριανούς, αλλά συνεχίζουμε να πουλάμε όπλα ε, στην περιοχή. Μιλάμε για ανθρωπιστική βοήθεια. Εγώ συμμετείχα εθελοντικά σε εκστρατεία κατά του έμπολα και θα είμαι εθελοντή και για την Ιγυρία. Είναι σωστέ αυτέ οι πρωτοβουλίε, αλλά πρέπει ακόμα να γίνουν πάρα πολλά. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Σαρντώνε τώρα από την ομάδα... Η κυρία Σαρντώνε, συγγνώμη, ε, ταυτότητα και δημοκρατία. Κάθε μέρα χάνουν τη ζωή του 12 χριστιανοί, ενώ είναι στην εκκλησία, ενώ πάνε στη δουλειά του, στο σχολείο, στου παιδικού σταθμού, ενώ ε, ε, προσεύχονται. Οι γυναίκες βιάζονται, τα παιδιά βασανίζονται. Καθημερινότητα είναι στην Ιγυρία η δολοφονία χριστιανών. 13.000 εκκλησίες έχουν εγκαταλειφθεί ή καταστραφεί. 1,5 εκατομμύριο είναι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Ε, ε, στην Ιγυρία οι χριστιανοί κυρίως στα βόρεια της χώρας ε, ε, διώκονται, δέχονται επιθέσεις, στερούνται δικαιωμάτων, ε, ακόμα και σε καθημερινές ανάγκες. Σε όλα αυτά η Ευρώπη σιωπά. Κανένα μήνυμα, καμία υπόσχεση προστασίας, καμία σοβαρή παρέμβαση. Όπως έλεγε η Οριάννα Φαλάτσι, Ξύπνα Δύση. Οι χριστιανοί που διώκονται ζητούν βοήθεια. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φιντάντζα τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 11 χριστιανοί... Ε, ε, εκτελέστηκαν ε, την ημέρα των Χριστουγέννων, μια ε, αιματηρά Χριστούγεννα στην Ιγυρία. Μπόκο Χαρά, μαζί με την Ίσβα, είναι το, το ένοπλο χέρι του Ισλαμικού κράτους. Παρά τις υποσχέσεις του νέου Προέδρου δεν έχει υπάρξει καμιά αλλαγή. Οι χριστιανοί διώκονται πουθενά. Στα σχολεία στο 2018 είχαμε 200.000 εσωτερικά εκτοπισμένους λόγω της Ισλαμικής Βία Διώκονται οι χριστιανοί λόγω της θρησκείας τους, λόγω της πίστης τους. Και ωστόσο, στο ψήφισμα που θα ψηφίσουμε σήμερα, η λέξη χριστιανή εξαφανίζεται. Και χθε τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι τροπολογίε για του χριστιανού που διώκονται απορρίφθηκαν από αυτήν την ε, ολομέλεια. Εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, πρέπει κυρίω να αναγνωρίσουμε τα θύματα και τι σφαγέ και να καθορίσουμε την ε, πολιτική συνεργασία μα με την Ιγυρία με σοβαρές προσπάθειες ε, καταπολέμησης της Ισλαμικής τρομοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σόκολ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι χριστιανοί είναι η ομάδα που διώκεται περισσότερο στον κόσμο σήμερα. Και αυτό δεν είναι προσωπική μου εντύπωση, αλλά είναι γεγονός. Λίγα νούμερα. Το 2018 πάνω από 4.000 ε, χριστιανοί έχασαν τη ζωή τους ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. 300, 250.000 ε, διώκονται λόγω και μόνο της πίστης τους. Ε, πραγματικά πρέπει να ε, σκεφτούμε τι σημαίνουν αυτά τα νούμερα. Η αντίληψή μας στη Δύση, τουλάχιστον στα μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είναι η αντίθετη. Στην Ιγυρία έχουμε μία ε, κλιμάκωση αυτής της κατάστασης. Ε, πέρυσι 130 χριστιανοί έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 6.000 τα τελευταία 5 χρόνια από το 2015. Χιλιάδες χριστιανοί δολοφονήθηκαν στην Ιγυρία μόνο και μόνο λόγω της πίστης τους. Πρέπει ειλικρινά να πούμε πως δεν πρόκειται για σύγκρουση μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά ότι πρόκειται για διωγμούς κατά των χριστιανών και που παρομοιάζουν σε, ε, γενοκτονία. Οι γυναίκες βιάζονται, διώχνονται, τα παιδιά βασανίζονται, είναι διωγμή αυτή. Η Νιγηρία είναι μια χώρα όπου 50% ήταν ε, χριστιανοί, 80 εκατομμύρια χριστιανοί ζουν εκεί και φανταστείτε τι αισθάνονται στη χώρα στις, στις άλλες χώρες όπου είναι μειονότητα. Πρέπει λοιπόν σαφώς να πάρουμε θέση κατά των διωγμών των χριστιανών στην Ιγυρία και σε άλλες χώρες και να μιλήσουμε εδώ ε, για τους διωγμούς κατά των χριστιανών σε ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει αυτό να τα πούμε ξεκάθαρα διότι πρόκειται για πρόβλημα το οποίο πρέπει να καταπολεμήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Βαλιέρη για το ID. Η χριστιανική κοινότητα στην ε, Νιγερία υφίσταται γενοκτονία. Τους τελευταίους μήνες έχουν δολοφονηθεί πάνω από χίλιοι χριστιανοί, αλλά δεν συλλαμβάνονται ποτέ οι ένοχοι. Τα δε Χριστούγεννα είχαμε μια τεράστια σφαγή 11 χριστιανών που ανέβηκε και στο διαδίκτυο. Λίγες μέρες ε, μετά τέσσερις ε, κινηματογραφιστές απήχθησαν σε μια περιοχή όπου επικρατεί η Σαρία. Συνολικά υπάρχουν 30.000 θύματα άμαχοι και δεκάδες χιλιάδες ακόμα που έχουν εξαφανιστεί. Έχουμε λοιπόν 1.300.000 άτομα τα οποία επίσης έχουν φύγει από τις ε, αιστείες τους. Δεν μπορεί λοιπόν να μην κάνουμε τίποτα. Οι Ισλαμιστές ε, φονταμεταλιστές δεν αποτελούν κίνδυνο μόνο για την Ιγυρία και τους ε, Νιγηριανούς χριστιανούς αλλά και για την Ευρώπη και για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ράισεν από το Κυρία Πρόεδρε, χιλιάδες ε, νεκροί, ε, εκατομμύρια πρόσφυγες, ε, καμένες εκκλησίες και σπίτια είναι ο θλιβερός απολογισμός των τελευταίων εβδομάδων στην Νιγηρία. Ο ιστορικός διαχωρισμός του Ισλαμικού Βορρά και του Χριστιανικού Νότου εντείνεται με την διάδοση του Μπόκο Χαράμ και του Ισλαμικού κράτους. εντείνεται επίσης, εντείνονται οι συγκρούσεις ε, μεταξύ των, ε, της φυλής ε, Φουλάνη και των χριστιανών. Και υπάρχει και θρησκευτική διάσταση. Βεβαίως η πραγματικότητα είναι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι διώκονται από τα σπίτια τους και καταστρέφεται η ζωή τους. Και βεβαίως η απάντηση της ε, κυβέρνησης είναι ελιπέστατη. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα κάνει συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει τη βία στην Ιγυρία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μπενχουμέα, Μπενχουμέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, η συζήτηση αυτή που γίνεται σήμερα εδώ ανταποκρίνονται σε κάποιες τραγωδίες, κάποια δραματικά που ε, ζήσαν στην Νιγηρία. Νιγηρία ανήμερα τα Χριστούγεννα δολοφόνησαν πιστούς χριστιανούς απλώς και μόνο επειδή ασκούσαν ε, τη λατρεία της θρησκείας τους. Γι' αυτό το συζητάμε, γιατί υπήρξε αυτή η τρομακτική επίθεση κατά των χριστιανών στην Ιγυρία. Δεν είναι μονομένη όμως αυτή η επίθεση, είναι συστηματικές επιθέσεις όλο αυτό τον καιρό. Απέναντι στην απάθεια της ε, ε, ε κυβέρνηση και των αρχών. Να σας δώσω κάποια στοιχεία από το 2015. Έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 6.000 χριστιανοί ε, από τζιχαντιστές τρομοκράτες στην Ιγυρία. Φυσικά η Ιγυρία ζει και άλλα δράματα και τον Μπόκο Χαράμ δολοφονεί και μουσουλμάνους και Εβραίους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως πρόκειται για μια τραγωδία που αφορά τους διωγμούς των χριστιανών παγκοσμίω. Και δεν θα πρέπει να χάσουμε την εστίαση μας. Λυπάμαι που κατά την διαπραγμάτευση για το ψήφισμα αυτό είχαν κάποιοι μεγαλύτερη αγωνία από το να βγει όρος από το ψήφισμα παρά να συζητήσουμε τι έγινε την περασμένη Ολομέλεια συζητήσαμε για τις επιθέσεις στην Μπουρκίνα Φάσο και σήμερα στην Ιγυρία. Φυσικά στέλνω τα συλληπιτήριά μου σε όλες τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων. Θα ήθελα τα τελευταία αυτά δευτερόλεπτα που έχω να σας θυμίσω μερικά αριθμητικά στοιχεία για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για διωγμούς χριστιανών στον κόσμο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να, παραμείνει ε, αδρανείς. Πρέπει να δράσουμε, να αντιδράσουμε. Εδώ πρόκειται για τις αξίες της δύση, τις ιουδεοχριστιανικές θρησκείες, επί των οποίων έχει οικοδομηθεί η Ευρώπη. Το 2020 έχουμε 4.305 χριστιανούς που δολοφονήθηκαν σύμφωνα με την έκθεση της Open Doors. Δεν μπορούμε να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Θα πρέπει να υπερασπίσουμε τις αρχές και τις αξίες αυτές, τι Ιουδεοχριστιανικές, τι οποίε εδράζεται και οικοδομείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκατσίνη από την ομάδα των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. μισό λεπτό. Ε, μπλε κάρτα προς την κυρία Μπεν Χουμέα. Δέχεστε την ερώτηση από τον κύριο Τόμας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η συνάδελφος παρέθεσε συγκλονιστικά αριθμητικά στοιχεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και πρέπει να το συζητήσουμε γιατί διώκονται πραγματικά οι χριστιανοί και οι χριστιανές και είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία ε, πόσο μάλλον όταν έγιναν τα Χριστούγεννα αυτά τα δραματικά γεγονότα. Θα πρέπει να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει όμως η αποφασιστική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστατεύσει τους χριστιανούς παγκοσμίω. Ευχαριστώ απάντηση κυρία Μπενχουμέα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μα, ειλικρινά το είπαν και κάποιοι συνάδελφοι προηγουμένως δεν μπορούμε να γυρνάμε την πλάτη στην πραγματικότητα της Αφρικής. Θα πρέπει να απαιτήσουμε από τις αρχές της χώρας να υπερασπίζουν, να προστατεύουν τους χριστιανούς. Τώρα κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια και οι ένοπλες δυνάμεις και ε, τα σώματα ασφαλείας δεν αντιδρούν. Εμείς θα πρέπει να απαιτήσουμε μέτρα. Ευχαριστώ, Προκατσίνη. Ε, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε θα υπερψηφίσουμε για να καταδικάσουμε τις διώξεις των χριστιανών στην ε, Νιγηρία. Αλλά δεν μπορούμε να αγνοούμε το πώς ε, έχει φύγει από την διατύπωση του ψηφίσματος η λέξη χριστιανή για τους ανθρώπους που κάθε μέρα ταπεινώνονται, βασανίζονται και δολοφονούνται στην Νιγηρία. Ιδίως ε, τα Χριστούγεννα ή τις γιορτές όπως ε, τις λέμε υποκριτικά. Ειδικά η ΜΚΟ Open Doors έχει σημειώσει πως ε, οι επιθέσεις ε, κατά χριστιανών αφορούν 220 εκατομμύρια άτομα και αφορούν επίσης πάρα πολύ περισσότερο αρκετές δολοφονίες. Και σε αυτήν την θλιβερή κατάταξη η Νιγηρία δεν βρίσκεται καν στις 10 πρώτες χώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Χέρμαν από το ΕΛΚ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στην Νιγηρία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από το 2015 το Μποκο και άλλες ε, τρομοκρατικές ομάδες έχουν σκοτώσει πάνω από 6.000 ε, χριστιανούς. Αντιμετωπίζουμε τεράστια απειλή και πρέπει ο πρόεδρος να καταδικάσει τις ε, απειλές αυτές και να δράσει για να αποκλιμακωθεί η ένταση. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει προστασία των πολιτών και ασφάλεια και να απευθύνουμε έκκληση για δικαιοσύνη αλλά αυτό πρέπει να γίνει <clears throat> στο πλαίσιο της δικαιοσύνης. Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται αφαίρετα. Ιδιαίτερος τα παιδιά, κανείς δεν μπορεί να κρατείται υπό τέτοιε εξευτελιστικές συνθήκες, όπως μας λέει η Human Rights Watch. Αυτό παραβιάζει το Σύνταγμα της Νιγηρίας και την ε, διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεν αρκεί μόνο ο στρατός. Πρέπει να δούμε τις αιτίε της ριζοσπαστικοποίησης, να υπάρξει ένας διάλογος, ελευθερία έκφρασης και ανεξιθρησκεία και να μειώσουμε τη φτώχεια. Αυτό είναι επίσης αποτέλεσμα της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης. Ε, πάνω από το μισό πληθυσμό, ε, πάνω από το μισό πληθυσμό ε, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και υπάρχουν πάρα πολλές επιθέσεις ακόμα και στην ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει λοιπόν να καταδικάσουμε τους διωγμούς των ανθρώπων που έχουν πάει και να βοηθήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε 7 συναδέλφους για το ΚΕΤΣΙΑΙ, θα τους ακούσουμε όλους. Πρώτος είναι ο Χέισελ για τους σοσιαλιστές. Είναι τεράστια χώρα η Νιγηρία. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ε, στην Αφρική και έχει πολύ μεγάλο δυναμικό όσον αφορά τις πρώτες ύλε. Θα μπορούσε να αποτελεί ηγέτη στην Αφρικανική Ήπειρο. Θα έπρεπε να έχουμε καλές σχέσεις μαζί τους. Ε, στην πράξη όμως ε, δυστυχώς ε, είναι ε, έρμεο φοβερών ε, φρικτών τρομοκρατικών επιθέσεων. Βέβαια, στόχος δεν είναι μόνο οι χριστιανοί, αλλά και οι μουσουλμάνοι. Και θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για κοινωνικο-οικονομική σύγκρουση ανάμεσα στους γεωργούς και εκείνους που προσπαθούν και τους κτηνοτρόφους. Ε, θα έπρεπε να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε διάλογο με την κυβέρνηση της Νιγηρίας και να επιμείνουμε για την προστασία των ελευθεριών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντάλι είναι η επόμενη. Ντέιλι, με συγχωρείτε, είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Προφανώ η βία δεν είναι νέο φαινόμενο. Η βία σε καμία περιοχή τη Νιγηρία Έχουμε στην Ιρλανδία ετούντε άσυλο που θεωρούνται ε, οικονομικοί πρόσφυγες, λέει, ε, και δεν τους προσφέρεται το άσυλο. Μα δείτε τι συμβαίνει. Δέκα χρόνια ε, ταλαιπωρούνται με τον Μποκο Χαράμ. Έχουν εκτοπιστεί χιλιάδες άνθρωποι. Δύο εκατομμύρια λένε. Δεκάδες χιλιάδες είναι αγνοούμενοι και οι περισσότεροι είναι παιδιά. Πώς γίνεται 50% του πληθυσμού να ζει σε ακραία φτώχεια σε μια χώρα που είναι η 12 μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου. Πρέπει να δούμε το ρόλο των ευρωπαϊκών ομίλων εκεί, όπως η Total, η Shell. Από, ε, ε, υπάρχουν ε, συμφωνίες με την Νιγηριανή Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου που δεν πληρώνει φόρους και δεν φροντίζει καθόλου το περιβάλλον. Πράγμα που καταλήγει στο να προσπαθούν ορισμένοι να υπερασπιστούν τις κοινότητές τους και τις περιοχές τους. Ναι, ε, ε, και ενώ οι Ρακινοί θρυνούν ε, τον Σολεϊμάνη που τους, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει γιατί αυτός τους έσωσε από τέτοιες καταστάσεις. Ευχαριστώ. Λέναρτζιτς. Ο κύριος Κέλλη, με συγχωρείτε. <coughs> Η Νιγηρία ταλανίζεται από την τρομοκρατική ομάδα Boko Haram εδώ και μια δεκαετία και είναι το βασικό αίτιο η οργάνωση αυτή για τα φρικτά που συμβαίνουν εκεί. Συμφωνώ, όπως είπαν και άλλοι, ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τα 100 κορίτσια τα οποία κρατούνται όμοιροι από ε, την Boko Haram. Ε, ιδιαίτερα γιατί η οι αρχές εκεί προσπαθούν ε, να καταπολεμήσουν τον Μπόκο Χαράμ. Ενώ είναι πλούσια σε πόρους, η Νιγηρία είναι μια από τις χώρες στην Αφρική. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε, ειδικά όσον αφορά τους πρόσφυγες, όπως ανέφερε η Κλέρ Ντέιλι, επίσης το χειρισμό και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την περάσπιση των χριστιανών στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Μπέργκερ, συγγνώμη. Έχετε το λόγο. Ναι. Ε, η κατάσταση στην Ιγερία, που είναι η μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής, με συγχωρείτε, μπορείτε να σηκωθείτε όρθια παρακαλώ. <coughs> Ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση στη Νιγηρία, που είναι η μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής, μας ανησυχεί όλους απέναντι στην επιδείνωση αυτής της κατάστασης σε θέματα ασφάλειας και γενικευμένης βίας που οδηγεί σε μαζικές μετακινήσεις των πληθυσμών και μια επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης. Το 2014 το Μπούκο Χαράμα πήγαγε νεαρές κοπέλες και γυναίκες και τις υπέβαλε σε σεξουαλική βία. Η βία έχει αυξηθεί και άλλο απέναντι στις γυναίκες και έχει και τις γενικές συνοριακών περιοχών όπως τα σύνορα με το Καμερούν. Πρόσφατα ε, μοναχές απέκτησαν και φυλακίστηκαν. Καταδικάζουμε αυτές τις θρησκευτικέ και εθνοτικέ ε, επιθέσεις. Υπολογίζεται ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι επηρεάζονται από την αδυναμία των ανθρωπιστικών οργανώσεων να έχουν πρόσβαση σε μεγάλα κομμάτια της χώρας. Δύσκολη πρόσβαση λοιπόν, γι' αυτό 70% των παιδιών πάσχουν ε, από ασυτεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανασκουμποηθεί, να βρει νέου τρόπου να συνεργαστεί με την Ιγυριανή κυβέρνηση, ώστε να μπορέσει να διοχετευτεί η ανθρωπιστική βοήθεια και κυρίω να τεθεί τέλο αυτή τη βία κατά των γυναικών και των θρησκευτικών κοινοτήτων. Τα όσα συνέβησαν τα Χριστούγεννα δεν πρέπει να επαναληφθούν ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δεσμευθεί με την κυβέρνηση του Ισνιγηρία ώστε να προωθήσει τα και τις ανθρωπιστικές αρχές, να ενισχύσει ε, το διάλογο με τις αρχές ώστε να σταματήσει αυτή η ε, επίθεση κατά των αμάχων και να σταματήσει και η σεξουαλική εκμετάλλευση που σοβεί εδώ και τόσα χρόνια. Αυτά ευχαριστώ. Please keep the minute. Παρακαλώ, λέει η Πρόεδρος, να μείνετε στο ένα λεπτό που σας αντιστοιχεί, γιατί αλλιώ δεν θα έχουμε χρόνο για τους υπόλοιπους ομιλητές. Ο κύριος Πόσπισιλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συμφωνούμε για τα προβλήματα που ε, αντιμετωπίζει αυτή η δυστυχισμένη χώρα. Είναι τεράστια η διωγμή και η βία κατά των χριστιανών. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να το τονίζουμε και στο μέλλον. Κάτι όμως το οποίο δεν δώσαμε έμφαση είναι ότι η Νιγηριανή ε, κυβέρνηση εμφανίζει μια χαλαρότητα απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις και όταν δεν είναι συνένοχοι, όταν δεν συμμετέχουν ε, ε, μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας θα πρέπει να πιέσουμε πολύ περισσότερο την κυβέρνηση της Νιγηρίας για να ε, καταπολεμεί πραγματικά ε, τους τρομοκράτες και όχι τους συνηθισμένους κανονικούς Νιγηριανούς πολίτες. Πρέπει ναι, είναι πιο αποτελεσματική η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εμείς να τους δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια και ό,τι άλλο χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνω η διαδικασία. Κατστιάη με τον συνάδελφο Γόλος από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταδικάζω τους διωγμούς των χριστιανών, των μουσουλμάνων, των Κούρδων, όπου και αν ζουν. Η σημερινή κατάσταση στην Νιγηρία είναι ένα μάθημα για την υπεραλιστική Ευρώπη. Είναι άμεση ε, απόρρια ε, της Βρετανικής υπεραλιστικής τάσης και ανάμιξης άνοιξαν τον δρόμο για τα Ισλαμικά στο βορρά με τις εκλογές. Και, ε, η Νιγηρία έχει ένα λαμπρό μέλλον, αλλά αυτό έχει καταστραφεί. Είδαμε τι έγινε με το χριστιανικό χωριό Μαλούλα πριν από δύο χρόνια ε, στη Συρία. Οι τζιχαδιστές, τους οποίους όπλησε η Δύση μπήκαν στη χώρα μέσω των τουρκικών συνόρων. Η ασυνέπειά μας είναι τρομακτική. Κοιτάξτε τι παθαίνουν οι Παλαιστίνοι ε, από το Ισραήλ, από τους Ελληνούς, ε, οι μουσουλμάνοι στην Ινδία, ε, στη Γενεμένη, τι γίνεται, έχετε δει, ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και τώρα το λόγο έχει ο Επίτροπος, ο κύριος Λέναρσιτς, για να κλείσει η συζήτηση και να απαντήσει και να σχολιάσει τις ομιλίες που ακούσαμε. Uh, Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, από πέρυσι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρωπιστική κατάσταση στην Ιγυρία έχει επιδεινωθεί σημαντικά σε μεγάλο βαθμό. Το περασμένο χρόνο έχουν γίνει τρομοκρατικές επιθέσεις και οι συγκρούσεις ε, έχουν στοιχήσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας ε, στις οικογένειες ε, των θυμάτων και την αλληλεγγύη μας με το λαό τις Νιγηρίες και κυρίως με τις κοινότητες που τόσο πολύ έχουν επηρεαστεί από την ανάδυση παρακρατικών ενόπλων οργανώσεων, κυρίως στα βορειοδυτικά της χώρας. Ο Μπόκο Χαράμ έχει σκοτώσει 36.000 και βάλε κόσμο στην Ιγυρία μόνο από το 2009. Επιπλέον ε, πρόκληση είναι η αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση. Πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμος φαίνεται να είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Πάνω από 7 εκατομμύρια χρειάζονται ανθρωπιστική ε, βοήθεια. Και πάνω από ένα εκατομμύριο θεωρείται ότι ε, είναι εκτός ανθρωπιστικής πρόσβασης. Ο ΙΕ παρακολουθεί την κατάσταση πάρα πολύ προσεκτικά. Έχουμε ε, ε, σχεδιάσει μία ε, πολύπλευρη προσέγγιση που στοχεύει στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην κοινωνική και ανθρωπιστική ανάπτυξη σε κοινοτικό επίπεδο. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ιγυρία να ανταποκριθεί στα προβλήματα ασφαλής στην κρίση ασφάλειας, ανάπτυξης και ανθρωπιστικής ε, κατάστασης, ιδιαίτερα στα βόρειο-δυτικά, το Δέλτα του Νίγηρα και αλλού ε, και ε, βεβαίως σε όλες αυτές τις υποθέσεις να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα αντιμετωπίζει τα αίτια του κακού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους βασικούς δωρητές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ιγυρία. Δίνουμε ε, κάλυψη των άμεσων ανάγκων, ε, αναγκών των πιο ευάλωτων ιστορικά εκτοπισμένων ανθρώπων και κοινοτήτων. Από το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χορηγήσει σχεδόν 245 εκατομμύρια ε, ευρώ για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στην Ιγυρία και το 2019 προσφέραμε 20 εκατομμύρια σε ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει, στοχεύει να χτίσει ε, μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και αντοχή ε, και στήριξη στις βασικές υπηρεσίες και την αποκατάσταση του τρόπου διαβίωσης, επιβίωσης, ώστε θέλουμε να... Πάνω από μισό δις έχουμε προσφέρει σε αυτή την προσπάθεια μέχρι το 2019. Από το 2014 επίσης γίνεται προσπάθεια κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του βίου εξτρεμισμού. Προσπαθούμε να στηρίξουμε ε, την ε, πολιτική προστασία, την ε, επανένταξη και την συμφιλίωση και προσπαθούμε να δώσουμε βοήθεια στο σύστημα ποινική, στο ποινικό δικαστικό κομμάτι στην Νιγηρία. Την επόμενη εβδομάδα θα μεταβώ στην Νιγηρία και στη βορειοδυτική πλευρά της ε, βορειοανατολική με συγχωρείτε πλευρά τη, ώστε να δώσω μήνυμα στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Ανησυχούμε πολύ λόγω τη συρρήκνωση ε, τη ε, δυνατότητα πρόσβαση ανθρωπιστική βοήθεια στο βορειοανατολικό τμήμα τη χώρα η καταπολέμηση της βίας είναι η πρώτη προτεραιότητα για μένα. Επιπλέον, η επόμενη σύνοδος ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νιγηρίας θα γίνει το... τον ε, προσεχώς και αυτό εκεί θα τονίσουμε όλα αυτά τα θέματα φυσικά. Πρόεδρος, Μάλιστα έλαβα 7 ε, προτάσεις ψηφίσματος, ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα, θα γίνει σήμερα στις 12 και στις 12 θα συνεχίσουμε και τη σύνοδο. Διακοπή μέχρι τις 12. Thank you very much, colleagues. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Sorry for the little delay. Συγγνώμη για τη μικρή αυτή καθυστέρηση. Αλλά είχαμε την υποχρέωση να περιμένουμε να τελειώσει η διάσκεψη των Προέδρων. Ερχόμαστε όμως τώρα στις ψηφοφορίες και αν είστε όλοι έτοιμοι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ψηφοφορία για τον Μπουρούντι. Διαδικαστικό ποιος, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Πρόεδρε, 196. Άρθρο 196. Την περασμένη Δευτέρα ο πρόεδρος είπε στους υπαλλήλους της Ολομέλειας να αφαιρέσουν τις μικρές σημεούλες που είχαν οι συνάδελφοί μου στα έδρανά τους. Θεωρώ ότι αυτή η απόφαση είναι αντίθετη στους κανόνες. Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου αποφάσισε να επιβάλλει απαγόρευση για τα μεγάλα, στις μεγάλες αφήσεις για να αποφύγει διαμαρτυρίες που γίνονταν με αφήσεις εντός της ε, Ολομέλειας και να επιβληθεί τάξη. Αλλά ε, για μας είναι αφίβολο, αφίβολη σημασία και ε, κανονικότητα στο ότι απαγορεύει τα μικρά σημαίακια που είχαμε των κρατών μας. Εμείς με περηφάνεια θα συνεχίσουμε αναφέρνουμε παρά την απαγόρευση αυτής της σημεούλης στην αίθουσα της Ολομέλειας και στα έδρανά μας. Μάλιστα, η Πρόεδρος. Αναφερθήκατε στο άρθρο 10 του κανονισμού. Θα το πω στα γερμανικά γιατί γνωρίζω καλύτερα και διαβάζω εδώ. Ε, τα μέλη δεν θα πρέπει να ενοχλούν τις εργασίες στην Ολομέλεια ε, και να ε, έχουν ανάρμαστη συμπεριφορά, δεν θα πρέπει να σηκώνουν πανό και να εκδηλώνονται. Ως πανό θεώρησε και τη σημαίες ο Πρόεδρος. Παρακαλώ να σεβαστείτε αυτή την απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου όσο είναι ακόμη ενισχύ. E Κοιτάξτε, δεν είναι τίποτα παλιόχαρτα, ούτε είναι σύμβολα τα οποία διαταράσσουν την τάξη στην Ολομέλεια. Οπότε δεν απαγορεύει τέτοιου είδου. Ε, Τι σημαίε των κρατών μα δεν απαγορεύονται στην Ολομέλεια. Αγαπητέ κύριε Τζάνη, δεν θα γίνει συζήτηση τώρα για τα θέματα αποφάσεων του Προέδρου. Αν θέλετε να την προσβάλλετε αυτή την απόφαση, μπορείτε να το κάνετε και θα αποφανθούν τα αρμόδια όργανα. Αλλά όσο ισχύει, σας παρακαλώ να τη σέβεστε αυτή την απόφαση. Another point of order. Άλλο διαδικαστικό. Άλλο διαδικαστικό. Ε, θα το κάνω μόνο εφόσον όλοι σεβαστείτε την εντολή του Προέδρου. Αλλιώς δεν συνεχίζουμε τη συζήτηση. Συγγνώμη συνάδελφοι, εσείς δεν τον αφήνετε να μιλήσει γιατί δεν ε, ε, ακολουθείτε τις εντολές του Προέδρου. Ε, για να τον αφήσετε να μιλήσει, για να του δώσω το λόγο πρέπει να γίνει αυτό που είπα. Υπάρχει κι άλλο διαδικαστικό. Mrs. I'm sorry. Από την κυρία Στρόγκαριτς. Αγαπητοί συνάδελφοι, διαβάστε παρακαλώ τον κανονισμό του Κοινοβουλίου προσεκτικά. Απαγορεύεται και το νεροπότηρο ε, επάνω στο έδρανο, μπορείτε να μαζέψετε τα σημαίακια και να τα βάλετε κάτω από τα έδρανα. Πάλι κοντά σας θα τα έχετε. Mr. Corbett. Madam Ο κύριος Κόρμπετ. Κυρία Πρόεδρε. Ο κανονισμός λέει ότι τα μέλη δεν θα πρέπει να σηκώνουν πανό. Μπάνερ. Τώρα η λάβαρο τι είναι το μπάνερ. Ε? Είναι θέμα ορισμού. Μόλις κοίταξα τον ορισμό στα αγγλικά της λέξης μπάνερ στο Wikipedia που λέει ε, ότι μπορεί να είναι σημαία ή άλλο ύφασμα που φέρει σύνθημα, ε, μήνυμα, ε, σλόγγαν ή κάτι άλλο. Αγαπητέ συνάδελφε, η πρόεδρος διακόπτη. Ο κύριος Κόρμπετ λέει παρακαλώ να αποσυρθούν οι σημαίες. Δεν λέω αν είναι σοφή αυτή η κατι αλλο αγαπητες συναδελφε η προεδρος αλλά έτσι έχει απόφαση η πρόεδρος. Κοιτάξτε, εγώ δεν βιάζομαι. Έχω πάρα πολύ χρόνο. Ε, λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Ε, όχι τώρα τι εστί μπάνερ και τι δεν εστί ε, σημαία λάβαρο, αλλά εάν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου παίρνει μια απόφαση, τότε η απόφαση αυτή θα πρέπει να τηρείται. Όσο παραμένει ενισχύ και δεν έχει αποσυρθεί και δεν έχει κυρωθεί, τόσο εύκολο και απλό είναι. So, I, yes, keep calm, keep calm. Ηρεμία. We have obviously... Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι πέμπτη και θέλουμε όλοι να φύγουμε και το κατανοώ. Τώρα αρχίζουν ψηφοφορίες. And we will start with... Μπουρούντι πρώτο. Παράγραφος 18. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Προχωρούμε στην Ιγυρία. Μετά την παράγραφο 18, η τροπολογία 1, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 21, τροπολογία 2, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, τελική σκέψη F δύο τμήματα. Το αρχικό κείμενο. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Αρχίζει η ψηφοφορία τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ά, με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος ψηφιπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Προχωρούμε. Βενεζουέλα. Ο κύριος Λόπες Χίλ έχει ζητήσει το λόγο. και ελπίζω να είναι ή διαδικαστικό ή προφορική τροπολογία. Είναι, είναι. Διαδικαστικότατο. Ήθελα να καταγγείλω τα σοβαρότατα γεγονότα που έγιναν το τελευταίο 24ωρο στο Καράκας. Οι παραστρατιωτικές οργανώσεις του καθεστώτος επιτέθηκαν με πέτρες και με ρόπαλα και με ξύλα στα οχήματα όπου ήταν ο πρόεδρος. Η πρόεδρος διακόπτη, δεν ξαναρχίζει η συζήτηση. Έχετε προφορική τροπολογία ή διαδικαστικό τροπολογία θέλω να υποβάλω. Προφορική τροπολογία. Καλώς. Ποια είναι η τροπολογία. Θέλω να ζητήσω ρητά να ζητήσουμε να υπάρχει εγγύηση, ε, πέρα από τα όσα λέει το ψήφισμα, για τη ζωή των νόμιμα εκλεγμένων ε, βουλευτών στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας. Και πού θέλετε να μπει αυτό, σε ποιο σημείο του ψηφίσματος. Τι λέξεις θέλετε συγκεκριμένα να προσθέσετε, διατύπωση. Δεν είναι αυτό ε, προφορική τροπολογία. Προχωρούμε. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε την παράγραφο 7, το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον, υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον. Ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Ψηφιπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση, η οποία αρχίζει τώρα. The vote is closed. Εγκρίνεται. Προχωρούμε. Εν εξέλιξη ακροάση σύμφωνα με το άρθρο 7, Πολωνία και Ουγγαρία. Παράγραφος 2 του αρχικού κειμένου με ονομαστική κλίση έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Η τροπολογία 2 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και το αρχικό κείμενο καταπίπτει. Μετά την παράγραφο 5 έχουμε η τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική αναφορά 12 έχουμε την τροπολογία 1. Ψήφιπε Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος, ε, όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται.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 το θέμα της βιολογικής ποικιλομορφίας και ψηφίζουμε πριν από την παραγραφό 1, τροπολογία 8, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ήταν ξεκαθαρό, οπότε θα κάνουμε ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αν δεν σηκώνετε τα χέρια σας δεν μπορώ να δω. Παράγραφος 4. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Η πλειοψηφία ήταν υπέρ νομίζω. Α, να ελέγξουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, Πέρας της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα το ψηφίσαμε ήδη. Έχουμε μετά την 16, τροπολογία 16. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ήθελα αυτό να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Έγκρινεται. Τροπολογία 22, ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 23 ονομαστική κλίση. Vote is closed. Πέρασε. Έκρινεται. Τροπολογία 11 μετά από την παράγραφο 22. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 ονομαστική κλίση πέρας εγκρίνεται τροπολογία 2 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19. Ε, Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 35. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ ναι, όχι, ήταν ξεκάθαρο. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Όχι, ήταν πραγματικά ξεκάθαρο. Από εδώ που είμαι εγώ φαινότανε, ναι. Υπέρ. Ε, είμαστε στο τρίτο τμήμα. Υπέρ ποιοι είναι, κατά, αποχές. Το τρίτο τμήμα να ελέγξουμε. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, έχει αρχίσει η ψηφοφορία για το τρίτο τμήμα. Παρακαλώ να ξαναρχίσουμε γιατί ε, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, κάνουμε ε, έλεγχο ηλεκτρονικό για το δεύτερο τμήμα και μετά για το τρίτο τμήμα. Για το δεύτερο τμήμα λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Για το δεύτερο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Και παρακαλώ την επόμενη φορά να σηκώνετε τα χέρια σας για να μπορώ να δω ξεκάθαρα τι συμβαίνει. Τρίτο τμήμα άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφο 40. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Υπέρ του πρώτου. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλιστα. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 μετά την παράγραφο 43. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφο 48. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Ε, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 56 Κοιτάξτε, εάν δεν σηκώνετε τα χέρια σας εδώ στα δεξιά, είναι πολύ δύσκολο, οπότε θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ναι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Είναι η τροπολογία 4. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 56 αρχικό κείμενο πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική κλίση. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται. Τροπολογία 20 είμαστε και ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην έκθεση ΓΙΑΡ, παράγραφος 4, τροπολογια ΔΕ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12, αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19, παράγραφος 1, άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εκρίνεται. Αρχικό κείμενο καταπίπτει. Μετά την παράγραφο 19 τροπολογία 2 άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 σε δύο μέρη, μέρος πρώτο με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται μέρος δεύτερο με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20. Αρχικό κείμενο σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 21, αρχικό κείμενο σε τρία μέρη. Μέρος πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και μέρος τρίτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 25, αρχικό κείμενο σε δύο μέρη, μέρος πρώτο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, μέρος δεύτερο με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 παραγραφός μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 41 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές να το ξαναδούμε υπέρ παρακαλώ παράγραφος 41 κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφος 43, αρχικό κείμενο σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 47 αρχικό κείμενο σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μέρος δεύτερο α, με συγχωρείτε εγκρίνεται δεύτερο μέρος με ονομαστική ψηφοφορία Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το δούμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 5. Πέρασε. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας R αρχικό κείμενο, μέρος πρώτο υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Μετά από το εκτιμώντας R, τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές να το ξαναδούμε. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και μετά το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ένα ψήφισμα ακόμα θεσμικά όργανα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το ψήφισμα σύνολό του υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε μερικά λεπτά για τις επεξηγήσεις ψήφου. Συνάδελφοι, όσοι δεν θέλουν να ακούσουν τις επεξηγήσεις ψήφου, παρακαλώ, αε, διαλυθείτε ησύχως. Και όσοι θέλουν να μιλήσουν, να μπορέσουν. Ξεκινάμε με τις επεξηγήσεις ψήφου και ε, θα ακούσουμε τις επεξηγήσεις ψήφου από χτες και μετά θα περάσουμε στις σημερινές ε, ψηφοφορίες. Ξεκινάμε με την έκθεση Danjean. Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ. Μπομπάρ. Παρακαλώ, ε, οι συνάδελφοι που δεν θέλουν να ακούσουν τη συζήτηση, είτε να βγουν έξω, είτε λίγο ησυχία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο κ. Μπομπάρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα ιδεώδες ειρήνης για να μην ε, καταστρέψει την Ήπειρό μας ποτέ πια πόλεμος. Ήταν και ένα ιδεώδες συνεργασίας μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών λαών. Εγνώρισε 50 χρόνια διχασμού και το μόνιμο κίνδυνο επιστροφής του πολέμου. Ε, εν ονόματι αυτού του ιδανικού που τόσο απέχει σήμερα δυστυχώς, αμφισβητώ το σχέδιο της Ευρώπης άμυνας. Άμυνα επάνω σε κάποιον. Στη Ρωσία, μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα που θα πρέπει να είναι τέρος μας, όχι αντίπαλός μας. Άμυνα με ποιον, με τον ΝΑΤΟ, που είναι απαρχιωμένος και πολεμοχαρής οργανισμός προσιλωμένος στο άρμα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού ε, που μας βάζει να είμαστε τσιράκια ε, του ανόητου ε, του Ντόναλτ Τραμπ. Η Ευρώπη τη άμυνα είναι η Ευρώπη του πολέμου. Θα πρέπει να ξαναπάρουμε το δρόμο τη ειρήνη και να οργανώσουμε μεγάλη διάσκεψη για την ειρήνη και τη συνεργασία στην Ευρώπη για να πέσουν οι εντάσει. Θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική και περιβαλλοντική πρόκληση και να μην βάζουμε τώρα και άλλες ε, φωτιές. Αρκετές έχει ο πλανήτης. Ο συνάδελφος Χάναν. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Θα είναι η τελευταία μου παρέμβαση αυτή την αίθουσα. Ε, δεν θυμάμαι πια τον κόσμο όταν βγήκα πρώτη φορά βουλευτής. Δεν υπήρχε wifi, υπήρχαν ταξιδιωτικά πρακτορία και κανονικά εισιτήρια ταχυδρομείο, υπήρχε σε φυσική μορφή. Πολλά πράγματα άλλαξαν, αλλά κάτι το οποίο δεν έχει αλλάξει είναι η κατεύθυνση του Κοινοβουλίου και των άνθρωπων οργάνων. Παρά τα δημοψηφίσματα στη Γαλλία, Δανία, Ελλάδα και βεβαίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξακολουθεί να πηγαίνει πρόσω ολοταχώς σε όλο πιο στενή ολοκλήρωση και αυτό νομίζω τελικά κατέστησε αναπόφευκτη την αποχώρηση της Βρετανίας. Φεύγοντας λοιπόν να ευχηθώ κάθε επιτυχία στους αγαπητούς φίλους εδώ, τους φεντεραλιστές. Μπορείτε πάντα να βασίζετε στις ανοιχτέ αγορές μας, στη στρατιωτική μας στήριξη, αλλά από εδώ φεύγουμε. Καλή τύχη σας εύχομαι και καλό κουράγιο. Σας ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομιλητής για το θέμα αυτό είναι ο συνάδελφος Ζαχραντήλ. Για ένα λεπτό. Mm. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω την αίσθηση ότι μετά από το Brexit κάποια πολιτικά κόμματα, κάποιοι συνάδελφοι έγιναν πάλι φιλόδοξοι όσον αφορά μια αυτόνομη πολιτική ασφάλειας και άμυνας αγνοώντας πλήρως ε, τους ε, ατλαντικούς δεσμούς ε, που αποτελούν μια ομπρέλα που μας προστατεύει, το ΝΑΤΟ δηλαδή. Για μένα λοιπόν και εξ ονόματος της χώρας μου θα ήθελα να πω ότι εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι, πάντα θα είμαστε προσιλωμένοι στους ατλαντικούς δεσμούς άμυνας και δεν θέλουμε να εξασθενήσει το ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο θέμα η θέση του Κοινοβουλίου για την διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και πάλι ο κύριος Μπομπάρ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει από τι ελεύθερε συναλλαγέ, τη λιτότητα ε, έχει, δεν, δεν ακούει πια την ε, λαϊκή κυριαρχία όταν, από όταν επέβαλε τη συνθήκη της Λισαβόνας στο γαλλικό λαό. Το Brexit είναι προφανής, ε, προφανές παράδειγμα για το όσα συμβαίνουν. Δεν έχουν νόημα όλα αυτά παρά μόνο αν προσπαθούσαμε να φτιάξουμε πάλι το θεσμό ανάμεσα στους λαούς και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πρέπει να γνωρίσουμε πως αυτή η συνθήκη της Λισαβόνας ε, είναι περιττή και να μην κάνουμε σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα. Να μιλήσουμε για τις με τις πολιτικές ε, που οι συνέπειές τους ε, απορρίπτονται σήμερα. Θα πρέπει επίσης να μιλήσουμε για τα απολέσματα οποιασδήποτε συνέλευση ε, για το μέλλον της Ευρώπης, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν στους λαούς μέσω δημοψηφίσματος παντού. Δυστυχώς απορρίφθηκε όμως γιατί σε θέλει να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εμπορία της παρά την ολοένα και μεγαλύτερη καχυποψία των πολιτών που δεν βασίζονται σε εμά ε, που θα τους προσφέρει ακόμα μεγάλη απογοήτευση. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενο θα έπρεπε να είναι ο κύριος Μίλλερ, αλλά δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Οπότε περνάμε στην Claire Φόξ. Εγώ απήχα γιατί είμαι διευθυντής ενός Ινστιτούτου Ιδεών στο Ηνωμένο Βασίλειο που στόχο έχει τη συμμετοχή των πολιτών και να ακούγονται οι πολίτες. Αυτό είναι αυταξία. Όμως η διάσκεψη αυτή που θα διοργανώσετε ε, κυρίως ε, πρόκειται για κάτι το οποίο έχει στόχο να σώσει την φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία είναι μια αυταρχική γραφειοκρατία και έχει δημοκρατικό έλεγμα. Είναι λοιπόν κάτι το σκηνοθετημένο. Περιέχονται φράσεις εδώ λέγοντας ε, που λένε ότι πρέπει να υπάρξουν προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις για να, για να προετοιμάσουμε τους πολίτες. Δηλαδή δεν εμπιστεύεστε τους πολίτες. Και ακόμα χειρότερα απορρίψατε τροπολογίες που λένε ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτό το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Και το απορρίψατε αυτό. Δεν ναι, θα γίνει λοιπόν ουσιαστική συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια χαμένη ευκαιρία που τελικά θα καταλήξει να είναι δημόσιες σχέσεις. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, αλλά πρέπει να αφήσετε τους πολίτες να μιλάνε ελεύθερα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βρετσιόνοβα. Ε, ευχαριστώ. η συζήτηση για το μέλλον ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο σε σχέση με τον Brexit, ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Η πρόταση που ψηφίσαμε είναι πολύ παραπλανητική και στενή. Δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε μόνο σε περαιτέρω παραχωρήσεις ε, κυριαρχίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σκεφτούμε και τις ε, υφιστάμενες αρμοδιότητες της Ένωσης, να ελεγχθούν αυτές και όσες δεν είναι αναγκαίες να επανέλθουν στα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει όμως αυτό μέσα στις ε, προτάσεις. Μόνο περισσότερη ολοκλήρωση και το γνωστό σοου αυτό πανευρωπαϊκών εκλογών που ήδη έχει αποτύχει Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ και όσον αφορά τι ακραίε δυνάμει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το καταψήφισα. Ευχαριστώ. Μπρουτζίνσκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χτες ε, έγινε μία συζήτηση και πολλοί ανέφεραν τα λόγια του Ρομπέρ Σούμαν του ιδρυτή της Ένωσης που είχε πει ότι είτε θα έχουμε χριστιανική Ευρώπη είτε η Ευρώπη δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, το σημαντικότερο πράγμα για το μέλλον της ε, Ευρώπης και δεν μιλάω για τα θεσμικά όργανα ε, μας λέτε εδώ πέρα ότι είναι η διαδικασία των υποψηφίων ε, ή η προσωπικότητα του κυρίου Φερχόφστατ που θα προεδρεύσει στην διαδικασία. πρέπει να προστατεύσουμε την παραδοσή μας γιατί ναι πρέπει να υπάρχει ένα όραμα για το μέλλον αλλά πρέπει να θυμόμαστε και από πού ε, προερχόμαστε. Μπορούμε να αντιδρούμε μόνο στα καθημερινά, χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο όραμα. Εγώ καταψήφισα αυτό το ψήφισμα γιατί από ό,τι άκουσα δεν ακούστηκε λέξη για την Ευρώπη ως κοινότητα αξιών οι αξίες αυτές, ε, η Αγία Γραφή, η ελληνική, η ελληνική φιλοσοφία και το ρωμαϊκό δίκαιο. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ε, είναι κάτι ε, το οποίο αφορά καλοπληρωμένους ε, εκπροσώπους πολιτικού του συστήματος. Αυτό δεν βοηθήσει. Αν θέλετε να είστε πιο κοντά στους Ευρωπαίους εργαζομένους, ε, καλό θα ήταν να αρχίσουμε από περικοπές μισθών. Η κυρία Φοντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα βγάζει το μήνα, 32 χιλιάρικα. Ο πρόεδρος Σαλ Μισελ του Συμβουλίου, επίσης, ένας βουλευτής εδώ εύκολα βγάζει 10.000 το μήνα. Πώς θα καταλάβετε τι ζουν οι εργαζόμενοι που δεν βγάζουν το μήνα με τους μισθούς που έχετε. Και μια που μιλάμε γι' αυτό, στο μέλλον θα πρέπει ε, να αποτρέψουμε να γίνονται ε, Ευρωπαίοι Υπουργοί, δηλαδή Επίτροποι, κάποιοι άνθρωποι που έρχονται από τις πολυεθνικές. Τότε μπορεί να έχουμε μια αμυδρή ε, αξιοπιστία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα συνεχίζουμε. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν εσά για να τα λέτε ευτυχώς. Ο κύριος Μόντρα από το ΙΣΙΑ. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Αποχαιρετούμε τους Βρετανούς συναδέλφους μας σε δύο εβδομάδες. Για τελευταία φορά ε, θα τους συναντήσουμε στην Ολομέλεια στις Βρυξέλλες και θα πρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και διδάγματα από αυτό με κοινή λογική. Δυστυχώς η συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ είναι ακριβώς το αντίθετο φυγή προς τα εμπρός, όλο και περισσότερη ένωση, όλο και στενότερη ένωση. Ενώ είμαστε διχασμένοι εδώ και διχάζουμε και τα έθνη και τους λαούς. Να μην αφήσουμε να εγκατασταθεί ένα χάσμα μεταξύ ημών και των Ευρωπαίων πολιτών. Χάρηκα τόσο πολύ που ξεφορτωθήκαμε τα κομμουνιστικά καθεστώτα και γίναμε μέλος της Δυτικής Ευρώπης. Αλλά αυτή τη στιγμή ε, είμαι συντετριμένος γιατί βλέπω το κόμμα μου, το ECR, να αποκλείεται από τη συζήτηση γιατί δεν σας αρέσουν οι απόψεις μας. Και οι κομμουνιστές εδώ στο Κοινοβούλιο θα ήθελαν να αγκαλιάσουν τον Πούτιν. Ο κύριος Τζαμπάσκι, παρακαλώ, από την ίδια ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ καταψήφισμα αυτό το ψήφισμα γιατί υποτίθεται ότι αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Δεν, δεν είναι όμως ένα ε, φάρμακο, αλλά είναι ε, ένα δηλητήριο και το δηλητήριο αυτό είναι ε, ο αριστερός φιλελευθερισμός. Περί αυτού πρόκειται. Η Ευρώπη όμως δεν είναι η δικτατορία των, της δεν είναι στη συνέχεια της ε, πολιτισμικότητας ή στη, σε λάθος οικογενειακά πρότυπα. Το μέλλον, όπως το βλέπουμε οι άνθρωποι που αυτοποκαλούμαστε πατριώτες, ανήκει σε, μια σε μια ένα ισχυρό ε, έθνος, μια Ευρώπη που σέβεται το εθνικό κράτος και την εθνική κυριαρχία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαχραντήλ επίσης από το ECR. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θυμάμαι ότι ήμουν ένας εξ αυτών που συμμετείχε στη συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης πριν από κάποια χρόνια. Είμαι της άποψης ότι αυτή η συνέλευση θα ακολουθήσει το παρόμοιο ε, πρότυπο και στο παρελθόν η συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης τότε μίλησε για ένα σύνταγμα το οποίο μετά βαφτίστηκε συνθήκη της Λισαβόνας και βασικά ήταν ε, το, η ιδέα των φεντεραλιστών ε, και το όνειρό τους ήταν περαιτέρω ολοκλήρωση και αυξημένες εξουσίες για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, και λιγότερες εξουσίες για τα εθνικά κράτη. Φοβούμε πως αυτό τη φορά θα έχουμε παρόμοιες εξελίξεις γιατί βλέπουμε τις ε, επικριτικές φωνές που είναι κατά της περαιτέρω ολοκλήρωσης να αποκλείονται από τη συζήτηση, πράγμα που βρίσκω απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ και κλείνουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Επόμενο θέμα είναι η κατάσταση στην Φενεζουέλα. Επεξηγήσεις ψήφου σε σχέση με αυτή την έκθεση. Πρώτος ομιλητής ο κύριος Μαριάννη ε, ID. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Γιώργο και ε, ο Γιώργο. Ε, Χουαϊάν Γουαϊδό και ο Μαντούρο αγνοούν κάθε δική μας ε, παρέμβαση και το Ευρωκοινοβούλιο τα βρίσκει αυτά φυσιολογικά. Αν αύριο βάλει στη φυλακή στους ε, δημοσιογράφους μας αυτό θα, σημειωθεί, θα, θα αφαιρεθεί επίσης σωστό. Ε, είμαστε εγκλωβισμένοι σε, μάλλον είναι εγκλωβισμένοι σε ιδεολογικές υπερβολές και καταδικάζει τον πληθυσμό του στην εξορία. Ε, οι αμερικανικές κυρώσεις ε, κατά του κράτους της Βενεζουέλας δεν αποδεικνύουν ότι πίσω από τις ανθρωπιστικές τάσεις κρύβεται μια πολιτική βούληση για άσκηση πολιτιστική και οικονομική ηγεμονία σε αυτό το κομμάτι του κόσμου. Ανθρωπιστική επίγουσα κατάσταση δεν μπορεί να λυθεί με οικονομικές κυρώσει. Αυτό το θέμα των κυρώσεων, του εμπάργου, τη επέκταση αυτών των κυρώσεων στις οικογένειε, τους ε, και κοντινούς τους και στου γείτονές τους ε, ασκεί τεράστια πολιτική πίεση. Ο κύριος Πόσπισιλ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα που επικρίνει τα, παράνομα βήματα του ε, δικτάτορα ε, Μαντούρου. Το έχουμε συζητήσει επανελειμμένα στην Ολομέλεια. Έχει αυξήσει την εξουσία του, παρανόμως αντικαθιστώντας τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Οφείλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις κατά του καθεστώτος του Μαντούρο και να αποφασίσουμε ε, εάν και κατά πόσο θα προβούμε σε σκληρότερες ενέργειες. Από την άλλη πλευρά, η ανθρωπιστική βοήθεια φυσικά και θα πρέπει να προσφερθεί. Είναι φρικτή κατάσταση. Ε, ανθρωπιστική καταστροφή εκτελήσεται στην Βενεζουέλα. Δεν είναι λάθος των, ε, των πολιτών που κυβερνώνται από αυτόν τον δικτάτορα. Κυρία Πρόεδρε, εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα. Εδώ και 20 χρόνια υποφέρει από την σοσιαλιστική δικτατορία η Βενεζουέλα. Και όπως σε κάθε χώρα, ο σοσιαλισμός έφερε φτώχεια και πείνα. Λοιπόν, η Βενεζουέλα είναι μια πλούσια χώρα. Έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Και παρόλα αυτά 70% ε, των παιδιών ε, υποσυτίζονται. Οι Βενεζολάνοι φεύγουν. Ε, πρέπει να τελειώσει κάποτε αυτό. Χρειάζεται επιτέλους ελευθερία και δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Wallace, από την η αναγνώριση του Γκουαϊντό είναι πλέον ακόμη πιο γελία γιατί 150 από τα 165 μέλη της Εθνοσυνέλευσης εξέλεξαν τον Λούις Πάρα ως νέο πρόεδρο. Ο Πάρα είναι από το κόμμα Πριμέρου Ζουστήσια, δεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης. Δεν εμποδίστηκε ο Γκουαϊντό να μπει στην Εθνοσυνέλευση όπως λέει ο κύριος Μπορέλ βλέπετε, είπε στις κάμερες ότι αρνήθηκε να μπει χωρίς τη συνοδεία 11 πρώην βουλευτών. Μετά οργάνωσε αυτή την διαδήλωση που ανέβηκε εκεί πέρα στο κάγκελο κλπ. Λοιπόν, είναι απογοητευτική κατάσταση και θλιβερή κατάσταση. Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζει αντιδημοκρατικά καθεστώτα για μία ακόμη φορά και αλλαγή. Είναι τρελό. Γιατί να αφήνουμε τους Βενεζουελάνους να αποφασίσουν μόνοι τους και να τους επιβάλλουμε μιζέρια και να αρθούν οι κυρώσεις και να αποφασίσουν οι Βενεζουελάνοι τη μοίρα τους. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Τόματς από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα και με τεκπλήξεως ακούω εδώ στην Ολομέλεια εκείνους εδώ που έχουν διαφορετική άποψη για τον Μαδούρο. Δεν τον θεωρούν δικτάτορα. Είναι δικτάτορας και οποιοδήποτε δικτάτορας που έχουμε δει σε όλη την ιστορία είδαμε ότι αψηφά το λαό πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης προς εκατομμύρια πολίτες στη Βενεζουέλα που υποφέρουν σε αυτή τη φάση. Πρέπει να δράσουμε πολύ πιο με μεγαλύτερη πίεση στις, ε, επ' αυτού του καθεστώτος όσον αφορά τα μέτρα που του επιβάλλουμε, να είναι πιο στεναρά. Είναι απίστευτη η κατάσταση επικρατική για εκατομμύρια πολίτε. Εγώ είμαι με του Βενεζουελάνου και θα πρέπει να παλέψουμε την ελευθερία αυτού του λαού. Ευχαριστώ κύριο Σαχραντήλ, εκ μέρου του ΙΣΙΑΡ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συζητούμε για άλλη μια φορά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, διότι σε ό,τι αφορά τη Λατινική Αμερική, η αριστερά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που βεβαίως δεσπόζει, ε, μιλάει για τη Βραζιλία, την Κολομβία, τα καθεστώτα εκεί, τα καθεστώτα δηλαδή που θεωρεί δεξιά, αλλά σιωπά όταν μιλούμε για καθεστώτα τα οποία είναι αριστερές δικτατορίες όπως η Κούβα ή η Βενεζουέλα. Καλό είναι λοιπόν να τα συζητάμε αυτά και νομίζω ότι όταν έχουμε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν έχουμε τραγικές οικονομικές καταστάσεις ε, όπου οδηγεί ένα σοσιαλιστικό καθεστώ, ε, νομίζω πω είναι σημαντικό να τα συζητάμε αυτά στο πλαίσιο εξωτερική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε στην επόμενη συζήτηση. Δηλαδή το άρθρο 7, τη δικασία άρθρο 7 κατά της ε, Πολωνίας και της Ουγγαρίας. Ο κύριος Φόξ, ένα ο πρώτος ομιλητής. Εγώ ψήφισα κατά, διότι το άρθρο 7 χρησιμοποιείται ως ε, ένα μέσο εκφοβισμού προς τους Πολωνούς ε, εκλογής. Οι Ούγγροι και οι Πολωνοί εκλογής είναι αυτοί που αποφασίζουν. Υπάρχει μια ένταση στο Κοινοβούλιο, υπάρχει μια πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς ένα ομοσπονδιακό σύστημα όπου όλες, όλοι οι εθνικοί πολιτισμοί, όλες οι διαφορές πρέπει να εκκριζωθούν, να, ε, κατα, να καταπατηθούν. Μιλάτε για ποικιλομορφία, αλλά στην πραγματικότητα δεν αποδέχεστε ε, τις διαφορετικές απόψεις. Ε, περιφρονείτε την εθνική κυριαρχία και απαγορεύεται ε, ολόκληρα εθνικά κινήματα εδώ στην Ουγγαρία και την Πολωνία την διώκεται επειδή διώκεται επειδή υποτίθεται ότι δεν σέβονται τι ευρωπαϊκέ αξίε. Οι ευρωπαϊκέ αξίε όμω ε, μιλάνε και για αυτοδιάθεση, για ε, λαϊκή κυριαρχία, για δημοκρατία και κυρίω ανοχή απέναντι στι πολιτικέ απόψει με τι οποίε ε, διαφων, διαφωνεί κανεί. Εγώ δεν συμφωνώ με την Πολωνία και την Ουγγαρία απαραίτητα και του κυβερνήσει του, αλλά πρέπει ελεύθερα να εκλέγουν τι κυβερνήσει του. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσαρνιέτσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στο επόμενο επεισόδιο της φάρσας ε, του τσίρκου που διαδραματίζεται εδώ και που αφορά τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Πολωνίας που την εξέλεξαν ε, οι πολίτες της χώρας. Ε, ακούμε πολλά να λέγονται η αριστερά ε, μιλά για τη σημασία που έχουν οι πολίτες και ότι πρέπει να ακουστεί η φωνή τους. Όταν όμως κάποιες κυβερνήσεις στρέφονται κατά του κατεστημένου των Βρυξελών, έχουμε αυτό το θέαμα εδώ πέρα, αυτό το τσίρκο. Εγώ καταψήφισα το ψήφισμα γιατί βρήθη ψευδών και μάλιστα περιλαμβάνει διατάξεις που αντιβαίνουν και στις συνθήκες. Τα κρατημέλη είναι αυτόνομα και έχουν ε, το δικαίωμα να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό σύστημα μέσω του Εθνικού Κοινοβουλίου τους. Είναι κράτος δικαίου, ασφαλές κράτος η Πολωνία σήμερα. Δεν μπορούμε ε, να συζητήσουμε και την ε, περίπτωση της Γαλλίας και το κράτος δικαίου που επίσης ε, με βίαιο τρόπο αντιδρά στους σκηγόρους ή στους διαδηλωτές οι αστυνομικοί εξασφαλίζουν την ασφάλεια των διαδηλωτών στην Πολωνία όσων θέλουν να διαδραματήσουν κατά τις μεταρρύθμιση του δικαστικού Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριο Μπροτζίνσκι και τώρα το λόγο ο κύριο Ζαμπάτσκι. Υπερψήφισα, μάλλον ψήφισα κατά του ψηφίσματος αυτού κατά της Ουγγαρίας και της Πολωνίας διότι είναι πονίδιστα τα κείμενα, είναι μια φάρσα αποτελεί κυνήγι μαγισσών αυτών ούτε η Πολωνία ούτε η Ουγγαρία παραβιάζουν πουδενή το κράτος δικαίου την ελευθερία της έκφρασης εντός των χωρών. Το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται έναντι αυτών των χωρών είναι ότι και οι δύο χώρες επέλεξαν κυρίαρχες τα, τις κυβερνήσεις τους, κυβερνήσεις πατριωτών που ξέρουν οι πατριώτες πώς να κυβερνούν τις χώρες τους, που δεν επιτρέπουν αντιχριστιανική προπαγάνδα στις χώρες τους, δεν μπορούσαν να επιτρέψουν τα διατάγματα του ψευδούς πολυπολιτισμικού ε, πλαισίου που επιβάλλονται από ΜΚΟ που πληρώνται από το Σόρος. Είναι κυρίαρχες χώρες η Πολωνία και η Ουγγαρία με κυρίαρχε ανεξάρτητε κυβερνήσει που ε, χρήζουν σεβασμού και δεν θα πρέπει να ακούμε αυτά που λένε οι αριστεροί Μπολσεβίκοι και προσπαθούν να μα επιβάλλουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεμπρετών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα κατά αυτού του ψηφίσματος για την Πολωνία και την Ουγγαρία για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα είναι απαράδεκτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χαίρεται που έχει ενεργοποιηθεί το άρθρο 7 ε, της ε, συνθήκης της Ένωσης κατά των χωρών αυτών. Λέμε εδώ ότι υπάρχει παραβίαση της ε, ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Η εθνική κυριαρχία της κάθε χώρας της δίνει το δικαίωμα να οργανώσει τη δικαιοσύνη όπως το θέλει. Η Ουγγαρία μπορεί να προστατευτεί σαφώς από τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης του Τζορτ Σόρο. Δεύτερον, ε, είναι απαράδεκτο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προτείνει ε, μια διαδικασία παρακολούθησης ε, από υποτίθεται ανεξάρτητους ε, ε, σοφούς. Δεν μπορεί να υπάρχει ιδεολογική ε, εποπτεία ούτε στην Ουγγαρία, ούτε στην Πολωνία, ούτε στην Γαλλία, ούτε σε καμία άλλη χώρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ζόγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε παίρνω το λόγο διότι χθες ε, στη συζήτηση ακούσαμε πραγματικά πολλά ψέματα. Ένας ε, Έλληνας βουλευτής, ε, κομμουνιστής φαντάζομαι, είπε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. όταν η Ελλάδα όμως στην οικονομική κρίση ε, έκανε όλες αυτές τις απάτες, πού ήταν ε, αυτός ο άνθρωπος. Δεν θέλουμε άλλα ψέματα. Στην Πολωνία ε, υπάρχει και κράτος δικαίου, υπάρχει και δικαιοσύνη. Ε, χρησιμοποιούμε πολύ καλά τα χρήματα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Αυτό το αποδεικνύουν τα στοιχεία του Eurostat. Οι άνθρωποι είναι όλο και πιο ευτυχισμένοι στη χώρα μας. Το κόμμα που έχασε βέβαια τις εκλογές ε, θέλει τη ρεβάνς κατά κάποιο τρόπο. Οπότε ξαφνικά οι δικαστέ πολιτικοποιούνται. Αυτό είναι μια πολύ κακή συνήθεια. Για όλου του λόγου ψήφισα κατά. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Προχωρούμε στο επόμενο σήμερα τη μέσα διάταξη. με επεξηγήσει ψήφου σε ό,τι αφορά τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα. Κύριο Ρόβετ. Η κυρία. Uh, Ευχαριστώ. Είμαστε στο χείλο μιας ανεπανόρθωτης καταστροφής για τη βιοπικιλότητα και πράγματι σήμερα εγκρίναμε ένα ψήφισμα στο Κοινοβούλιο για την 15η διάσκεψη των μερών για τη βιολογική ποικιλότητα. Είναι μια στιγμή που αύξησε σημαντικά τις πράσινες ψήφους στο Κοινοβούλιο και υπάρχει και μετακίνηση της κοινή γνώμης, αλλά είναι απογοητευτικό να βλέπουμε πληθώρα ε, ψηφοφόρων από την άλλη πλευρά, ε, στην άλλη πτέρυγα, που προσπαθούν να βάλουν φρένο και στρέφονται κατά των προτάσεων αυτών. Προδώνουν τα ζώα, προδίδουν τα ζώα, προτείνουν τον άνθρωπο, αυτό το συλλογικό project που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μας αποτρέπουν, γιατί μας εμποδίζουν από τη μαριτερισμή της κοινής γεωργικής πολιτικής, γιατί μας κρατάνε πίσω από αυτά που πρέπει να γίνουν τώρα που ο πλανήτης κινδυνεύει. Πρόεδρος. Και περνάμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης που είναι τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Ένωσης πρόκειται των συγκρούσεων συμφερόντων υποστήριξε αυτό το ψήφισμα αναφυσβήτητα. Θέλει ο λαός να δει διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά. Από όταν υλοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Νομισματική Ένωση, οι σκεπτικιστέ, οι λαϊκιστές και οι προασπιστέ του Brexit έλεγαν ότι είναι μια καταστροφή και ότι η ευρώ σίγουρα θα κατέρε. Λάθο έκαναν. Έσφαλαν. Βαθισών των περιστάσεων το ευρώ τα πήγε πολύ καλά, αξιοσημείωτα καλά και εγώ διατείνομαι ότι θα εξακολουθεί να υπάρχει πολύ αφού τελικά έχουν λησμονηθεί ανοήσίε τους. Ο χρόνος είναι τα πάντα. Εγώ φαίνεται να είμαι ο τελευταίο βουλευτή του Ηνωμένου Βασίλειου που μιλά σε αυτήν την αίθουσα. σω να μην ξαναμιλήσω ξανά στη Σύνοδο των Βρυξελών, αλλά πρέπει να ευχαριστήσω κάποιου. Εσά και του αντιπροέδρου και του φίλου, συναδέλφου θέλω να ευχαριστήσω και αντιπάλου, αλλά ποτέ εχθρού σε αυτή την αίθουσα. Πάνω απ' όλα είναι κανεί όσο καλός, καλό είναι το προσωπικό του. Δημοσία ευχαριστώ την Κέι Βέλξορ, Σάρα Μακίνλε και, την Κιμ Τσάπμαν στο γραφείο μου του Ηνωμένου Βασιλείου και την ομάδα των Βρυξελών που ήταν πολύ πιστή μέχρι τελευταία στιγμή και ε, ευχαριστώ πολύ ξανά κάνει όταν επαξενελέγει τον Μάιο ευχαρίστησα την αστυνομία και το εκλογικό προσωπικό και λησμόνησε έναν άνθρωπο που, άνευ του οποίου δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Η Τζέιν Kearney, Τζέιν, δεν μπορώ να τα πω πιο δημόσια από τότε. Η χειρότερη πτυχή από όλε τι θέσει μου θα είμαι μακριά από σένα. Ευχαριστώ πολύ. Σε αγαπώ. Όλοι μου ζητούν να πω τι θέλω σαν επόμενο. Εγώ θέλω εσένα. Ezzel a napi rendi pontunknak a végére értünk. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι επεξηγήσεις ψήφου και η συνεδρίαση θα επανθήσει στις 3.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 16 Ιανουαρίου η διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε την πρόταση ε, ημερολογίου για τις συνόδους του 2020 και 2021 και 2022. Οι ημερομηνίες έχουν ως εξής. Για το 2021, 18 με 21 Ιανουαρίου, 8 με 11 Φεβρουαρίου, 8 με 11 Μαρτίου, 24 και 25 Μαρτίου, 7 και 8 Απριλίου, 26 με 29 Απριλίου, 7 με 20 Μαΐου, 7 με 10 Ιουνίου, 23 και 24 Ιουνίου, από 5 μέχρι 8 Ιουλίου, 13 με 16 Σεπτεμβρίου, 4 με 7 Οκτωβρίου, 18 με 21 Οκτωβρίου, 10 και 11 Νοεμβρίου, 22 με 25 Νοεμβρίου, 13 με 16 Δεκεμβρίου. Για το 2022, 17 με 20 Ιανουαρίου, 14 με 17 Φεβρουαρίου, 7 με 10 Μαρτίου, 23 και 24 Μαρτίου, 4 με 7 Απριλίου, 2 με 5 Μαΐου, 18 και 19 Μαΐου, 6 με 9 Ιουνίου, 22 και 23 Ιουνίου, 4 με 7 Ιουλίου, 12 με 15 Σεπτεμβρίου, 3 με 6 Οκτωβρίου, 17 με 20 Οκτωβρίου, 9 και 10 Νοεμβρίου, 21 με 24 Νοεμβρίου, 12 με 15 Δεκεμβρίου. Η διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να αποφασίσει να προσθέσει ε, συνόδους ε, ελέγχου κοινοβουλευτικού Τετάρτη απόγευμα ε, των εβδομάδων πολιτικών ομάδων και επιτροπών στις Βρυξέλλες. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 28 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα. Η ψηφοφορία θα γίνει την 5η στις 30 Ιανουαρίου στις 11.30. Οι ημερομηνίες διατίθενται και στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Επόμενο θέμα στη μέσα διάταξη, παράνομα αντικείμενα τρισδιάστατη εκτύπωση. προφορική ερώτηση. Μπορείτε να ζητήσετε το λόγο στο ΚΑΣΤΙΑΙ με μπλε κάρτα, με την παραδοσιακή μέθοδο ή με τη νέα ηλεκτρονική. Θα βρείτε σχετικές οδηγίες στην είσοδο του ημικυκλίου. Θα ε, δώσω τώρα το λόγο στη συντάκτρια για πέντε λεπτά, ε, η κυρία Σχράινμαχερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια τεχνολογία με σημαντικές ε, δυνατότητες για μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις. Και πολλές χώρες έχουν αρχίσει να αυτούν στρατηγικές προώθησης αυτής της ε, τεχνολογίας. Υπάρχουν όμως ε, νομικά και διαντολογικά ζητήματα. Διάφορες μελέτες κομισιών έχουν δείξει την ύπαρξη κάποιων παραθύρων είχαμε κάποια πρόσφατα τραγικά γεγονότα που εγείρουν ανησυχίες ε, και την ανάγκη άμεσης δράσης. Σε 9 Οκτωβρίου 2019, δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλα δύο τραυματίστηκαν στο Χάλε, στη Γερμανία, όταν προσπάθησε ένας επιτιθέμενος να μπει στην συναγωγή κατά τη διάρκεια της αργίας του Γιώμ Κιπούρ. Χρησιμοποίησε ένα όπλο τυπωμένο σε τρισδιάστατο εκτυπωτή και είχε ανεβάσει τα σχέδια στο Twitter – Ήδη το 2018 η Επιτροπή Γιουρή είχε εκφράσει τις ανησυχίες της ε, για την κατασκευή όπλων εκρηκτικών και ναρκωτικών. Αλλά και σε σχέση με ζητήματα αστικής ευθύνης ε, και ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα θέλαμε λοιπόν να ρωτήσουμε την Κομισιόν το εξής. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα. Προβλέπετε κάποια νομοθετική δράση με βάση υφιστάμενες ή προηγούμενες μελέτες. Εάν ναι, ποια μέτρα προβλέπετε να επηρεαστούν και με τι χρονοδιάγραμμα. Τι θα κάνετε για να διασφαλίσετε μια έγκαιρη αντίδραση. Και τέλος, τι έχει ε, δεσμευτεί να κάνει η Κομισιόν μετά την έκθεση της Επιτροπής Γιούρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Επίτροπο. Να έχετε τον λόγο, κύριε Ελένα Τσίτση. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, συμφωνώ με την άποψη του Κοινοβουλίου, όπως αυτή εκφράστηκε στην έκθεση του 2018, την οποία αναφέρετε κι εσείς ότι δηλαδή η τεχνολογία αυτή μπορεί να γύρει ζητήματα ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας ειδικά όσον αφορά την κατασκευή όπλων εκρηκτικών, ναρκωτικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα ζητήματα. Το πρόβλημα με τα πυροβόλα όπλα που έχουν τυπωθεί δεν είναι ότι θα είναι ελαττωματικά και θα υπάρχει ζήτημα ευθύνη. Είναι ότι έχουν κατασκευαστεί και χρησιμοποιούνται παράνομα. Σύμφωνα με την οδηγία περί όπλο κατοχής, ε, πυροβόλων όπλων, η, παρα... η κατασκευή των όπλων είναι ήδη παράνομη, ε, εκτός αν έχει δοθεί άδεια από την αρμόδια αρχή ε, κράτους μέλους ε, όπου λαμβάνει η χώρα η κατασκευή συναρμολόγηση. Και αυτό ισχύει και για την τρισδιάστατη εκτύπωση και για την χρήση προδιαγραφών που υπάρχουν ε, διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση και λαμβάνουμε υπόψη και τον κύκλο χάραξης πολιτικής της Ένωσης. Το επιχειρησιακό σχέδιο 2020 περιλαμβάνει μια δράση που στόχο έχει να ενημερώσει για τον κίνδυνο από τις νέες τεχνολογίες. Η Europol πέρσι τον Οκτώβριο απέστειλε ένα σήμα σε όλες τις ε, διοκτικές αρχές για το θέμα αυτό. Η Κομισιόν προετοιμάζει μια έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας που καλύπτει ζητήματα συγκεκριμένα των αντίκτυπων νέων τεχνολογιών όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση. Η έκθεση αυτή θα αξιολογήσει το εάν απαιτείται περαιτέρω δράση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες για δύο λεπτά. Ο κύριος Γκαρσία Δελμπλάνκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη, ξεχάστηκα γιατί είμαι εδώ με την οικογένειά μου. Μάλιστα, είμαστε στην οικογενειακή ατμόσφαιρα. Θα μιλήσω ισπανικά. Όσοι ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, θα συμφωνήσουμε ότι Πρόκειται για ένα τεχνολογικό εργαλείο, μια τεχνολογική πρόοδο εκδημοκρατισμού και από τη μια είναι τεράστια ευκαιρία. Η τρισδιάστατη εκτύπωση ε, φυσικά έχει πολλές πτυχές και εκφάνσεις, αλλά είναι προφανές ότι μπορεί να μας βοηθήσει ακόμα και από τη σκοπιά ε, της εξοικονόμησης υλικών. Λιγότερη ρήπανση, δηλαδή η παραγωγή μπορεί να γίνεται αποκεντρωμένα όλο και περισσότερο, με περισσότερα και μεγαλύτερα μηχανήματα στον τόπο όπου χρειάζεται ε, ε, να ασκηθεί η δραστηριότητα και έτσι αποφεύγουμε περιττές μεταφορές. Εκδημοκρατισμός γιατί ο κόσμος έχει πρόσβαση σε κάποια πράγματα. Από την άλλη όμως υπάρχει ε, και σημαντική πρόκληση για διάφορα πράγματα. Μεταξύ αυτών είναι και ασφάλεια. ακούσαμε ότι έχει να κάνει με τη δυνατότητα δυνατότητα, χωρίς να πάμε μακριά, να ε, τυπώσουμε όπλα. Τους τελευταίους μήνες και χρόνια είδαμε πόσο δύσκολο είναι ακόμα να ελεγχθούν διάφορα όπλα και μπορείς από το βαθύ ίντερνετ να τυπώσεις και να κατεβάσεις οδηγίες να τυπώσεις ένα όπλο. Έλεγα λοιπόν ότι είναι προκλήσεις που δεν έχουν ακόμα ρυθμιστεί καλά νομικά και επ' ευκαιρία θέλω να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το λάβει υπόψη της. Να το κοιτάξει και από τη σκοπιά της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ε, ε, ο έλεγχος έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολύ αποτελεσματικός για την πνευματική παραγωγή προσώπων ή ομάδων που τα παράγουν αυτά. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις πολύ αθολές, συγκεχημένες και ευρείες. Τώρα είναι πώς ρυθμίζεις το ίδιο το, διαδίκτυο, το παγκόσμιο ιστό και την ε, πρόσβαση σε πνευματική ιδιοκτησία και πολιτισμικά αγαθά. Τελειώνω και ζητώ συγγνώμη που μακρηγορώ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ να καλύψει κάποια νομικά κενά που υπάρχουν για να μπορέσουμε καλύτερα να ελέγξουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της ομάδας Renew Europe και πάλι κυρία Σχράινμαχερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Επίτροπο για την απάντησή του. Θα ήθελα να συνεχίσω στη γλώσσα μου που είναι τα Ολλανδικά. Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια τεχνολογία η οποία καλπάζει και έχει πολύ μεγάλο δυναμικό για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και μεγάλες και μικρομεσαίες. Οι δυνατότητες ε, δεν έχουν τέλος. Έχει βελτιώσει πάρα πολύ τη ζωή μας. Σκεφτείτε ότι ε, στην ιατρική τυπώνουν ε, τεχνητά μέλη ή ακόμα και στις οικοδομές μπορεί να χτίσουν μέσα σε 48 ώρες σπίτια ολόκληρα τυπωμένα. Ε, αλλά άμα πέσει σε λάθος χέρια, όπως κάθε τεχνολογία, είναι επικίνδυνη. Ε, Είδαμε στο Χάλε που προσπάθησε κάποιος ε, να μπει σε μια συναγωγή και σκότωσε δύο και άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Είναι πολλά τα καλά από τη τρισδιάστατη ε, εκτύπωση, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και επικίνδυνες εφαρμογές, τυπώνουν ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικά. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε εάν τα ρυθμίζουμε πάρα πολύ καλά. Και υπάρχει το επιχειρησιακό σχέδιο δράση βεβαίω ε, και οι διοκτικές αρχές, οι ασχολούνται, αλλά το ερώτημα είναι αρκούν όλα αυτά. γιατί εκεί υπάρχει θέμα ευθύνη ευθύνης πνευματικής ιδιοκτησίας και οδηγία για τα πυροβόλα όπλα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με το θέμα όταν κάπως τυπώνονται παράνομα ε, τα όπλα. Και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνετε. Είπατε τι προτίθεστε να κάνετε και τι έχετε ήδη κάνει. Χρειάζεται νέα νομοθεσία, θα έρθουν νέα πρότυπα. Γιατί συμφωνούμε όλοι εδώ ότι δεν πρέπει να ξαναζήσουμε τέτοια φαινόμενα όπως στη Γερμανία. Σε ευχαριστώ πολύ. Για τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς, ο κύριος Τζαμπάσκη για τρία λεπτά. Λοιπόν, ας μετρήσουμε. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις άνθρωποι στην αίθουσα. Πριν μπω στο θέμα μας, απευθύνομαι σε εσά, κυρία Πρόεδρε να πω κάτι που είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση και στην προπροηγούμενη και θα το ξαναπώ και σήμερα. Με τόση λίγη στην αίθουσα πέμπτη απόγευμα είναι ντροπή. Πρέπει να αλλάξουμε πρακτική. Είτε πρέπει να καταργήσουμε αυτές τις συνεδριάσεις ή ο κόσμος να παίρνει τη μισή ημερήσια αποζημίωση. Να το ξαναπώ, είναι έσχος. Σας παρακαλώ λοιπόν να μεταφέρετε το μήνυμα αυτό σε αρμόδιες αρχές. Στο θέμα μας τώρα. Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι πάρα πολύ σημαντική τεχνολογία. Θα οδηγήσει παραδείγματος χάρη σε καινοτομίες ε, στην ιατρική. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει πράγματα τέτοια. αλλά υπάρχουν εδώ πέρα κάποιοι κίνδυνοι και πρέπει να λάβουμε μέτρα. Δεν είναι δυνατόν ανήθιοι άνθρωποι να έχουν όπλα στα χέρια τους ανοίγοντας μόνο έναν φιλομετρητή στο διαδίκτυο. Δηλαδή αυτά τα όπλα μπορούν να φτάσουν στα χέρια τρομοκρατών. Το γεγονός και μόνο ότι ανοίγεις ένα browser και μαθαίνεις πόσο θα φτιάξεις όπλο μας δείχνει ότι υπάρχουν παραθυράκια που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Στη χώρα μου δε, την Βουλγαρία, υπάρχει ένα πρόβλημα με την εγκληματικότητα σε μικρές πόλεις ε, και χώρια. Ε, καμιά φορά χρειάζεται όπλο για να προστατεύσει κανείς την οικογένειά του. Άλλες φορές, ε, καμιά φορά μπορεί να σταματήσει κάποιον όπλο μόνο αν έχει όπλο. Λοιπόν, Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να εμποδίζει κάποιον που θέλει να αποκτήσει όπλο νομίμως. Μιλήσαμε στο παρελθόν για απαγορεύση των κυνηγετικών όπλων. Αυτό θα οδηγήσει μόνο στην καταστροφή ε, παλαιών ε, συνηθιών. Χρειάζονται λοιπόν άλλα μέτρα για να προστατεύσουμε τις ε, παραδοσιακές δραστηριότητες. Και μην ξεχνάτε ότι ελεύθερο είναι κανείς μόνο όταν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. And uh, my last speaker... Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Λομπάκοφ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω μια δήλωση, αλλά έχω και μια-δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Τζαμπάσκι, αν μου επιτρέπετε. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε ένα τυπωμένο ε, όπλο και ένα πραγματικό. Δεν υπάρχει πραγματική διαφορά. Κύριε Τζαμπάσκη, αυτή είναι η ερώτησή μου. Εσείς πιστεύετε πως υπάρχει ερώτηση. η ερωτηση μου εσει πιστευετε πω υπαρχει ερωτηση εγω αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχω ένα σπίτι, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω στο σπίτι μου. Κανείς δεν μπορεί να μπει αν εγώ δεν το επιθυμώ και μπορεί εγώ να θέλω να τυπώσω και να καλάσνικοφ. Μπορεί να μου αρέσουν αυτού του είδους τα όπλα. Και δεν καταλαβαίνω Πώ γίνεται ο άνθρωπο να μην μπορεί να, ένας άνθρωπος να μην μπορεί να, να προστατέψει τη ζωή του. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Εάν κάποιο μου επιτεθεί με μια αξίνα, θα πρέπει και εγώ να, το, να μπορώ να α, απαντήσω με το ίδιο όπλο. Μπορεί να έχω μια ολόκληρη βαλίτσα δίπλα μου. Κοιτάξτε, εγώ κατάλαβα από την κάρτα σα ότι πρόκειται για κάτι αλλά καταλαβαίνω καλύτερα τώρα πώ πρόκειται περισσότερο για μπλε κάρτα προ τον κύριο Τζαμπάσκι. Ναι, μάλιστα. Κύριε Τζαμπάσκη, δέχεστε την ερώτηση που σας ετέθη. Μάλιστα, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. για να μην ε, τυπώνουν όπλα οι πολίτες, νομίζω πως οποιοδήποτε νομοταγής πολίτης που δεν έχει καταδικαστεί θα πρέπει να έχει την επιλογή να προστατεύει τον εαυτό του χωρίς να παραβιάζει οποιαδήποτε νομοθεσία. Μάλιστα. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο και πάλι στον Επίτροπο Λέναρτιτ. Σας ευχαριστώ για αυτή τη σύντομη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ε, τα αναφέρω όλα αυτά στους συναδέλφους και σας διαβεβαιώ πως θα δούμε το θέμα από όλε τις πτυχές που αναφέρατε σήμερα, αλλά να σας δώσω κάποιο αρχικό feedback. Να αρχίσω με το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Κομισιόν πρόσφατα ανέθεσε ε, μελέτη περί δικαιωμάτων ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και των επιπτώσεων αυτών στην βιομηχανική τρισδιάστατη εκτύπωση. Το στόχος είναι να μελετήσουμε και να αναλύσουμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του είδους η εκτύπωση σε βιομηχανικό επίπεδο. Θα μελετήσουμε λοιπόν τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της μελέτης και μετά θα αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα. Φυσικά ο αγώνας κατά των νοθευμένων ή παραχαραγμένων προϊόντων, είτε είναι τρισδιάστατα είτε όχι, τρισδιάστατη εκτύπωση είτε όχι, συνεχίζεται. Τώρα, ε, ευθύνη για ε, του παραγωγού του προϊόντος ε, σας δημοσιεύσαμε την πέμπτη μας έκθεση σε σχέση με την οδηγία για την ευθύνη και την αξιολόγηση αυτής το 2018. Επίσης δημοσιεύσαμε ένα έγγραφο εργασίας για την ευθύνη για τις αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες τον ίδια χρονιά. Επιπλέον η Κομισιόν εργάζεται για ένα έγγραφο ε, καθοδήγησης σε σχέση με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας ε, ένα εγχειρίδιο εφαρμογής το οποίο θα εκδοθεί αργότερα φέτος. Επίσης θα δούμε κατά πόσο είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αυτή η οδηγία για την ευθύνη για το, του προϊόντος. Και τέλος για την παράνομη παραγωγή όπλων. Το περιστατικό που αναφέρατε στο Χάλε φυσικά εξετάστηκε πάρα πολύ ε, εξονυχιστικά από τις γερμανικές αρχές και μεταξύ άλλων το γερμανικό Bundestag ε, κατέληξε ότι δεν χρειάζεται νέα νομοθεσία διότι ο ισχύων γερμανικός νόμος ρητά ε, καταδικάζει την παράνομη κατασκευή όπλων άσχετα από τον τρόπο παραγωγής τους, τη μέθοδο παραγωγής τους. Ωστόσο, η Κομισιόν θα υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας περί πυροβόλων όπλων καθώς και έναν έλεγχο καταλληλότητα των διατάξεων που θα συνοδεύεται αν χρειάζεται από νομοθετικές προτάσεις που θα αφορούν τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση αλλά και η χρήση των κωδικών QR και των ραδιοσυχνοτήτων. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ολόκληρον τη συζήτηση. Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνόδου. Αν δεν διαφωνείτε θα διαβιβάσω αρμοδίως τα ψηφίσματα που εγκρίναμε σήμερα. Σε αρμόδια πρόσωπα και όργανα. Διακόπτεται η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λέει τη συνεδρίαση. Καλό σας απόγευμα.